Ladies and gentlemen, so let us start. Λοιπόν, ε, να σας καλωσορίσω και ξεκινάμε. Σας καλωσορίζω στην Ολομέλειά μας. Την τρίτη για το τρέχον έτος. Να κρίνουμε την ημερήσα διάταξη. Έλαβα ένα τελευταίο αίτημα για το σημείο 18 της σημερινής διάταξης να τεπτά 5-4 δεν μπορεί να παρευρεθεί ο εισηγητής προς το τέλος οπότε θα αναβληθεί ως τελευταία γνωμοδότηση για αύριο το πρωί εάν συμφωνείτε όλοι με αυτή την αλλαγή στην της διάταξη υπάρχει κανείς που να είναι κατά εγκρίνεται λοιπόν η ημέρηση διάταξη Ευχαριστώ πολύ. Να εγκρίνουμε τα πρακτικά της Ολομέλειας στις 20 και 21 Φεβρουαρίου στο κτίριο Σαουλεμάνια. <clears throat> Λάβατε εγκαίρως <clears throat> τα πρακτικά. <clears throat> Έχετε σχόλια. Όχι και ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνονται. Λοιπόν, έγκριση της γνωμοδότησης των γνωμοδοτήσεων χωρίς συζήτηση. Κατευθείαν ψηφίζουμε. Οπότε ψηφίζουμε την γνωμοδότηση ΙΝΤ κάθετος 878 Ευρωπαϊκή Τυποποίηση για το 2019. Η συγγήτρια Ελσβιέτα Ζατζίνσκα. η ψηφοφορία. The vote is closed. 122 υπέρ και μία αποχή εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το INT 879. Εναρμονισμένα πρότυπα. Ο εισηγητής Τζεράρντο Λάργκη. Άρχεται η ψηφοφορία. 125 υπέρ 2 αποχές. Εγκρίνεται. Γνωμοδότηση ε, κατηγορίας Γ. ΣΟΚ 617. Πόροι για το δικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Τροποποίηση. Άρχεται. Πέρας. 132 υπέρ και μία αποχή. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Now we'll go. Και τώρα θα έχουμε τη δήλωση του Πρόεδρου. και θα παρουσιάσουμε παράλληλα την πρώτη επί της ουσίας συζήτηση της Ολομέλειάς μας. Αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω στην Ολομέλειά μας και υπενθυμίζω ότι ο ιστορικός κανόνας, ο κανονισμός και ο κώδικας διοντολογίας που εγκρίναμε τον ε, περασμένο Φεβρουάριο άρχισαν να ισχύουν στις 15 Μαρτίου. Λάβατε όλοι μέσω email τα κείμενα αυτά. Ο κώδικας ε, δεοντολογίας λέει ότι τα μέλη θα πρέπει να υπογράφουν αυτό το κώδικα δεοντολογίας στην αρχή της θητείας τους. Σας ενημερώνω ότι χθες το πρωί επισήμως υπέγραψα μαζί με τους δύο αντιπροέδρους την Μιλένα Αγγέλοβα και την Ζαμέλ Κάνιο αυτό το κώδικα δεοντολογίας. <clears throat> Ήθελα να δείξω ότι δεν περιμένουμε την ανανέωση. Οποιοδήποτε μπορεί να υπογράψει αυτόν τον κώδικα δεντολογίας για να δείξουμε ότι δεσμευόμεθα ως προς τις αρχές που περιέχει. Ο Γενικός Γραμματέας σύντομα θα σας αποστείλει μια ειδική σελίδα στο ίντρανετ ούτως ώστε όσοι το επιθυμούν και ελπίζω να είναι οι περισσότεροι ήδη να προσυπογράψουν. Σας ευχαριστώ να το κάνουμε όλοι για να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ε, εναντίον αυτών που συνεχίζουν να μας, ε, συνεχίζουν να μας επικρίνουν δημοσίως. Παρά τις θετικές δράσεις που έχουμε λάβει για τα θέματα αυτά ήδη, για την ενημέρωσή σας. Πρόσφατα έστειλα μια πολύ κατηγορηματική απάντηση στην επιστολή που εστάλει προς όλους σας από τον κύριο Σεμπαστιάνη, τον πρόεδρο της, του κλάδου της του Συνδικάτου ε, Ανανέωση και Δημοκρατία, του κλάδου τη Κομισιόν λοιπόν αυτού του Συνδικάτου, όπου σα καλεί να μην υπογράψετε αυτό το κώδικα δοντολογία. Επίση, υπενθυμίζω ότι τα έγγραφα αυτά εγκρίθηκαν με πολύ ευρία πλειοψηφία. Ο νέο κώδικα δοντολογία, αποδεικνύει ότι κάνουμε συνειδητέ προσπάθειε για να κατοχυρώσουμε τη σημασία τη προστασία, τη ε, αξιοπρέπεια στον τόπο εργασία. Ω πρόεδρο ε, τη Επιτροπή μα. Είμαι περήφανο για τη δέσμευση των μελών μα και τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει εγκρίνοντα αυτό το σημαντικό έγγραφο. Δεν θα αποδεχθώ κανέναν άλλον εκβιασμό ή αβάσιμε κατηγορίες που έχουν απευθυνθεί κατά τη ε, επιτροπή μας. Οποιοδήποτε έχει θέματα, ας απευθυνθεί στις δικαστικές αρχέ. Παράλληλα με την έγκριση αυτών των δύο κειμένων, αξιοποιώ την ευκαιρία να λάβει υπόψη ένα mail που εστάλει από τον φίλο Γιώργη Πεταδολίτση που με ενημέρωσε ότι δεν μπόρεσε να κάνει επεξήγηση ψήφου στο τέλο τη ψηφοφορία. Έχει δίκιο, Γιώργη. Ο εσωτερικό κανονισμό προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν επεξηγήσει ψήφου μετά την ψηφοφορία και δεν θα πρέπει να υπερβεί το χρόνο που ε, χορηγεί ο πρόεδρο. Επειδή την προηγούμενη φορά είχαμε πολλά θέματα και επειδή οι συντάκτε των τροπολογιών είχαν ήδη εκφραστεί, αποφάσισα να μην χορηγήσω χρόνο για επεξηγήσει ψήφου. Με αυτόν τον τρόπο παραβίασα τα δικαιώματά σα ω μέλου και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ειλικρινά. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα το πιο πολιτικό τμήμα τη δήλωσή μου. Ζούμε σε κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη. Μένουν λιγότερο από 65 μέρε από τι ευρωεκλογέ και λιγότερο από 8 μέρε από την προθεσμία για το Brexit. Και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Αυτό θα έχει επίπτωση στους ε, πολίτες και του Ηνωμένου Βασιλείου και ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επηρεάσει και την προεκλογική εκστρατεία. Η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο και μεθαύριο έχει πολύ σημαντικά θέματα. Εργασία, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμένου για το 2019 και μια πρώτη συζήτηση για την επόμενη περίοδο του στρατηγικού θεματολογίου της Ένωσης που θα συζητηθεί από το Συμβούλιο τον Ιούνιο. Αλλά επίση ε, την κλιματική αλλαγή, μακροχρόνιο θεματολόγιο μέχρι το 2030, εξωτερικές σχέσεις, κυρίως οι σχέσεις μεταξύ Ένωση και κίνα. Παραπληροφόρηση, προστασία των ευρωεκλογών και η κατάσταση πραγμάτων για τι διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το τι θα συμβεί στη συνέχεια για το Brexit. Ο Γκέορκ Τσάμπα, ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, είπε χθε το απόγευμα, μετά τη λήξη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, και παραθέτω, ο χρόνος ε, λύγει. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θέλουν απαντήσεις, να ξέρουν τι τους περιμένει. Η Ένωση έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν υπάρχει λύση στο σημερινό αδιέξοδο, αυτή η λύση βρίσκεται στο Λονδίνο. Ως Προεδρία κάναμε σημαντικές προσπάθειες, ούτως ώστε η Ένωση να είναι έτοιμη για οποιοδήποτε ενδεχόμενο, ακόμη και άτακτη έξοδο. Δεν έχουμε νέα βέβαια για έτοιμα από την Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου για το Συμβούλιο. Και μάλλον θα υπάρξει και μία ίστατη συνεδρίαση του Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα. Άρα συμφωνώ απόλυτα με τον ε, Υπουργό Τσάμπα. Βεβαίω είμαστε όλοι περήφανοι από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της εκδήλωσής μας στις 21 Φεβρουαρίου. Η κοινωνία των πολιτών για την αναγέννηση και από πλευρά συμμετοχή, την ποιότητα των ομιλιών και προσκεκλημένων, την ε, πολυμορφία των ε, μηνυμάτων αλλά και κυρίως την ε, ορατότητα στα μέσα σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Έχετε στα εγγραφά σας μια σύντομη έκθεση που μπορείτε να αξιοποιήσετε στις δράσεις σας, στις περιοχές σας. Επίσης, τονίζω πόσο πλούσιες ήταν οι επτά συζητήσεις τρογγυλής Τραπέζης το απόγευμα. Σας καλώ να πάτε στον ε, τόπο μας και να δείτε τον εντυπωσιακό κατάλογο προτάσεων που προέκυψαν από τις συζητήσεις αυτές στρογγυλής τραπέζης. Όλο αυτό το υλικό μπορεί να στηρίξει μία έντονη επικοινωνιακή εκστρατεία ε, στην πορεία προς το Σύμπιο, τις ευρωεκλογέ και επέκεινα. Και η επικοινωνιακή μας δουλειά συντονίζεται πολύ καλά από την αντιπρόεδρό μας και τους συνεργάτες της. Στην εκστρατεία αυτή ενισχύσαμε τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ τον Πρόεδρο Ταγιάννη για αυτή την ε, εδρεωμένη και επιτυχή συνεργασία στον τομέα της επικοινωνίας. Τώρα πολλά κόμματα και ηγέτες παρουσιάζουν ε, το εκλογικό τους πρόγραμμα για τις ευρωεκλογές και συμμετείχα σε κάποιες τέτοιες συζητήσεις. Επίσης, δράτω με τις ευκαιρίες, όπως θα είδατε σε διάφορες εφημερίδες χωρών της Ένωσης, για να απαντήσω στην επιστολή του Προέδρου Μακρόν προς τους πολίτες της Ένωσης, με τον τίτλο «Για μια Ευρωπαϊκή Αναγέννηση». Πολύ καλό είναι να έχουμε εμπνευσμένου τίτλους. Καλό είναι που εμπνεύσαμε εμείς αυτό το τίτλο. Δεν θα ζητήσω δικαιώματα. Στην ε, επιστολή μου λέω ότι η αναγέννηση είναι το μέλλον. Και στην απάντησή μου ακριβώς αυτή παρουσιάζω το κύριο περιεχόμενο της εκδήλωσής μας στην 21η Φεβρουαρίου. Την προηγούμενη Παρασκευή ήμουνα στο Βουκουρέστι για τη συνάντηση κορυφής των πόλεων και περιφερειών της Επιτροπής Περιφερειών. Ο τίτλος της ήταν πολύ κοντά στο δικό μας ανανέωση της Ευρώπης. Συμμετείχαν πάνω από 1.200 συμμετέχοντες από όλες τις γωνιές της Ευρώπης και την Παρασκευή ενέκριναν μια πολύ κατηγορηματική δήλωση του Βουκουρεστίου η οποία δόθηκε στον ε, πρόεδρο Ιωάννης. Δέκα σημεία όπου αναφέρεται η ανανομένη Ευρώπη χρειάζεται τις περιφέρειες, τις πόλεις και την κοινωνία των πολιτών στη δημόσια δήλωσή μου στον τύπο μαζί με τον Καρλ Χάιντ Λάμπερτς είπαμε ότι μπορείτε να βασιστείτε και σε εμά. Όπω και εμεί ξέρουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε σε εσά. Σήμερα έχουμε την ε, τελευταία ολομέλειά μα πριν από την ε, συνάντηση κορυφή στο Σύμπιου. Έχουμε πολλέ σημαντικέ γνωμοδοτήσει για το μέλλον τη Ευρώπη στην μέση διάταξή μα. Ε, παραπληροφόρηση, δημοκρατία, δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για να ψηφίσουν, πολιτική συνοχή, εκπαίδευση, η ειρήνη, η πρωτοβουλία για να σταματήσει ο εξτρεμισμός και η συζήτηση με τον πρόεδρο Περνοσκόνη για το μέλλον της Ευρώπης. Και το πολύ σημαντικό θέμα, η γνωμοδότηση που αποφασίσαμε να εκπονήσουμε και να αποστείλουμε στη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του ΣΥΜΠΙΟΥ. Ο τίτλος είναι «Να ακούσουμε τους πολίτες Ευρώπης για ένα βιώσιμο μέλλον». Θέλω να συγχαρώ τους συγητές αυτής της νομοδότησης. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή ε, έκανε έντονη προσπάθεια για αυτή τη διαδικασία. Όταν διαβάζω το σχέδιο γνωμοδότησης, καταλαβαίνω ότι οι συγητές ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση ενός ε, φιλόδοξου πονήματος. Ε, το κείμενο είναι πολύ καλό. Αγαπητοί Βλαντιμίρ, Πίτερ και Ήβε, υπό την Προεδρία του Εμμανουέλ. Εσείς και με τη βοήθεια και πολλών άλλων συναδέλφων υποβάλλατε ένα κείμενο το οποίο είναι και ισορροπημένο και φιλόδοξο. Το κείμενο είναι ισορροπημένο γιατί υπάρχει μια δυναμική ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών και τα δύο σε ένα βιώσιμο πλαίσιο. Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ουσιώδης και πρέπει να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν έναν ισχυρό βιώσιμο ρόλο στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας. Επίσης, πρέπει να έχουμε ισχυρή φιλοδοξία για μια κοινωνική Ευρώπη. Έτσι καταλαβαίνω εγώ την έκκλησή σας για μια νέα κοινωνική κατάσταση που να ευνοήσει όλους τους πολίτες προσφέροντάς τους μια πιο δίκαια κοινωνία. Και επίσης τονίζεται ότι η Ευρώπη πρέπει τάχιστα να υιοθετήσει ένα βιώσιμο θεματολόγιο. Καλείται επίση για μια φιλόδοξη υπεράσπιση των θεμελιωδών αξιών μας. Ε, η ειρήνη, η δημοκρατία, θεμελιώδεις αξίες, κράτος δικαίου. Αυτά πρέπει να συνεχίσουν να είναι στο πυρήνα της περαιτέρω εξέλιξης του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και πολιτικών. Και η Επιτροπή μας θα πρέπει να παίξει τον ουσιώδη ρόλο της για να συνδέσει την Ευρώπη με του πολίτε. Βεβαίω πρέπει να τον αναγνωρίσει καλύτερα η Ένωση, να τον αναγνωρίσει καλύτερα αυτό το ρόλο. Και πρέπει να υπάρξει σαφή ανάγκη τους επόμενου μήνες και χρόνια και εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ουσιώδεις να εισαγάγουμε ουσιώδεις καινοτομίε, γιατί έχει αλλάξει πολύ η διαδικασία επαφής και διαλόγου με τους πολίτες. Πρέπει λοιπόν και τα επόμενα χρόνια να ηγηθούμε, να διατηρήσουμε αυτό το ρόλο δίδοντας ακόμη περισσότερη σημασία και ορμή στο διάλογο με τους πολίτες. Είναι ένα πολύ καλό κείμενο αυτό, μια πολύ καλή βάση, ούτω ώστε η Επιτροπή μας να στείλει σαφή και απαραίτητα μηνύματα προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και εν ώψη των ε, ευρωεκλογών. Και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αφού θα εγκρίνουμε το κείμενο αυτό σήμερα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε το μήνυμά μας να περάσει, να εισακουστεί και γιατί όχι επίσης να εφαρμοστεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ζητήσω τους ε, τρεις ηγητές, Βλαντιμίρα Ντορμπάλοβα, Πίτερ Σμιτ και Ιβ Σομβίλ, να έρθουν εδώ για να πάρουν τον λόγο, για να παρουσιάσουν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 The, the, gender fairness. Ladies first. Ισότητα των φίλων. Οι κυρίες προηγούνται. Ό,τι θέλετε εσείς, όπως θα συμφωνήσετε μεταξύ σας. You agreed. Τι έχετε κανονίσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, Λούκα. Ευχαριστώ, Λούκα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ότι δεν σεβόμαστε τη σειρά ή δεν θέλουμε να αφήσουμε πρώτα τις κυρίες, αλλά συνεννοηθήκαμε να αρχίσω εγώ με την παρουσίαση αυτή του θέματος και γνωμοδότηση να κάνω κάποιες εξηγήσει έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα σε ποιο πλαίσιο βρισκόμαστε και έχουμε εκπονήσει αυτή τη γνωμοδότηση. Πριν αρχίσω όμως, θα ήθελα στην αρχή, στην αρχή όχι στο τέλος, να πω δύο λόγια για την αγαστή συνεργασία που είχαμε στην ομάδα εργασίας υπό την ε, αιγύδα της Εμμανουέλ που καταφέραμε τελικά να καταλήξουμε σε πολύ καλά αποτελέσματα και ήταν και πρόκληση όλο αυτό. Για ποιο λόγο. Διότι, αν δεν απατώμε, την 1η Φεβρουαρίου ε, μας εξέλεξαν οι ομάδες μας και μας ανέθεσαν μέσα σε τέσσερις εβδομάδες να εκπονήσουμε ένα έγγραφο για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, και αυτή δεν είναι καθόλου απλή πρόκληση, πόσο μάλλον όταν έχει τέσσερι εβδομάδε. Γιατί τη χαρακτηρίζω πρόκληση, διότι δυστυχώ δεν είχαμε την ευκαιρία λόγω χρόνου να πάμε και στις επιμέρους ειδικέ ομάδες για να συζητήσουμε με όλες τα θέματα που τους απασχολούν και είναι αρμοδιότητά τους. Ήταν πολύ στενό το χρονικό περιθώριο που είχαμε και δεν καταφέραμε να εκπονήσουμε ένα έγγραφο για το μέλλον της Ευρώπης και για τις δικές μας θέσεις στην ΕΟΚΕ. Άρα, έχουμε ε, κερδίσει το δικαίωμα να έχουμε ένα επίδομα ε, βαρέας και ανθυγινής εργασίας, τουλάχιστον στο γερμανικό εργασιακό δίκαιο υπάρχει αυτό. Όταν έχεις βαρύ ανθυγινό επάγγελμα, δουλεύεις νύχτα, Σαββατοκύριακο, θα δούμε, θα το διαπραγματευτούμε αυτό με τον πρόεδρο. Πώς έχει τώρα η δομή και η διάρθρωση του εγγράφου. Ε, θα το έχετε διαπιστώσει ότι ακολουθεί το θεματολόγιο της αηφορίας στην Ευρώπη. Γιατί είπαμε ότι αν θέλουμε να συζητήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης, πρώτα αυτή θα πρέπει να είναι μια βιώσιμη αηφόρος Ευρώπη και μια Ευρώπη που να έχει ένα ηγετικό ρόλο παγκοσμίω για τη βιωσιμότητα και την αηφορία. Διότι διαπιστώνουμε ότι σε μερικά επίπεδα αυτό δεν είναι ακριβώς όπως θα επιθυμούσαμε. Για όλους εκείνους που θα διαμαρτυρηθούν ότι είναι πάρα πολύ μακροσκελές το κείμενο αυτό, γιατί ήδη έχω δεχτεί κάποιες κρούσεις, θέλω να σας πω ότι σε περίπτωση που καταλήξουμε σήμερα σε ένα κοινό έγγραφο, στο, για το τέλος έχουμε προετοιμάσει ένα δισέλιδο το οποίο θα περιλαμβάνει και θα παρουσιάζει τα όσα θα αποφασίσουμε. Και στο συμπίου αλλά και επέκεινα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό, γιατί το έχουμε συμφωνήσει οι τρεις μας. Και πάντα με την πρόεδρο, αν μου επιτρέψεις να το πω, Εμμανουέλ, ότι αυτό το έγγραφο είναι και λίγο πολιτικό ε, θέσεων και στρατηγικής για το μέλλον και της ίδιας μας της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής. Άρα θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο αυτό. Και δανείζομαι τα λόγια της Βλαντιμίρα ε, να δημιουργήσουμε πρώτα την πηγή. Η πηγή είναι όλο αυτό το έγγραφο. Και από την πηγή μετά έχουμε την κεντρική ιδέα που παρουσιάζει ε, πολύ ευσύνοπτα και συγκεκριμένα τα πολιτικά μηνύματα. Ε, δεν μπορέσαμε να εξεργαστούμε την κάθε λεπτομέρεια, αλλά στην πολιτική διαδικασία στην Ευρώπη τα πολιτικά μηνύματα είναι αυτά που θέλουμε να ε, συμπεριληφθούν. Και όπως λέει και η επικεφαλίδα μας, θέλουμε να αφογκραζόμαστε τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί από από την ε, οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, εμείς από τη φύση μας την ίδια, ε, έχουμε τη δυνατότητα να αφουγκραζόμαστε στους πολίτες. Και μιλούμε για μια Ευρώπη κοινωνική, την Ευρώπη των πολιτών, ένα υφόρο περιβάλλον και μια βιώσιμη οικονομία. Και δίκαιη φορολόγηση. Είχαμε και το θέμα της μετανάστευσης και προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα και προσανατολιστήκαμε στις ε, ήδη ε, ψηφισμένες νομοδοτήσεις. Αλλά προχωρούμε και λίγο παραπέρα από ό,τι ε, έχει συζητήσει η Επιτροπή μας και έχει εγκρίνει ως νομοδοτήσεις. Γιατί πιστεύουμε ότι το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί πλέον να το χειριζόμαστε όπως το παρελθόν. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι. Εκπονήσαμε λοιπόν αυτό το έγγραφο. Ο καθένας πρόσφερε τη δική του συνεισφορά, ισότιμα, ω ηγητή. Έχουμε και 17 τροπολογίες και σε μερικέ από αυτές συμβιβαστικέ προτάσεις. Σε κάποιες άλλες είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούμε ένα συμβιβασμό. Α, μου λέει ο πρόεδρο πρέπει να τηρήσω το χρόνο μου. Τρία λεπτά δεν είχα, όχι, όχι, γιατί κάτι τέτοιο άκουσα. Εν πάση σταματώ εδώ και ε, αναλαμβάνει η Βλαντιμίρα τώρα. Πέντε λεπτά έχει κάθε εισηγητή. Και τα ξεπέρασε. You should imagine. Βλαντιμίρα, five minutes. Βλαντιμίρα, πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Έχουμε εδώ συνεννοηθεί ώστε να είμαστε ουδέτεροι ως προς την επιλογή των φίλων και την ισότητα. Θα συνεχίσω λοιπόν από εκεί που σταμάτησε ο Πέτερ. Το όλο κείμενο είναι καρπός της δουλειάς της ομάδας μας, όπου συνεισφέραμε όλοι ισότιμα. Δεν διαιρέσαμε τα μέρη του κειμένου ανάλογα με τις απόψεις των τριών ομάδων, διότι θέλαμε να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τη Σύνοδο του Συμπίου και να περιλάβουμε και κάποιες συστάσεις. Σε αντίθεση λοιπόν με τις κλασικές γνωμοδοτήσεις, δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα. Θέλαμε κάτι διαφορετικό να καταφέρουμε εδώ. Θέλαμε ένα ξεκάθαρο κείμενο. Είναι χαρά μου που καταφέραμε να βρούμε και συμβαστικέ λύσεις. Η δουλειά μας έγινε με πνεύμα καλής συνεργασίας. Ο μόνος μας εχθρός ήταν το ρολόι. Και για να συντομεύω, αυτό που τώρα θέλω οπωσδήποτε να πω είναι ότι το βασικό μας μήνυμα είναι να δούμε τι χρειάζεται η Ευρώπη στο μέλλον. Τι θέλουμε δυνατή και βιώσιμη την Ευρώπη. Γι' αυτό επικεντρωθήκαμε στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Και πέραν αυτού, Έχουμε συμπεριλάβει και κάποιους παράγοντες που θεωρούμε σημαντικούς για την βιωσιμότητα ακριβώς της Ευρώπης. Στα συμπεράσματα και ολοκληρώνοντα και εγώ την παρέμβασή μου, να πω ότι χαίρομαι πολύ που οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει επίση αναφέρονται και έχουν τη θέση του στην όλη διαδικασία τη βιώσιμη Ευρώπη. Θέλουμε ακριβώ να δώσουμε έμφαση στο ρόλο των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, διότι στο μέλλον θέλουμε να θαρρύνουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εταιρείε να βρεθούν στην εμπροστοφυλακή της βιωσιμότητας και μάλιστα να γίνουν και παγκόσμιοι πρωταγωνιστές. Να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές μου για την άριστη συνεργασία μας και τον πρόεδρό μας ο οποίος ε, στάθηκε ουδέτερος ε, στην καθ' τη διάρκεια της σύνταξης της νομοδότησης για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πραγματικά ήταν ε, εκπληκτικό ότι πετύχαμε να έχουμε συνένεση ε, παρόλο που κάποιες τροπολογίες τις λάβαμε αλλά θα τις συζητήσουμε αργότερα και πιστεύω ότι το έγγραφο αυτό βασίζεται στη συνένεση. Ευχαριστώ Βλαντιμίρα. Τελευταίος ο Ιβ Σομβίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές μου και την Πρόεδρο που πραγματικά ε, δείχνει με τρόπο αντικειμενικότατο τις συζητήσεις και μας βοήθησε να καταλήξουμε σε συνένεση. Ευχαριστώ τους την εμπειρογνώμονά μου για κάποιες από τις συνεισφορές της και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Πατρίκ Φεύ και στους ε, συναδέλφους του, ιδίω την Γιούμπια. Ευχαριστώ λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε, την υπομονή σας και την αποτελεσματικότητα. Ήταν σημαντικό να υποθεί και αυτό. Επειδή είμαι ο τρίτος που τοποθετείται, δεν έχω τίποτα να πω. Απλώς μια δική μου παρατηρήση, ένα σχολιασμός, αν επιτρέπετε. Χθες ξαναδιάβαζα το Ευρωβαρόμετρο του 2018 και εντόπισα τρία στοιχεία που είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει αφοσίωση στον ευρωπαϊκό σκοπό, μετά ότι πρώτα είναι η ησυχία των Ευρωπαίων είναι το μεταναστευτικό, δεν μα εκπλήσει, και μετά ότι αναδεικνύεται ω πρώτη προτεραιότητα το κλίμα. Σε ό,τι αφορά την ε, αφοσίωση στον ε, σκοπό τη Ένωση τη Ευρώπη. Εδώ ε, με εξέπληξε ότι 62% των ε, ερωτηθέντων της Ευρώπης των 28 πέρσι είπαν ότι το να είναι κανείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλό για τη χώρα τους. Είναι τα καλύτερα αποτελέσματα που είχαμε ποτέ από το 1983. Τώρα βέβαια όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και στη σχετική τους διάσταση, δηλαδή τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης ε, βορρανό του Ανατολής Δύσης. Και όλα αυτά για να πω ότι στην επικοινωνιακή μας πολιτική προσεχώ, όταν θέλουμε να προασπιστούμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα και να δείξουμε τι έχουμε πετύχει ως τώρα και τι επομένει ακόμα να πετύχουμε, να κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και βεβαίω να προσαρμόζουμε την προσέγγιση μα ανάλογα με τι καταστάσει. Μετά για τη μετανάστευση. Δεν θα σα ευνηδιάζει που βλέπετε ότι είναι το πρώτο που ανησυχεί ε, του Ευρωπαίου με το 50% των ερωτηθέντων τουλάχιστον να λένε ότι είναι ένα μείζονο σημασία ζήτημα και μετά θέματα όπω οικονομική ανάπτυξη, η καταπολέμηση τη ανεργία των νέων, η καταπολέμηση τη τρομοκρατία του απασχολούν. Κάθε φορά βλέπουμε ότι τα ποσοστά αυξάνονται στα κράτη-μέλη. Ιδίω αυτά που τα πλήττει το φαινόμενο. Ε, πέραν των γεωγραφικών διαφορών όμω, βλέπουμε ως προς τη μετανάστευση ότι και η ένταση των απαντήσεων αλλάζει με το χρόνο. Δηλαδή το 2012 ω προς τη μετανάστευση θεωρεί το σημαντικό από 8% των ερωτηθέντων το θέμα βλέπετε πώς έχει ενταχθεί πλέον στην οτροπία μας και στη σκέψη μας. Και μετά αναδεικνύεται και το θέμα του κλίματος ως πρώτη της σημασίας. Ούτε αυτό μας εκπλήσει, διότι το θέμα αυτό ε, μεταξύ του Ιανουαρίου 2018 και του Σεπτεμβρίου 2018 κέρδισε πέντε ποσοστιαίες μονάδες στις δημοσκοπήσεις ως πλέον σημαντικό θέμα ή έστω σημαντικό. Με διαφορά πάλι μεταξύ Βορανότανα Δύσης και η κατάσταση κυμαίνεται βέβαια τα ποσοστά κυμαίνονται. Πρέπει όμω και αυτό να το εντάξουμε στην όλη μα μελέτη. Και το τελευταίο που θέλω να σα πω σε σχέση με όσα διάβασα χθε είναι η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Συστήματο. 46% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι με το δημοκρατικό σύστημα τη Ευρώπη. 9 ποσοστιαίε μονάδε σε, παραπάνω σε σχέση με τα εθνικά του ε, δημοκρατικά όργανα. Και εδώ βεβαίω υπάρχουν διακυμάνσει μεταξύ των κρατομέλων. μελών. Γιατί τα αναφέρω τα αποτελέσματα αυτά τώρα. Γιατί θέλω να αναδείξω τη δουλειά που κάναμε ω προ την ε, προσέγγιση των πολιτών που προσπαθήσαμε και θα πρέπει βεβαίω να κάνουμε την κατάλληλη διάκριση μεταξύ των κρατών μελών ή των διαφορετικών ευρωπαϊκών περιοχών. Πάντω, σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω ότι όλοι εδώ είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό, μπορεί να εντατοκοποιήσει την ε, αλληλεπίδραση και την επικοινωνία τη με του Ευρωπαίου πολίτε για να του εντάξει στην ε, προσπάθεια ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώνω πρώτα εντό ολίγου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει έναν ε, καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει. Θέλω να επιμείνω στο γεγονό ότι ο ρόλο αυτό, ο ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ε, είναι μια δουλειά κοινή. Ε, έτσι θα κοινοποιήσουμε μόνο του πολίτε. Και θέλω να πω τα εξή στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, ακρόαση, μετά διάλογο, μετά σαφήνεια του μηνύματο, ε, στοιχεία χειροπιαστά και όχι top-down, από πάνω προ τα κάτω. Ε, προσέγγιση. Αυτά είναι τα πέντε βασικά στοιχεία. Συζητήσαμε το περιεχόμενο λοιπόν με του δύο συνεισηγητέ και χθε μόλι, αλλά νομίζω ότι με την γνωμοδότηση που υποβάλλουμε θα ευνοήσουμε καλύτερα το κλίμα για ένα τέτοιο διάλογο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ιβ. Α περάσουμε και στα ε, λογιστικά τώρα. Μετά την παρέμβαση του Ιβ, ανοίγει η συζήτηση. Θα έλεγα δύο λεπτά στον καθένα. Εκτός των εξαιρέσεων της κυρίας Μπαταστούφ που ήταν ε, η πρόεδρος της ομάδας. Για να παραμένουμε στα 21 λεπτά που προβλέπονται για αυτό το θέμα. Έχετε το λόγο, κυρία μου, για τρία λεπτά και οι υπόλοιποι δύο. Ε, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, καλοσύνη σας. Τρία μηνύματα ένα για το πλαίσιο, τα αποτελέσματα και το μέλλον. Για το πλαίσιο προετοιμασίε αυτή τη έκθεση, τη νομοδότηση όλα υπόθηκαν, είχαμε πολύ λίγο χρόνο. Τρει συνεισηγητέ ε, με έντονε προσωπικότητε, άρα η διαχείριση ήταν όντω δύσκολη. Υπήρξαν ε, πολύ έντονε συζητήσει. Πραγματικά ο καθένα να παρουσιάζει με ένταση τι απόψει του. Και είχαμε τη φιλοδοξία να παραγάγουμε ένα κείμενο πολιτικού χαρακτήρα το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το κείμενο των 17 σελίδων. Δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω ότι έχει όντως μια πνοή. Και ο βασικός στόχος ε, αναφέρεται στην παράγραφο 1-1. Ζητάμε ότι λίγο ούτε πολύ η Ευρώπη να γίνει η πρώτη βιώσιμη δύναμη στον κόσμο. Έχουμε, για παράδειγμα, λιγότερη επιφάνεια από τον Καναδά και τη Ρωσία, έχουμε λιγότερο πλαισμό από την Κίνα, έχουμε λιγότερες φυσικές, ε, λιγότερους φυσικούς πόρους από τη Ρωσία, αλλά θέλουμε να είμαστε η πρώτη βιώσιμη δύναμη στον κόσμο. Και με βάση τους τρεις πυλώνες, ε, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Να είμαστε πρώτοι τελικά που θα εντάξουμε στο σύνολο των πολιτικών μας, εσωτερικών και εξωτερικών, το θεματολόγιο του ΟΗΕ. Πιστεύω ότι αυτά τα θέματα θα μπορέσουμε να τα προωθήσουμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτή είναι η εντολή που δίνουμε στις νέες θητείες. Είδατε τα παραδοσιακά κεφάλαια, δημοσιονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αλλά υπάρχουν και δύο πρωτότυπα, νέα στοιχεία. Πρώτη, τρόπος παρουσίασης. Είναι δύσκολο να ανανεώσουμε από πλευρά ε, παρουσίας των αλλά παρόλα αυτά σε κάθε κεφάλαιο θέλουμε να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ των γενικών αρχών και κατόπιν ε, σε ένα πλαίσιο θελήσαμε με συγκεκριμένα υποσημεία, με κουκίδες μπροστά, να βάλουμε τις κυριότερες προτάσεις. Και θα δείτε και διάφορες παραγράφους κατόπιν που αφορούν την επικοινωνιακή μας πολιτική, την ευαισθητοποίηση των ε, συμπολιτών μας και ένα κεφάλαιο για τους λαούς και τους πολίτες της Ευρώπης. Με αυτού θέλουμε απευθεία να έρθουμε σε επαφή. Και τέλο μία επιθυμία για το μέλλον. Ελπίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι ο πρόεδρο ε, θα κάνει να ακουστεί η φωνή, η φωνή μας στο Συμπίου. Ελπίζουμε, ελπίζουμε η φιλοδοξία να γίνουμε η πρώτη βιώσιμη δύναμη στον κόσμο να εφαρμοστεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ελπίζουμε να έχουμε την κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική με τις κατάλληλες μορφές και ελπίζουμε στην επόμενη θητεία τα θεσμικά όργανα να εμπνευστούν από την πλατφόρμα αυτή, την φιλόδοξη που προτείνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Εμμανουέλα. Γιάτσε Κράτσικ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτό που είπε η μόλις τώρα. Συγχαίρω τους ε, εισηγητές μας Καταλαβαίνω ότι ε. επιτυχάνουμε συμβασμούς για αυτό το σημαντικό θέμα και επειδή συμβαίνουν ε, τόσα πράγματα γύρω μας στην Ευρώπη αυτές τις μέρες το ότι καταλήξαμε σε κοινή θέση για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης κορυφής είναι κάτι το πολύ σημαντικό και χαίρομαι που ανταποκριθήκαμε σε αυτό το καθήκον. Ευχαριστώ λοιπόν τους ηγητές, ευχαριστώ τον Πρόεδρο και ευχαριστώ και τις τρεις ομάδες για την καλή συνεργασία για το θέμα αυτό. Νομίζω καταφέραμε να ε, μείνουμε κατά μέρος άλλων συζητήσεων στην Επιτροπή για να μπορέσουμε να καταλήξουμε με αυτή τη συνεισφορά για το πρόγραμμα εργασιών της νέας Επιτροπής και για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Η γνωμοδότηση αυτή αναφέρει πολλά από όσα ήδη έχει κάνει η Επιτροπή μας και αυτά επί των οποίων έχουμε μέχρι στιγμής συμφωνήσει. Και αξιοποιώ την ευκαιρία καταλήγοντας να κάνω έκκληση προς όλους μας να καταλήξουμε και με ένα ψήφισμα μέχρι το τέλος της επόμενης Ολομέλειας ίσως, ούτως ώστε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τις επικείμενες ευρωεκλογές. Ευχαριστώ και πάλι για τη θαυμάσια εργασία σας, για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και είμαι πεπισμένο ότι θα υπερψηφιστεί. Σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιάντσεκ. Άντε Μιλέν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές ανισότητες οξύνονται μεταξύ κρατών μελών και εντός. Οπότε αυξάνονται και ανησυχίες για το μέλλον του πλανήτη μας, για ενδεχόμενες νέες οικονομικές κρίσεις και χρηματοπιστωτικές και άρα πρέπει να δώσουμε ακριβή και ισορροπημένο ορισμό του τι θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα είναι κάτι το θεμελιώδες. Ουσιώδες για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη οι συμπολίτε μας που είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί έναντι της δράσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και γενικότερα η πολιτική, άνδρες και γυναίκες και ελπίζω να αποτελέσει πηγή έμπνευσης στο συμπίου φυσικά αλλά και για τα προγράμματα εν ώψη των εκλογών των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και την περαιτέρω δράση τους. Αλλά πρέπει επίσης να είναι κάτι το οποίο να έχει απήχηση και πέρα των ε, συνόρων μας πρέπει να συνεχίσουμε να ηγούμεθα τις προσπάθειες προς πιο προς ε, κοινωνίες με πολύ λιγότερες ανισότητες στα πλαίσια των νέων συνθήκων. Πολύ ενδιαφέρουσα εργασία και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αν. Λουτς Ρίμπε, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ να συγχαρώ τους τρεις ε, εισηγητές. νομίζω ότι περιέχει ισχυρά, ισχυρότατα μηνύματα. Το 2-1 για παράδειγμα. Οι πολίτες της Ευρώπης, άνδρες και γυναίκες, ε, θεωρούν όλο και λιγότερο την Ευρώπη ως λύση και όλο και περισσότερο ως πρόβλημα. Το υπογραμμίζω αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτή είναι η επίκρισή μου θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα για να περιγράψουμε γιατί όμως σημαίνει αυτό. Και να πω το εξής. Αισθάνομαι ότι η Ευρώπη δεν εκπληρεί τις υποσχέσεις της. Κοιτάξτε πόσο έχουν υποσχεθεί πολιτικοί στην Ευρώπη, που δεν τηρήθηκε μετά. Είναι μακροσκελέστατος ο κατάλογος και με λυπεί. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ο τίτλος του λέει «Να ακούσουμε τους πολίτες». Στην τελευταία Ολομέλεια ήμουν στο νοσοκομείο και παρακολουθούσα τη συζήτηση στο ίντερνετ και είδα πως ακούσαμε τους νέους για το, την κλιματική αλλαγή. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι ναι, νέοι ικανοποιήθηκαν. Γιατί τον ακούς δεν σημαίνει ότι και κατανοείς. Δηλαδή πρέπει να βρούμε άλλες διαδικασίες. Και καταλήγω. Και κάτι που, για το οποίο πρέπει να επικρίνω τους ΣΥΤΑΣ. Ένα τόσο βασικό κείμενο να είναι ε, αυτή η τελευταία στιγμή. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ακούσουμε τον εαυτό μας. Οι διαδικασίες για κάθε γνωμοδότηση να μην συζητιούνται και στις ε, επιμέρους ειδικέ ομάδες. Θα έπρεπε να έχει υπάρξει περισσότερη συμβολή στην κατάρτιση του κειμένου και ελπίζω για τέτοια βασικά κείμενα να έχουν περισσότερο χρόνο στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ είναι δύο λεπτά. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους τρεις συγγητές για το έργο τους. Είναι πολύ καλό να έχουμε τέτοια γνωμοδότηση με τόσο σαφή μηνύματα για θέματα που μας απασχολούν τακτικά στο Κοινοβούλιο αλλά αποφεύγουμε να τα αναφέρουμε με τέτοια σαφήνεια και χαίρομαι που πλέον είμαστε τόσο σαφείς ε, για τη βιωσιμότητα και ε, για τα θέματα του ανταγωνισμού και της εσωτερικής αγοράς. Εκεί θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση ακριβώς και το γεγονός ότι κατάφεραν τρεις ομάδες να συμφωνήσουν για τον εισηγητών του σε μια κοινή θέση ενωμένοι θα μας δώσει μια πολύ γερή βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά στο μέλλον. Αυτό το καιρό είμαι εισηγητής ε, για την αντίδρασή μας για το έγγραφο θέσεων για τη βιωσιμότητα το 2030. Και αυτή τη στιγμή εγκριθεί από την Ολομέλεια θα είναι και αυτή ε, άλλη μια γερή βάση για τη μελλοντική μας εργασία. Ευχαριστώ και πάλι τους τρεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Ο Στέφαν Μπακ για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι δεν συμμετείχα στην ομάδα εργασίας, αλλά ε, παρόλα αυτά έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ σημαντική η γνωμοδότηση αυτή. Είναι λόγος και για την κλιματική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η κοινωνία με την ευρύτερη έννοια θα πρέπει να συμμετέχει και στην εκπόνηση των δικών μας νομοδοτήσεων. Δεν είχαμε πολύ χρόνο, λίγο χρόνο είχαμε και καταλήξαμε σε πολύ καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Έχω υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες. Δεν θέλω να επικρίνω τα όσα λέει η γνωμοδότηση. Διευκρινιστικές είναι περισσότερο ε, και ε, αφορούν κάποιες παραθέσεις που θα πρέπει να γινόνται με ακρίβεια. Τέτοιου τύπου τροπολογίες έχω υποβάλει. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, υποστηρίζω την γνωμοδότηση και όλο το έργο που γίνεται. Thank you. Ευχαριστώ. Η κυρία Τέλερ Ράχη Λαβώνα. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Εχθές ε, είδα ε, κάτι και ε, είπα ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της βιωσιμότητας και της αηφορίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι στην πρωτοπορία. Οι εταιρείε, οι επιχειρήσει θα πρέπει και αυτές να ε, πρωταγωνιστούν, να καινοτομούν, να επενδύουν και να δημιουργείται ένα καλό περιβάλλον για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλη την κοινωνία, όχι μόνο τους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις. θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι δικές μας επιχειρήσεις και οι κοινωνίες μας ε, θα πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια. Το θέμα δεν είναι να ψάχνουμε ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Ε, μας ενδιαφέρει να είναι αμοιβαία επωφελής αυτή η προσπάθεια, να έχουμε ωφέλη και οικονομικά και ε, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά αξίζει τον κόπο να προχωρήσουμε έτσι και προς την κατεύθυνση αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι οι στόχοι μας θα μπορούσαν να είναι λίγο, πιο φιλόδοξοι ε, από ότι ε, διατυπώνει αυτή η γνωμοδότηση. Και δεν είναι όλα αρνητικά. Δεν θα πρέπει πάντα να εκφράζουμε τη λύπη μας και θα πρέπει να είμαστε πιο θετικοί, πιο αισιόδοξοι ε, αν θέλουμε να έχει αποτελέσματα αυτή η προσπάθεια. Σε 25 ε, χρόνια σταδιοδρομίας ε, που έχω, ε, μπορώ να σας πω ότι δεν πρέπει να είμαστε πάντα αρνητικοί αλλά και θετικοί. Μπορώ να σας πω, λέει ο Πρόεδρος, ότι κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας μπορούμε να κάνουμε βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Όλιβερ Ρόκε για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά την παρουσίαση των τριών συνεισηγητών, είναι σαφές ότι δεν είναι μια κλασική γνωμοδότηση αυτή. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα αυτό της Επιτροπής μας ε, που θα αποσταλεί αν αγκριθεί η γνωμοδότηση. Μιλάμε για μια συνεισφορά ε, σφαιρική και συνολική στο, στη Σύνοδο του Συμπίου και πέρα. Εδώ είναι σαν να έχουμε συντάξει ένα μανιφέστο, ε, μια δήλωση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τους πολίτες. Δεν ήταν εύκολο τρεις συνεισηγητές να συμφωνήσουν, όμως χαίρομαι πολύ που βρήκαν λύσεις και το αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό. Ε, νομίζω λοιπόν ότι το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την ε, δύναμη της επιτροπή μα. Το κείμενο είναι ένας φιλόδοξος ε, τρόπος να προτείνουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τα πλέον επιτυχημένα εγχειρήματα από οικονομικής, κοινωνικής άποψης και άποψης της ειρήνης στην Ευρώπη. Βέβαια περάσαμε και δύσκολες ώρες. Τα κράτη-μέλη καλούνται ε, στο μέλλον αναλάβουν ευθύνε ω προ τη μετανάστευση που έχει αναδείξει την έλλειψη αλληλεγγύη ή να αντιμετωπίσουν τα διέξοδα τη οικονομία. Το ΕΒ πρόκειται να φύγει, ανισότητε εντείνονται μεταξύ των διαφορετικών περιοχών τη Επίρου. Δεν είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε. Θέλουμε μια Ευρώπη διαφορετική. Μια Ευρώπη που να προασπίζεται τι γυναίκε, του νέου και να δημιουργεί ποιοτικέ θέσει εργασία. Για τον σκοπό αυτό θέλουμε ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο μέσω τη γνωμοδότηση αυτή. Θέλουμε ε, δικαιότερη, πιο ισότιμη κοινωνία, να υπάρχει ένα κοινωνικό πρόγραμμα δράση ώστε η Ευρωπαϊκή Ατζέντα 2030 να μεταφερθεί και να ισχύσει σε όλα τα επίπεδα. Συνάδελφοι, δύο μήνε πριν τι ευρωεκλογέ, είναι η στιγμή ω Ευρωπαίοι να υψώσουμε τον αίσθημά μα, να προασπιστούμε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να προτείνουμε ένα φιλόδοξο εγχείρημα με σαφή αιτήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Μπρέντα Κίνγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να προσθέσω τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μου προς τους τρεις συνεισηγητές ε, στην ομοδότηση αυτή και στον πρόεδρο ο στην πρόεδρο η οποία διεύθυνε την όλη δικασία. Ήθελα κι εγώ να μιλήσω για να εκφράσω την υποστήριξή μου, γιατί υπέβαλα μια τροπολογία και ήθελα να εξηγήσω το γιατί. Ε, σε σχέση με όσα ακούσαμε και όσοι εκφράστηκαν, νομίζω ότι είναι πολύ καλή έκθεση, με πολύ ισχυρά μηνύματα, αλλά όπως είπε και ο τελευταίος ομιλητής, Υπάρχει, υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα ε, που συζητιούνται και απασχολούν την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ένα από αυτά είναι η μετανάστευση. Και βλέπω ότι στη γνωμοδότηση όταν φτάνει το θέμα στους μετανάστες, η ευθύνη για την ένταξη βαραίνει μόνο τους ώμους των ίδιων των μεταναστών. Ε, αυτοί αναλαμβάνουν την ευθύνη και επιφορτίζονται με το καθήκον. Είναι δύσκολο να προχωρήσει το θέμα αυτό όταν και να πάει κανείς ελεύθερα προς το μέλλον όταν του βάζουν εμπόδια. Ε, παράδειγμα, ε, όσοι ήρθαν από την Καραϊβική τη δεκαετία του 50 και του 60 προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα είναι όλοι διευθύντες των σπιτιών τους. Γιατί? Γιατί συνεργάστηκαν. Ε, γιατί όταν ήθελαν να νοικιάσουν υπήρχε η πινακίδα όχι μαύρη, όχι Ιρλανδοί, όχι σκύλοι. Ε, δεν μπορούσαν να βρουν Βρετανοί ιδιοκτήτες και με τους Ιρλανδούς ε, στην ΠΑΜΠ ακούγαμε να λένε ότι υπήρχαν άνθρωποι που προτιμούσαν να νοικιάσουν σε μαύρο και σε σκύλο από ότι σε Ιρλανδό, ας πούμε. Ε, ανάλογα λοιπόν με τη γειτονιά, ανάλογα με την περιοχή, ήταν πολύ δύσκολο να ενταχθεί κανεί τότε. Άρα οι ευθύνε υπάρχουν αμφίδρομα, και τις, ε, μάλλον ένθεν και ένθεν, και από τι δύο πλευρέ. Γι' αυτό υπέβαλα αυτή την τροπολογία και ελπίζω να γίνει δεκτή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Μπρέντα, ο Σάιμον Μπόλαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ και να επενέσω τους τρεις συνεισηγητές και την πρόεδρο της ομάδας. Και εγώ θα συμφωνήσω με όσα είπε η Μπρέντα Κίνγκ ως Ιρλανδός. Κάτι ξέρω κι εγώ γι' αυτά. Να πω απλώς ότι η έκθεση όντως είναι μια καλή έκθεση με ισχυρά μηνύματα. Θα πρέπει να την λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά. Έχουμε, έχουμε όμως και κάποιες μικροαντηρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακούμε οι μεν τους δε, αλλά κάποιες φορές ζούμε και σε, μια, ε, χρυσή, σε ένα χρυσό κλουβί. Εάν πάει κανείς στην Ιρλανδία και αρχίσει να μιλάει με τον κόσμο για τη βιώσιμη αλλαγή, Εγώ άκουσα τους πολίτες και η σύσταση που μου λείπει αυτή την έκθεση είναι αυτή για τη φτώχεια. Αυτή έπρεπε να είναι πιο δυνατή και ισχυρότερη. Δεν κάναμε αρκετά ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκριζώσουμε και να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Έχουμε την περίφημη συμφωνία του 2020, αλλά δεν κάναμε αυτό που έπρεπε. Και επειδή δεν το καταφέραμε, το αγνοούμε τελικά. Τη βιώσιμη αλλαγή και την βιωσιμότητα θα την πετύχουμε μόνον εάν ε, χτυπήσουμε τη φτώχεια. Ε, μπορεί να λέει κανείς ότι ε, υπάρχουν ε, αντιρρησίες της, ε, αυτοί που έχουν αντιρρήσεις προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, ότι είναι λαϊκιστές και ούτω καθεξής. Όμως εγώ πολύ φοβάμαι ότι στην ουσία θα δημιουργήσουμε περισσότερη φτώχεια. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι λέμε στα πλαίσια αυτής της συζήτησης. Πρέπει να ακούμε λίγο καλύτερα τους πολίτες, διότι εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ακούμε όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Και πρέπει να σκεφτούμε και την αρχή του 20 και του 60. 20 είναι υπέρ της Ευρώπης, 20 την πιστεύουν, το 60% όμως είναι τελείως κατά. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πολύ, Σέμος. Ελπίζω ακόμα να είμαστε σε θέση να διευρύνουμε τη δυνατότητά μας να αφουγκραζόμαστε, να βλέπουμε, να παρατηρούμε. Θα ξαναδώσω το λόγο στους εισηγητές μας για να απαντήσουν. Ποιος θα μιλήσει πρώτος. Don't Καλά, μην κάνετε τρία λεπτά να αποφασίσετε τώρα. Ε, με την ίδια σειρά. Ευχαριστούμε πολύ, ε, κύριο Σμιτ, για τα σχόλιά σας. Βεβαίως, ήταν περιορισμένος ο χρόνος. Γι' αυτό δεν θα τα βρείτε όλα στο έγγραφο αλλά έχει σημασία. Κάποιος είπε προηγουμένως ότι αυτή είναι η αφετηρία και η βάση. Και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουν διάφορα κεφάλαια, συστάσεις, από κοινού θα τα αναπτύξουμε όλα αυτά. Πηγαίνουμε σε διάφορους τομείς και τώρα πώς αυτό θα ε, συγκεκριμενοποιηθεί θα το δούμε κατά τη διάρκεια της βιώσιμης αυτής πορείας. Έχουμε και τις τροπολογίες και θα σας παρακαλούσα να μας υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντορμπάλοβα. Βασικά, επένους ακούσαμε από πλευρά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα κείμενο πολιτικό η γνωμοδότηση αυτή και ήλπιζα ότι θα έβρισκε τη συμφωνία σας. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι ένα κείμενο 17 σελίδων που αποτελεί τη βάση για τη συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει και θα αποτελέσει πηγή έμπνευση. Έχουμε συστάσεις για όλα τα κεφάλαια, αλλά συμπερασματικά θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που είπε προηγουμένως ο κύριος ε, Βέβερ ότι δεν θα πρέπει απλώς να φουγκραζόμαστε τους πολίτες, αλλά και να κατανοούμε αυτά που μας λέγουν. Λοιπόν, είναι ένα πρώτο βήμα, αυτό που προσπαθούμε να τους ακούσουμε και όπως είπε και ο Σίμους, θα πρέπει να φουγκραζόμαστε καλύτερα, πιο προσεκτικά και Ελπίζουμε να τους κατανοούμε καλύτερα στο μέλλον από ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα και ελπίζω να στεφτεί με επιτυχία η γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, λέει κύριος Σομβίλ. Οι, οι τρεις συνεισηγητές εδώ θέλαμε να προχωρήσουμε πιο πολύ, αλλά είχαμε ήδη ένα μακροσκελές κείμενο, οπότε δεν μπορέσαμε να το αναπτύξουμε να απαντήσω σε κάποιες παρεμβάσει στο Λούτς, τον κύριο και που μίλησε για μανιφέστο. Για το Λούτς βεβαίω είναι ένα έγγραφο στρατηγικής και θα έλεγα με δύο λόγια τώρα αρχίζει η δουλειά. Και είναι πρόγραμμα εργασία για τους επόμενους μήνες, για τα επόμενα έτη για την Επιτροπή μας. Και ελπίζω να έχουμε περισσότερο χρόνο εκεί για να τα συζητήσουμε επιμέρους. Ο συνάδελφος Μπακ ε, ανέφερε ότι ε, και που αναφερόμαστε και στη στρατηγική καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής με σαφήνεια και ακρίβεια. Ως πολίτης εγώ, αλλά και μέλος της ε, ΕΟΚΕ, αλλά κυρίως ως πολίτης και Βέλγος, πολλό δε μάλλον, με όλες αυτές τις ε, διαδηλώσεις που βλέπουμε υπέρ του κλίματος τις τελευταίες εβδομάδες στο Βέλγιο, που διεξάγονται με αξιοσημείωτη ηρεμία θα έλεγα ότι θα πρέπει να δοθεί μια συνέχεια στο κείμενο αυτό. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το συζητήσουμε. Η Ολομέλεια του Φεβρουαρίου ήταν μεν καλή, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα και περισσότερο. Και το δεόδες, γιατί δεν πειράζει να ε, είμαστε και ονειροπόλοι, να καλέσουμε τους νέους αυτούς, όχι να τους ε, κλητεύσουμε, να τους καλέσουμε πραγματικά για να τους δείξουμε τι συνέχεια δώσαμε στην προσπάθειά τους με συγκεκριμένα στοιχεία και θα τελειώσω με την παρατήρηση του ΣΥΜΟΣ. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών είναι κάτι το οποίο διατρέχει όλο το κείμενο. Ο υπαριθμόν ένα στόχος είναι η καταπολέμηση της ένδυας. Ειλικρινά, δεν μπορείτε να μας καταλογίζετε ότι δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Αυτό διαφαίνεται από πολλές παραγράφους. Θα σας αναφέρω το κεφάλαιο για την κοινωνική Ευρώπη και τη δίκαιη φορολόγηση. Δύο παραδείγματα μόνο, αλλά και αλλού αναφέρονται αυτά. Δεν προλάβαμε. Ε, ίσως να πούμε σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά αν κανείς διαβάσει προσεκτικά το κείμενο θα καταλάβει ότι και οι τρεις συνεισηγητές ε, θέλαμε να εντάξουμε αυτή την της φτώχειας. Τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Για τη συζήτηση. Καταληκτικά. Να κάνω και εγώ ένα κλείσιμο. Είναι σημαντικό το ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε πλήρως τους νέους στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθε. Ελπίζω να μην ε, παραμείνει κενός λόγος. Πρέπει να είναι πρωταγωνιστές, όχι απλώς να τους κάνουμε μαθήματα. Ακούσαμε τους νέους, οι οποίοι εκφράστηκαν σαφέστατα, είτε ήταν η Μαγδαλένα και η Γκρέτα Τούμπερ. Η γνωμοδότηση αυτή επιμένει επίσης δεν το είπαμε ήδη, στο ρόλο του πολιτισμού που είναι ζωτικός και αναφέρει ότι για την επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι οριζόντιος στόχος η βιωσιμότητα και μην ξεχνάμε για να προχωρήσει αυτά που λέει η γνωμοδότησή μας για να υπάρξει αυτή η προοπτική δημοσιότητας το βασικό είναι τι θα γίνει με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι υποσυζήτηση και το λέμε στην γνωμοδότησή μας. Το πλαίσιο αυτό όπως υποβλήθηκε δεν επαρκεί. Δεν είναι στο επίπεδο των φιλοδοξιών μας για μια πραγματικά βιώσιμη Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι πολύ θαραλέα η γνώμη μας. Πρέπει όμως ε, να είμαστε έτοιμοι για την επερχόμενη μάχη. Δεν αρκούν τα κεκτημένα το 40% για παράδειγμα. Έχουμε τους ε, συμμάχους μας, την Επιτροπή των Περιφερειών και το Κοινοβούλιο, το οποίο όμως ε, θα αλλάξει. Θα αλλάξει και θα εκλεγεί ε, μια νέα θητεία. Έχω ήδη συζητήσει με τον πρόεδρο Λάμπερτ της ε, Επιτροπής των Περιφερειών, ούτω ώστε να έχουμε συγκλίνουσες στρατηγικέ για να ξαναξεκινήσουμε τη μάχη το Σεπτέμβριο που θα ξαναξεκινήσει η διαπραγμάτευση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και καταλήγοντας. Ζατώθηκα. Και η Επιτροπή μας πρέπει να αποφύγει τα πολλά λόγια, να περάσει στην πράξη. Πρέπει να τολμήσουμε την καινοτομία, να ρισκάρουμε. Δεν θα ήθελα τα λόγια αυτά να τα απευθύνουμε ως ε, προτροπές μόνο προς τους άλλους. Και εμείς επίσης πρέπει να έχουμε το θάρρος να καινοτομούμε, να ρισκάρουμε, να αλλάζουμε. Αλλιώς τα αιτήματά μας ε, προσαρμογής μέσω καινοτομιών ε, στις αλλαγές των καταστάσεων δεν θα προχωρήσουν. Πρέπει να παίξουμε το θεσμικό μας ρόλο που αναφέρθηκε στις συνθήκες να δώσουμε φωνή στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να έχουμε το θάρρος, να είμαστε πιο καινοτόμοι, να έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική στον τρόπο προσπάθειας κινητοποίησης του κοινωνικού διαλόγου, του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 της συνθήκης. Και τώρα να περάσουμε στην ανάλυση των τροπολογιών με βάση την τακτική διαδικασία. Τροπολογία 1.5. 1. Της κυρίας Τέλερ. Amendment number Τροπολογία 1. Στο σημείο 1.5. Τροποποιηθέν κείμενο ε, της κυρίας Τέλερων. Το δέχεστε ή το απορρίπτετε. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε λέει ο εισηγητής. Είμαστε σε ένα βασικό σημείο της ε, τροπολογίας. Η θέση μας ήταν της γνωμοδότησης, συγγνώμη. Η θέση μας είναι ότι πρέπει να υπάρξουν ε, σαφείς ορισμοί για το μέλλον. Αν θέλουμε να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη ή βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, δεν χρειάζεται στις ομάδες εργασίας να συζητάμε τους ορισμούς. Γι' αυτό υπάρχει συνένεση για συγκεκριμένο ορισμό για την επιτροπή μας. Και η τροπολογία τέλευο δεν ε, διευκρινίζει την κατάσταση θα μας οδηγούσε σε ατέρμονες συζητήσει επί των ορισμών. Θέλουμε να μείνουμε στο κείμενο όπως είναι. Και ελπίζουμε να μας καταλαβαίνετε, αλλά δυστυχώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε αυτή την τροπολογία. Ε, I thank the report. Ευχαριστώ τον συγκριτή. αλλά διαδικαστικά. Πρέπει να μας πείτε αν δέχεστε ή όχι. Αν δέχεστε, αν δεν δέχεστε, πρώτα θα πάρει το λόγο ο συντάκτης της ε, ε, τροπολογίας και μετά θα πάρετε το λόγο εσείς. Τώρα το κάναμε αντίστροφα, δεν σωστή διαδικασία, αλλά από ό,τι κατάλαβα βεβαίω την απορρίπτεται. Ωραία, παρακαλώ κύριε να υποβάλλετε την τροπολογία σας. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, αναφέρομαι στα υλικά μονής χρήσης. Δεν νομίζω είναι σωστός ο ορισμός. Το έχω πει επανειλημμένα και δεν καταλαβαίνω. Ο τρόπος που αναφέρεται στο σημείο 4 είναι περίεργος. Εγώ ακολουθώ το πρότυπο. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι σωστό το κείμενο που έχω. Ωραία, όπως ήδη επεξηγήθηκε. Ο συγητή είναι κατά τη τροπολογίας. Άρα ψηφίζουμε τροπολογία 1. The vote is closed. Πέρασε η ψηφοφορία. 132 against, 11 abstention is refused. Amendment number two on the point 1.6, always from Televo. Στο σημείο 1.6, κυρία Τέλερβο. Το δέχεστε? Όχι, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Όχι. Κυρία Τέλερβο, παρουσιάστε την τροπολογία σας. Μα δεν καταλαβαίνω το κείμενό σας λέμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ισορροπία και τα λοιπά και την συμπερίληψη όλων την κοινωνική ένταξη με τους δείκτες αυτούς που αναφέρετε όμως ήδη το αναφέρετε δύο φορές ευχαριστώ πολύ οι συνεισηγητές συζητώντας το είπαμε ότι είμαστε στην αρχή του κειμένου με ορισμούς ιδιαίτερα σημαντικούς ήδη αναφερθήκαμε σε έναν άλλο ορισμό τώρα εδώ μιλάμε για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και έχουμε και μία υποσημείωση που αναφέρεται σε διάφορες εργασίες για τα θέματα αυτά θεωρούμε ότι το κείμενό μας είναι σαφέστερο από αυτού που προτείνει η Τέλεργο. Ευχαριστώ πολύ, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Υπέρ 64. 148 κατά. 13 αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Πάντα από την κυρία Ρουόναλα. Υπέρ κατά. Μια συμβαστική λύση. Η τροπολογία αφορά την τελευταία πρόταση. Θα θέλαμε να την αποδεχθούμε κατά μέρος, την πρότασή της δηλαδή. Αλλά να διατηρήσουμε τη βάση του δικού μας αρχικού κειμένου. Να σας διαβάσω λοιπόν τη συμβαστική τελευταία πρόταση. Μια σωστά λειτουργούσα οικονομική ελευθερία και οι κανόνες του ανταγωνισμού πηγαίνουν παράλληλα με, τη θεμελι... με τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, αλλά δεν θα πρέπει να τα ανταγωνίζουν, να τα υπονομεύουν. Συγγνώμη. Κυρία Τέλερβο, το δέχεστε αυτή τη συμβαστική λύση. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάτι που να είναι κατά του συμβασμού αυτό. Όχι, ωραία. Δεκτή. Τώρα έχουν τροπολογία 5 για το πρώτο πλαίσιο μετά το σημείο 1.14. Πάτε την κυρία Ρουόναλα. Τη δέχεστε ή όχι. Όχι. Πρέπει να το δούμε σε σχέση και με το επόμενο. Αλλά είμαστε κατά αυτής της τροπολογίας. Είστε κατά. Οπότε κυρία Ρουόναλα, παρακαλώ, παρουσιάστε την τροπολογία σας. στην εντολογική έκθεση δεν καταλαβαίνουμε πώς η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών στις αγορές μπορούν να μετρηθούν. Όλα εξαρτώνται από την άποψη του καταναλωτή, ο οποίος αλλάζει συνεχώς. Ευχαριστώ πολύ. Εισηγητές. Όπως είπα, πρέπει να το δούμε σε σχέση και με την επόμενη τροπολογία του Στέφαν Μπάξιν όπου έχουμε ένα συμβιβασμό που αποδέχεται σχεδόν τα πάντα. Ε, μόνο ένα σημείο δεν δεχόμαστε. Αυτό δεν πάει εδώ. Αλλά υπάρχει και ένα σοβαρό λόγο για μα. Αν ε, διαγράψουμε την τελευταία πρόταση, θα ξανακάνουμε τη συζήτηση που έχουμε κάνει επανειλημμένα, ιδιαίτερα για τα συστήματα τροφίμων, όπου υπάρχει καταστροφικό ανταγωνισμό με βάση την τιμή και πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε πιο ποιοτικά κριτήρια. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την τροπολογία. Και στην επόμενη τροπολογία όμως έχουμε μια πρόταση όπου ακριβώς θα συμφωνήσουμε με την τροπολογία του Στέφαν Βάξ. Οπότε κυρία Τέλερβο, οι συγγητές λένε ότι θα ε, συμπεριλάβουν τμήμα της δικής σας τροπολογίας στη συμβαστική διατύπωση για την τροπολογία Στέφαν Βάξ. Ε, επιμένετε ή αποσύρετε την τροπολογία σας. Επιμένω. Είναι πραγματικά σημαντικό για μένα. Και δεν έχει να κάνει με το επόμενο κείμενο. Ωραία, ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. υπέρ, 148 κατά και 9 απόχέ. 149 κατά μάλιστα. 9 απόχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Επί του σημείου 1.14. Στέφαν Μπακ. Υπάρχει μια συμβαστική διατύπωση. τροπολογία αυτή ε, είναι κάτι που επιχειρήσαμε να το συνδυάσουμε και με άλλα ε, κείμενα. Αλλά δεν ήταν δυνατό, γι' αυτό το ε, διατηρήσαμε χωριστό. Κρατάμε το αρχικό κείμενο και προσθέτουμε αυτό που προτείνει ο Στέφαν στο τέλος της παραγράφου. όπου βάζουμε τη λέξη βιωσιμότητα, εκεί θα βάλουμε ή αηφορία και βάζουμε κόμμα, στα πλαίσια μιας πλήρους ανεπτυγμένης και αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς. Έτσι δεχόμεθα εν μέρη την πρόταση και βελτιώνουμε την πρότασή του προσθέτοντας τη λέξη αποτελεσματικά λειτουργημένες που να είναι πλήρως αναπτυγμένη και ε, σωστά λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Η αποτελεσματική. Στέφαν, δέχεσαι. Δέχεσαι, ωραία. Είναι κανείς κατά. Ωραία. Όχι. Ωραία. Δεκτό. Τροπολογία 6. Επί του 1.14. Η πέμπτη κουκίδα η κυρία κυρία Χαράκα Ρουόναλα. Παρακαλώ. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Κυρία Ρουόναλα, θέλετε να παρουσιάσετε την τροπολογία σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το θέμα που συζητήσαμε και προηγουμένως, βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι θέμα που αφορά και αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Η απάντησή μου είναι ότι μίλησα με τον συντάκτη και εδώ θέλαμε να επικεντρωθούμε στις επιχειρήσεις. Θέλουμε οι επιχειρήσεις να γίνουν φιλοδοξότερες και να αναλάβουν δράση και μάλιστα στο διεθνές προσκήνιο. Αυτό είναι το μήνυμά μας, να επικεντρωθούμε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Άραγε, θεωρώ ότι είναι άστοχη η τροπολογία, διότι αναφέρει την κοινωνία των πολιτών, τους καταναλωτές και τους εργαζομένους. Δεν λέγαμε αυτό. The vote is closed. 56 προς 4, 139 κατά και 9 αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Δεκτή. Υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση. 17 στο δεύτερο κουτάκι μετά το 2-2, δεύτερο πλαίσιο μετά το σημείο 2-2, πέμπτη περίπτωση. Αυτή είναι πρόταση της ομάδας 2, αλλά θα την υποβάλω εγώ εκ μέρους τους, γιατί τη συμφωνήσαμε και στην ομάδα μας. Η τροπολογία αυτή αφορά το κεφάλαιο 2 για τους πολίτες. Έχει να κάνει με το δεύτερο σημείο, με τη δεύτερη κουκίδα. Προτείνουμε να δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα στην Επιτροπή μας που να συνεννοηθεί με μια ανάλογη ομάδα της Επιτροπής των Περιφερειών και να έχει ένα μόνιμο συμβουλευτικό χαρακτήρα για διαρθρωμένες διαβουλεύσεις και διάλογο με τους πολίτες. Και αυτό για να υποστηρίξουμε την δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης και να έχουμε και ρεαλιστικές ε, αντιδράσεις από τους πολίτες για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε την πρόταση αυτή και να αφήσουμε τον συμβουλευτικό μηχανισμό κατά μέρο, γιατί τελικά δεν είχαμε χρόνο να το συζητήσουμε διεξοδικά. Και σε δεύτερη φάση θέλαμε να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας ε, ατόφια ως Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Θέλουμε να ε, μας ε, αντιμετωπίζουν ως μοναδική πλατφόρμα αυτό είναι ο στόχο μα, να εκπροσωπούμε την κοινωνία των πολιτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το ρόλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να παραμείνει η πρώτη πρόταση, ωστόσο κάναμε κάποια αλλαγή και θα το διαβάσω αγγλικά. Η ΕΟΚΕ θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και θα συνεχίσει να είναι ένας ενεργός πρωταγωνιστής στην χάραξη πολιτικής. Τελεία. Anyone is Είναι κανείς κατά σε αυτό που προτείνει η εισηγήτρια. Κρίστοφ Πάτερ. Δεν είμαι ακριβώ κατά, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε θεσμικό όργανο. Δεν είμαστε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Νομικός μιλώντας, είμαστε συμβουλευτικό όργανο, αλλά όχι θεσμικό. Δεν είμαι βέβαιο. Για να το ελέγξουμε καλύτερα πριν το γράψουμε. From the formal point of view, you are... Από τυπική άποψη έχετε απόλυτο δίκιο το επιβεβαιώνουν οι συναδελφοί μου, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πρόταση τώρα. Ή θα παραμείνουμε στην αρχική ή θα περάσουμε στη, σε αυτή. Εάν παραμείνουμε στην αρχική, Μπορείτε να το ξαναδιαβάσετε γιατί δεν ήταν σαφές. Ναι, θα παραμείνει η πρώτη πρόταση με μια μικρή αλλαγή στο τέλος. Η ΕΟΚΕ ως θεσμικός εκπρόσωπος της Οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσει να αποτελεί ενεργό πρωταγωνιστή σε αυτή τη διαδικασία, τη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Τελεία. No one is against. Δεν έκανε κατά. Ωραία, ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Δεκτή. Ωραία. Είναι κανείς κατά. 9. Τροπολογία της κυρίας Σβέγγ. Έχουμε βρει ε, συμβαστική λύση. Διαβάστε την παρακαλώ. Το συζητήσαμε διαμακρών το θέμα αυτής της τροπολογίας και προτείνουμε την εξής διατύπωση που θα αντικαθιστά το αρχικό. Στο πλαίσιο της, των αυξανόμενων ανησυχιών για την ε, αποκλίνουσα πρόοδο των κρατών μελών θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για έναν κατώτατο μισθό και ένα κατώτατο εισόδημα ως μέρος ενός κοινού, μιας κοινής διαδικασίας σύγκλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό στοιχείο κοινωνικής προστασίας και αυτό θα βοηθούσε να πετύχουμε αξιοπρεπή βιωτικά, ε, ένα αξιοπρεπέ ε, πρότυπο βιωτικού επίπεδου σε όλε χώρες και θα υποστηρίζαμε την ανάπτυξη ενισχύοντας την σύγκληση του και να ε, αποφύγουμε τις αποκλήσεις εντός της Ένωσης. Είναι κανείς κατά της συμβαστικής? Όχι, οπότε γίνεται δεκτή. Τροπολογία 10. Στέφαν Μπακ, τρίτο πλαίσιο. Δέχεστε ή αρνείστε. Δεκτή. Είναι κανείς κατά. Ευχαριστώ. Τροπολογία 11. Πάλι του Στέφαν Μπακ. Δεκτή. Έχουμε συμβαστική. Λοιπόν, ο Στέφαν θέλει να διαγράψουμε το 100% και να γίνει υψηλότερο επίπεδο την πρόταση. Εμείς θα πούμε το, δυνατότερο υψηλό, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Highest possible. Δεκτή συμβαστική. Είναι κανείς κατά. Όχι. Δεκτή 12. Τροπολογία 12. Δεκτή απορρίπτεται. Και εδώ συμβαστική η λύση. Πέστα. Η δική μας πρόταση ήταν να μην ε, πούμε ότι θα ιδιωτικοποιηθούν σταδιακά οι κρατικέ υπηρεσίε και να υπάρχει πρόσβαση μόνο ορισμένου. Γι' αυτό προτείναμε την εξή συμβαστική. Διαβάζω. Οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες, τα βασικά δημόσια αγαθά όπω το καθαρό πόσιμο νερό, ο καθαρός αέρας και το παρθένο έδαφο. πρέπει να είναι δωρεάν. Και προσθέτουμε και προσιτά σε όλους με χαμηλό κόστος. Προσθέσαμε το N affordable cost με χαμηλό κόστος. Γίνεται δεκτή η συμβαστική. Ωραία, ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Ωραία, πέρασε. Τροπολογία 13. Και εδώ έχουμε συμβαστική. Πείτε την. Η πρόταση του Στέφαν είναι να υλοποιηθούμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές συμπεριλαμβανομένων. Εμείς αυτό θέλουμε να διαγραφεί, να παραμένει το driving. Άρα στο τέλος της πρώτης φράσης να λέει το εξής. Όταν ορίζουμε και υλοποιούμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές διότι θέλαμε να παραμείνει αυτή η πρώτη θέση Δεν έχει πιστεί πολύ ο συγκριτή τη τροπολογία, αλλά τη δέχεται. Είναι κανεί κατά. Δεκτή, περνάει. Τροπολογία 14. Παρακαλώ. Θα διαβάσω απευθεία όλο το κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές της πολιτικές είναι συνεκτικές και ευθυγραμμίζονται με τους ΣΒΑ, τους κοινωνικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι, η αρχή της αναλογικότητας και της βιωσιμότητας λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Συμπληρώσαμε τον όρο αρχές, για να είναι σαφές γιατί μιλάμε. Είναι κανείς κατά. Τροπολογία 14. 15. Μπρέντα Κίνγκ πάλι. Δεκτή ή απορρίπτεται. Πάλι συμβαστική. Έχει να κάνει με το 15. Στο 10, στο, με το 16 το 15 προτείνουμε να διαγραφεί η λειτουργία σε δύο κατευθύνσεις κτλ και η πρότασή μας θα καλυφθεί από το 16 ούτως ή άλλως. Το 15 λοιπόν η συμβαστική είναι να διαγράψουμε την αναφορά ε, αυτό που προτείνει να προσθέσουμε η Μπρέντα. Δεν κατάλαβα τη συμβαστική. Ναι, να τα ξαναπώ. Η τροπολογία 15 και η 16. Είναι δύο διαφορετικές τροπολογίες. Η δική μας συμβαστική είναι να τις ενώσουμε. Σου προτείνουμε, Μπρέντα, να διαγράψουμε αυτό που είπες στη 15 και δέξου το σε παρακαλώ γιατί θα το πάμε στο 16 εισηγητά, σου προτείνω να διαβάσει την ε, τροπολογία. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα έτσι όπω τα λες. Ωραία, λοιπόν, πάω στη 16. Επαναλαμβάνω αυτό που λέει η Μπρέντα. Στο 15 διαβάζω. Η ένταξη είναι... Και εδώ υπάρχει μια μικρή αλλαγή. Αυτή είναι η συμβαστική. Η ένταξη είναι μια διαδικασία αμφίδρομη και οι δύο πλευρές έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και πρέπει να ε, το βάλεις αυτό στην πρότασή σου και μετά συνεχίζουμε. Οι ευθύνε θα πρέπει να είναι κοινέ και η πρότασή σου συνεχίζεται κανονικά. Μετά δεύτερη φράση, για να διευκολυνθεί αυτή η αμφίδρομη ένταξη, διαγράφουμε το ένταξη και λέμε για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία αντί για αμφίδρομη ένταξη πάλι. Εντάξει. Και μετά όλο το υπόλοιπο δεκτό. Στο 16. Το τέλος δηλαδή και διαχόμαστε να διαγραφεί το για τους ίδιους μετανάστες αλλά και τα λοιπά. Για λόγους σαφήνειας, διότι είναι σαφές. Δεν δέχεστε το 15 γιατί θα συμπεριληφθεί έτσι καλώς το 16 που αναθεωρήθηκε. Μπορείτε να διαβάσετε το τελικό κείμενο του 16 να το καταλάβουν όλοι. Η ένταξη είναι μια διαδικασία αμφίδρομη. Και οι δύο πλευρές έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Άρα, η ευθύνη πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και των μεταναστών. Δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε βιώσιμο να έχουμε την αξίωση οι νεοαφιχθέντες να ενταχθούν χωρίς βοήθεια και απέναντι σε αξιόλογους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς φραγμούς. Για τη διευκόλυνση της αμφίδρομης, της διαδικασίας μάλλον αυτής, οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους φόβους, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες διαφορετικών τμήματων του πληθυσμού της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται οι εχθρικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξενοφοβικές ρητορίες. Προ τούτο, οι σχετικές πολιτικέ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σαφέ, συνεπές και αιτιολογημένο σύνολο υποχρεώσεων, καθώς και μια συνεπή καταγγελία της αντιμεταναστευτικής ρητορία και συμπεριφοράς. Άρα ε, φεύγει 15, αποσύρεται, 16 να θεωρήθηκε όπως είπαμε. Μπρέντα Κίνγκ, είστε υπέρ. Υπάρχει κανείς που να έχει αντίρρηση. Σαφή για όλους. Ωραία. Γίνεται δεκτό. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία.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 Λοιπόν, προχωρούμε. Στο επόμενο θέμα, ΣΟΚ 605. Εισηγητή Κριστιαμό. Ανθεκτική δημοκρατία μέσω μια ισχυρή και πολύμορφη κοινωνία των πολιτών. Thank you very much, dear President. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η παρούσα γνωμοδότηση είναι ιδίας πρωτοβουλίας και αποτελεί καρπό κοινής ε, εργασία στην ομάδα με, μελέτης και στην πολύτιμη συνεισφορά επίσης οφείλεται πολλών μελών που ε, ενδιαφέρθηκαν για το θέμα αυτό και τη γνωμοδότηση. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που βοηθήσατε για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και να μπορούμε σήμερα να σας το παρουσιάσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον Χωσέ Αντώνιο Μορένο Ντίας, ε, Πρόεδρο της Αρμόδιας Ομάδας κάτω Δικαίου και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που προφανώς ε, συνδέεται άρρηκτα με το θέμα αυτό. Δημοκρατία και κοινωνία των πολιτών. Ουσιαστικά λοιπόν ε, προσπαθούμε λοιπόν να συγκεντρώσουμε όλα αυτά που λέμε και ζητούμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι καινούριο δυστυχώς αυτό που αναλύουμε τώρα. Οι εξελίξεις συνεχίζονται σε καθημερινή βάση και βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι είναι σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτή. Σε ό,τι αφορά και το χώρο έκφρασης των πολιτών, τη δημοκρατία και την ακαιρεότητά της. Έχουμε πολλές νομοδοτήσεις για τη δικαιοσύνη, για τα δικαιώματα, για τις αξίες ε, στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ένα εξάμεινο για τη δημοκρατία. Όλα αυτά τα έχουμε προσθέσει, καθώς επίσης και νέες συστάσεις και νέα δεδομένα και ευρήματα. Υπάρχουν και κάποιοι ορισμοί που τους θεωρούμε πολύ σημαντικούς. Τι εννοούμε όταν ομιλούμε για δημοκρατία. Μιλούμε εδώ για τη φιλελεύθερη δημοκρατία, για την πολυφωνική κοινωνία των πολιτών και πώς και αυτά τα δύο συνδέονται άρρηκτα. Ο πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη που διακόπτω τον εισηγητή. Παρακαλούνται θερμά όσοι θέλουν να κάνουν ιδιωτικές συζητήσεις να αποχωρήσουν από την αίθουσα και όσοι θέλουν να ακούσουν τον ομιλητή να τον ακούσουν με την ισχύ τους. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι μια διαδικασία συνεχής. Θα ακολουθήσουν και άλλες νομοδοτήσεις. Μία συνάδελφος προσεχώς θα αρχίσει μια δική της νομοδότηση, πάλι ε, πρωτοβουλία. πρωτοβουλίας. Και φοβούμε ότι θα το βρούμε και θα το βρίσκουμε συχνά μπροστά μας αυτό το θέμα. Ελπίζω να βοηθήσει κάπως η γνωμοδότηση, γιατί έχει να κάνει και με την ταυτότητά μας και δεν αντιδρούμε σε κάποια νομοθετική διαδικασία τρέχουσα και επίκαιρη προσπαθούμε να ορίσουμε το ποιοι είμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Ελπίζω να μπορέσει αυτό να αποτελέσει τη βάση για τη συνεχιζόμενη εργασία και τη διαρκή συνεργασία ε, της Ομάδας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για μελλοντικές νομοδοτήσεις. Ας συνεργαστούμε για να υπερασπιστούμε ε, το χώρο έκφραση των πολιτών ε, και τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Κρίστιαν. Μακρύς ο κατάλογος των ομιλητών. Κλείνει τώρα. Πρώτη παρέμβαση, Λεκ Πιλάσκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πολωνικά. Το έχω ξαναπεί στη συζήτηση που έγινε ε, στο αρμόδιο τμήμα ε, των κοινωνικών υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ για την γνωμοδότηση αυτή και τον εισηγητή και όλη την ομάδα. Ε, γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή αυτή η γνωμοδότηση, όπως και η προηγούμενη, πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ μονοσήμαντη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εδώ έναν ορισμό βάσει του οποίου να ξέρουμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται και τι είναι παραδεκτό και τι είναι απαράδεκτο. Επίσης, ε, περιγράφουμε και ορίζουμε πολύ καλά τα φαινόμενα, κυρίως τα αρνητικά φαινόμενα που σήμερα αντιμετωπίζουμε στην Πολωνία. Και είναι καλές και οι συστάσεις, διότι εμείς δεν μπορούμε να ε, αρκούμαστε στο να κάνουμε διαπιστώσεις και μια αποτύπωση της κατάστασης, τα θετικά και τα αρνητικά, θα πρέπει να πάρουμε και θέση. Έτσι ώστε οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα που συνδέονται με την ε, δημοκρατική πολιτική τάξη να γίνονται σεβαστά στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ για το κείμενο αυτό. Η Καρολίνα Ντρέσνες Μάλετς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνήσω και εγώ με τον προλαλήσαντα. Πραγματικά είναι πολύ θετικό που μας απασχολεί αυτό το θέμα, το τόσο σημαντικό. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη και θα πρέπει να δούμε ποιο δρόμο θα επιλέξουμε. Ευχαριστώ τον εισηγητή Κριστιαν Μος αλλά και όλη την ομάδα που ε, ανέλησε την κατάσταση. Είχα και εγώ την ευκαιρία να βάλω το λιθαράκι μου. Ε, δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα ήδη ακούσαμε, απλώς να πω και πάλι πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέει και ε, ο ίδιος ο τίτλος «Ανθεκτική δημοκρατία μέσω μιας ισχυρής και πολύμορφης κοινωνίας των πολιτών». Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε να διαβιβάσουμε και να έχουμε πάντα υπόψη μας πέρα από τους διάφορους κοινωνικούς κανόνες που εγκρίνουμε, ο καθένας από εμά είναι πολίτης. Και όταν επιστρέφουμε στη χώρα μας και προβληματιζόμαστε για τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζούμε, δεν είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν βασιστούμε στις αρχές και τις αξίες μας. Μια Ευρώπη ε, που να σέβεται όλους τους πολίτες με πολυμορφία αλλά όπου να μην αποκλείεται κανείς. Επίσης, η ελευθερία της κοινωνίας των πολιτών είναι θεμελιώδης, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να περιστέλλεται αυτή. Γιατί αυτό ανοίγει το δρόμο στην ενίσχυση κάποιων αυταρχικών τάσεων που παρατηρούμε σήμερα στην Ευρώπη ο περιορισμός ας πούμε, της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων, ο περιορισμός της ε, δυνατότητας ε, να λειτουργούν απρόσκοπτα τα μέσα ενημέρωσης οδηγεί και σε άλλους περιορισμούς. Ε, το περιθώριο χειρισμών και λιγμών των ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών, γιατί είναι οι πρώτοι που αντιδρούν σε όλες τις αδικίες και οθούν και τις ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις στη συνέχεια να αντιδράσουν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κοινωνία, γιατί αυτό είναι ένα εχέγγυο για μια ισχυρή δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Τζούντι Μακνάιτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ ε, τον Κρίστιαν. Εξαιρετική η γνωμοδότηση. Εγώ δεν είμαι μέλος τυπικά της ομάδας μελέτης, αλλά πήγα και στις δύο συνεδριάσεις και σε, ε, συνεδρίες και σε μια εξαιρετική ακρόαση που διοργανώθηκε. Είναι πραγματικά υπόδειγμα ομάδας ε, μελέτης. Και ο Κρίστιαν άκουγε όλους τους συναδέλφους και πραγματικά βοηθήσαμε όλοι να φτάσουμε σε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί θεωρώ ε, άλλη μια έκφραση και έκφανση του λαϊκισμού την ψηφοφορία και το δημοψήφισμα για το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία. Και κάτι που λέει και το έγγραφο στην παράγραφο 622 προς το τέλος είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα δούμε απαγκιστρωμένα από τα υποκείμενα κοινωνικά προβλήματα. Υπάρχει η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και μια ε, καλώς λειτουργούσα αγορά εργασίας, δίκαιη φορολόγηση, αποτελεσματικές κοινοφελείς υπηρεσίες κτλ. Και ε, ε, εξού και το Brexit, γιατί είχαν ατονίσει ή είχαν παραγωνιστεί ε, στις περιφέρειες που ε, ψήφισαν υπέρ της εξω. ελπίζω λοιπόν να αποτελέσει μια πολύ καλή βάση αυτό το κείμενο για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Μπέρν Σλούτερ. Και εγώ συμφωνώ με τους επένους που εκφράστηκαν. Αυτή η γνωμοδότηση ίσως να την χρειαζόμασταν και νωρίτερα. Αλλά είναι καλό που την έχουμε έστω και τώρα να αναφερθώ σε δύο σημεία επί των οποίων θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε στην Επιτροπή μας. Το πρώτο είναι η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων. Ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μήπως ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα εκτενέστερο κείμενο για το σημείο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση κατά κάθε παραπληροφόρηση και κακής χρήση των μέσων και άρα και των πολιτών από τους ε, ολιγάρχες, τους δισεκατομμυριούχους, είτε τις κυβερνήσει, είτε τα κόμματα Θυμάμαι ακόμη ότι υπήρχε η δημόσια ραδιοτηλεόραση και υπάρχει. Δεν είναι τέλεια, αλλά είναι μια μορφή όπου η κοινωνία των πολιτών συναποφασίζει για το περιεχόμενο και τα προγράμματα. Υπάρχουν ήδη κράτη-μέλη όπου δεν είναι πια δεδομένη η δημοκρατική διαμόρφωση άποψης της κοινή γνώμης. Τα κριτήρια της Κοπενχάγης που είναι κριτήρια ένταξης για μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πληρούνται πλέον. Και τίθεται λοιπόν το ενδιαφέρον ερώτημα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Δεύτερον, η επιτήρηση της, ε, του διαλόγου για την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Ο δικαστής Διφάμπιο ε, είπε ότι πρέπει να μην γίνεται σε πολιτικό επίπεδο η συζήτηση, αλλά μεταξύ νομικών μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι... Όχι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω για αυτή την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ Γιώργο Σιμπίον. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ε, και εγώ να συγχαρώ τον Κρίστιαν. Πολύ καλή γνωμοδότηση. Νομίζω ότι υπογράμμισε πολλά σημαντικά θέματα. Χαίρομαι που έχει τόσο σημαντικά στοιχεία αυτό το κείμενο κάποια θέματα που νομίζω ότι θα προσέθεταν ε, αξία. Πρώτα απ' όλα, εφόσον πρόκειται να έχουμε ένα εξάμεινο για τη δημοκρατία, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κριτήρια για την ε, ποιότητα της δημοκρατίας. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια σωστή μεθοδολογία για να μετρήσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας. Χρειαζόμαστε ένα εργαλείο που να μας επιτρέπει να καταδικάζουμε και τις παραβιάσεις της δημοκρατίας. Υπάρχουν διάφορα κείμενα από διάφορους φορείς. Καλό θα ήταν ε, να ε, δούμε πώς μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε σε μία επόμενη γνωμοδότηση. Αναφέρονται πολλά και για τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών. Χαίρομαι πολύ που το αναφέρεις αυτό στη γνωμοδότησή σου. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε με το άρθρο 2 της συνθήκης. Συμφωνώ απόλυτα ότι οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Ένωσης που κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, συνάδει με τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης. Και κάτι που είναι καλό είναι επίσης ότι μπόρεσαν να συμβάλλουν τα τελευταία χρόνια ε, στην εργασία αυτή και Διάφορε οργανώσεις και μη κυβερνητικέ, αλλά και το όργανο για την ε, διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Θαυμάσια γνωμοδότηση γενικώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία η Μαρίτα Τεσίνγκερ. Όχι, ο Μαρίτα Τεσίνγκερ. Ναι. Πολύ καλή γνωμοδότηση. Θέλω να ενισχύσω ορισμένα τα οποία υπόθηκαν και μας δίνει και στοιχεία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες νομοδοτήσεις είναι σημαντικό για να υπάρχει δημοκρατία στην Ένωση και να διατηρηθεί τώρα και εν ώψη των ευρωεκλογών. Διάφοροι ευρωσκεπτικιστές βέβαια θα έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο και μόνο για να το υπονομεύσουν. Πρέπει λοιπόν να καταγγείλουμε το αρνητικό τους χαρακτήρα των παρεμβάσεών τους δηλαδή και να επανέλθω σε κάτι που είπε η Τζούλι Νάιτ μέσω του Brexit διαπιστώνουμε στον Ηνωμένο Βασίλειο τι παραπληροφόρηση αξιοποιήθηκε την οποία ε, την κατάπιε το εκλογικό σώμα. Ένα παράδειγμα. Ο Νάιτζελ Φαράτζ ο οποίος καθόταν μπροστά από μία ε, αφίσα που έδειχνε κάποια άτομα και καταδίκαζε την ε, μετανάστευση. Και τα άτομα αυτά στην εικόνα ήταν άτομα που έφευγαν από την Συρία. Και ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματο ε, τα κατάπια μάλιστα όλα αυτά τα ψέματα, της ανοησίε. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να μα προστατεύει από τέτοια φαινόμενα. Εφόσον θα έχουμε ευρωσκεπτικιστέ στο Κοινοβούλιο, πρέπει να του καταγγείλουμε. Από την αρχή. Ευχαριστώ, Κριστιαν. Δύο λεπτά. Ναι. Σας ευχαριστώ όλους. Όπως είπα, είναι συλλογικό έργο. Πολλοί από τους ε, ομιλητέ συνέβαλαν, τόσο άλλο είναι αργά, όντως. Έχουμε και ορισμένα σημεία που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για περαιτέρω γνωμοδοτήσεις. Το θέμα της ελευθερίας του τύπου βεβαίως, πολύ σημαντικό θέμα. Το δημοκρατικό εξάμεινο βεβαίως. Όπως θα είδατε είναι μια βελγογερμανική πρωτοβουλία. Από χθες έχει εγκριθεί επισήμως Οπότε νομίζω ότι έγκαιρα τοποθετούμεθα και εμείς. Με την γνωμοδότησή μας. Τέλος. Πρέπει παντού να ακουστεί η φωνή μας. Οπουδήποτε συμβαίνει κάτι, γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι από τους ε, εκδηλωμένους ε, εξτρεμιστές. Ξέρουμε ποιοι είναι και πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Αλλά εδώ που είμαστε σήμερα πρέπει να τονίσω ότι αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό είναι πολύ ψηλά ιστάμενοι εκπρόσωποι της Ένωσης να είναι πλευρό ε, δίπλα-δίπλα με φασίστες δικτάτορες και να έχουν καλές σχέσεις. Και αυτό με ανησυχεί εμένα προσωπικά. Και είναι ε, πράγματα που συμβαίνουν όλο και συχνότερα σε όλες μας τις χώρες. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να είμαστε καρτερικοί και ανθεκτικοί για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τροπολογίες. Έχουμε δύο τροπολογίες. Η πρώτη για το σημειο 616. Και η άλλη συνδέεται. Είναι δεκτή, τη δεχόμαστε όλοι. Υπάρχει κανείς κατά. Ωραία. Η δεύτερη είναι στα πορίσματα. Σχετίζεται με την πρώτη. Και η δεύτερη είναι δεκτή, έτσι δεν είναι. Υπάρχει κανείς κατά. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Και να ψηφίσουμε τώρα. Άρχεται. You vote against, no? Ο Κρίστιαν Μόλ θα καταψηφίσει λοιπόν την γνωμοδότησή του. Έτσι για να φανεί πόσο δημοκρατικοί είμαστε. Ε, Πέρας. 146 υπέρ, 5 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Now we'll go to examine the... SOC. Και τώρα, SOC 554. ενημερωτική έκθεση. Για ένα σημαντικό θέμα. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να ψηφίσουν στις ε, ευρωεκλογέ. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Είναι μόνο μια γενική συζήτηση. Και μετά ψηφοφορία. Για να μπορέσει το Προεδρείο να μεταβιβάσει την έκθεση προς τα άλλα θεσμικά όργανα. Και το λόγο στον Κρίστοφ 5 λεπτά. Good οι ευρωεκλογέ είναι πρώτων πυλών. Η προεκλογική εκστρατεία έχει ξεκινήσει. Πολλοί κόσμοι συζητάει τι πρέπει να κάνει για να αυξηθεί η συμμετοχή στις, και η προσέλευση στις ερχόμενες εκλογέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τώρα να φροντίσει να υπάρξουν περισσότεροι ψηφοφόροι. Και εμείς ως ΟΚΕ okay, ε, συντάσσουμε τις δυνάμεις μας με τους υπόλοιπους ε, ε, Πολλοί έχουν προχωρήσει στην ε, έκφραση συνθημάτων και σλόγγαν. Όμω πρέπει να δούμε πόσο πολιτικοί θύνοντε και τα μέσα μαζική ενημέρωση θα κινητοποιήσουν του πολίτε για να ψηφίσουν. Είναι ένα πρόβλημα. Ιδίω και πρέπει να πω δυστυχώ ω συνήθω κανεί δεν ασχολείται με τα εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που είναι αμαία. Αυτού που έχουν δηλαδή ειδικέ ανάγκε και αναπηρίε. Θέλουν, αλλά δεν μπορούν να ψηφίσουν. Είναι σημαντικά τα πραγματικά τους δικαιώματα και η άσκησή τους. Θέλουν να ψηφίσουν στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου. Γι' αυτό η ομάδα μας στις αρχές Μαρτίου ενέκρινε ε, αυτό το πρόγραμμα μια διαπαθή για την Ευρώπη, μια πραγματικότητα που είναι μακριά από τις δικές μας ε, καθημερινές ενασχολήσεις. Περίπου 800.000 Ευρωπαίοι πολίτες από 16 κράτη-μέλη δεν μπορούν να πούν αυτή τη φορά ψηφίζω θα πούν πάλι ε, δεν μπόρεσα να ψηφίσω. Επειδή από την εθνική τους νομοθεσία στερούνται το δικαίωμα ψήφου λόγω της αναπηρίας τους. Εκατομμύρια λέει αντί να πούν και αυτή τη φορά ψήφισα, το μόνο που θα μπορούν να πούνε είναι και αυτή τη φορά δεν μπορούσα να ψηφίσω επειδή υπήρχε τεχνικό ή διοργανωτικό πρόβλημα ε, στη χώρα μου. Σε κάθε μια από τις 27 ευρωπαϊκές ε, χώρες Υπάρχουν νόμοι ή διευθετήσεις ε, οργανωτικού τύπου που αποκλείουν ορισμένους ψηφοφόρους με αναπηρίες από τη συμμετοχή τους στις εκλογές. Σε οκτώ κράτη-μέλη, οποιοδήποτε δεν μπορεί να φτάσει σε εκλογικό κέντρο, σε κάλπη, δεν θα ψηφίσει, διότι δεν υπάρχουν εναλλακτικέ μορφές ε, να ρίξει κανείς την ψήφο του. Σε 12 χώρες η εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει να αλλάξει το εκλογικό κέντρο στο οποίο έχει εγγραφεί κανείς ανάλογα με το ε, τόπο κατοικίας του σε άλλο που μπορεί να είναι πιο βολικό για τον ψηφοφόρο με αναπηρία. Η τεράστια πλειοψηφία των εκλογικών κέντρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προσαρμοσμένα στι ανάγκε ε, των ανθρώπων με διαφορετικέ αναπηρίε και οι δημόσιε αρχέ δεν κατανοούν το πρόβλημα. Πολύ συχνά ορίζουν τα εκλογικά κέντρα ω προσβάσιμα μόνο εάν μπορεί κάποιο με αναπηρικό καροτσάκι να μπει ω εκεί. Ενώ δεν λαμβάνει υπόψη τι ανάγκε των ανθρώπων με άλλου είδου αναπηρίε. Σε 18 κράτη-μέλη οι τυφλοί ψηφοφόροι δεν έχουν κανένα τρόπο να ψηφίσουν ανεξάρτητα. Σε 7 κράτη-μέλη οι ψηφοφόροι πρέπει να σημειώσουν στο ψηφοδέλτιο τον αριθμό εγγραφής τους, τον αριθμό του υποψηφίου επιλογής τους, το όνομα του κόμματος για το οποίο ψηφίζουν. Αυτή η διαδικασία πραγματικά είναι επαχθής. Σε περίπου ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών οι ψηφοφόροι ε, που ζουν σε ιδρύματα με 24 ώρη φροντίδα ή βρίσκονται σε νοσοκομεία δεν έχουν κανένα τρόπο να ψηφίσουν. Σε κάποια κράτη-μέλη κάποιος με αναπηρία ε, δεν έχει καν το δικαίωμα να δεχτεί υποβοήθηση για να φτάσει να ψηφίσει. Εάν οι καλύτερε πρακτικέ όλων των χωρών εφαρμόζονταν, θα υπήρχε ένα ιδανικό σύστημα όπου κάθε Ευρωπαίο πολίτη όχι απλώ θα είχε την πλήρη δυνατότητα να ψηφίσει, αλλά θα μπορούσε και να επιλέξει ο ίδιο ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να ψηφίσει. Σκοπός της έκθεσης αυτής που περιέχει τουλάχιστον 200 θετικά παραδείγματα προς παραδειγματισμό από τα κράτη-μέλη είναι να προσφέρει ενημέρωση σε όλου του πολιτικού ηθήνοντε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικό επίπεδο για το πώ να προσαρμόζουν την νομοθεσία του στι ανάγκε ενό μεγάλου αριθμού Ευρωπαίων πολιτών. Οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, ιδίω αυτέ που επικεντρώνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, ή τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίε, θα έχουν τουλάχιστον στα χέρια τους ένα οδηγό ε, με οδηγίες χρήσης που θα βοηθήσει να ε, υπερασπιστούν τα δικαιώματα ψήφου όλων των πολιτών σε εθνικό επίπεδο. Όμω δεν μπορούμε να του εγκαταλείψουμε μόνο του σε αυτόν τον αγώνα. Εμεί ω ΕΟΚΕ οφείλουμε να του βοηθήσουμε. Πρέπει σήμερα να λάβουμε την απόφαση να διανεμηθεί η έκθεση αυτή σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη έκθεση θα βοηθήσει να θεμελιώσουμε κανόνες που θα διασφαλίσουν το 2024 στις επόμενες εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο κανένας Ευρωπαίος πολίτης, αλλά ούτε ένας δεν θα αποκλειστεί από το δικαίωμά του στην ψήφο. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να αναγνωριστεί όχι μόνο ως ένα στοιχείο των ένομων δικαιωμάτων, αλλά πρωτίστως και καταρχάς ως πρώτο ε, στοιχείο και σημαντικό στοιχείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κλείνει ο κατάλογος. Κρίστοφ Μπάλλον πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ Λούκα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξίστοφ, Σα ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή. Πραγματικά αφορά μια πάρα πολύ ευάλωτη ομάδα στην Ευρώπη και τα προβλήματα και οι φραγμοί είναι πάρα πολύ διαφορετικά και τα εμπόδια. Και δεν πρόκειται μόνο για κάποιες χώρες, όπως η δική μου Πολωνία, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και πολλές άλλες, στη Δυτική Ευρώπη. Για να μην μακρηγορώ, πιστεύω επίσης ότι η έκθεση αυτή παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία την Επιτροπή μας και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Πραγματικά αξίζει να τη διαδώσουμε γιατί είναι επιτυχία ε, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Thank you, Lina. Ευχαριστώ. Λίνα Σαλαουζιάσκας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. γνωρίζετε ότι είμαι πρόεδρος της ε, ομάδας που έκανε αυτή την έρευνα. Είχα την τιμή να προεδρεύω. Και πρέπει να πω ότι αυτό το έγγραφο που εκπώνησε ο Ξίστοφ Πάτερ θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και υπόδειγμα για την Επιτροπή μας όταν εκπονούμε τέτοιου είδους ενημερωτικά έντυπα και φυλάδια ε, που είναι και ενδιαφέροντα και ελκυστικά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ε, για εθνικές οργανώσεις, για ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κλπ. Ήδη είπε ο εισηγητής ότι σε εννέα ε, συστήματα των κρατών μελών, εκλογικά συστήματα και νόμους, δεν προβλέπεται δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ε, οι άνθρωποι με αναπηρία. Αυτό είναι ένας περιορισμός που αντιτίθεται στην ίδια την αξιοπρεπή ζωή. Η αρχή της αξιοπρεπούς ζωής περιλαμβάνει και την έννοια της ε, αξιοπρεπούς ε, άσκησης του εκλογικού σου δικαιώματος. Σε 11 κράτη-μέλη υπάρχουν προβλήματα κάθε είδους. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές ε, την τελευταία τριετία και τώρα ε, ε, οι άνθρωποι με έχουν περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν στις εκλογές και να ψηφίζουν. Ελπίζω και η δική μας πρωτοβουλία να συνεισφέρει. Μια προσωρινή λύση έχει επιλεγεί σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά πιστεύω ότι η λύση αυτή δεν είναι πολύ αντικειμενική και πολύ συχνά βασίζεται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις. Φέτος έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές και σε πολλά κράτη-μέλη και βουλευτικές ε, ή δημοτικές εκλογές. Γι' αυτό θα ήθελα να ενθαρρύνω τους συναδέλφους μου να διαδώσουν την έκθεση αυτή ε, στους θεσμούς, στις χώρες και στις περιφέρειές τους και στα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πολύ σημαντικό διότι πρέπει να αλλάξουμε κάποιες πρακτικές που είναι βαθιά ριζωμένες στα κράτη-μέλη. Είναι 200, έχουμε μετρήσει 200 ε, τεχνικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους με αναπηρίες να ψηφίσουν. Και πολλές φορές ε, δεν υπάρχει και νομοθεσία για να καταργηθούν αυτά τα εμπόδια και τα προβλήματα. Ευχαριστώ κυρία Μαρή Τσβόλσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι όπως είπε και ο εισηγητής, ο κόσμος συχνά διαμαρτύρεται για τη μεγάλη αποχή στις εκλογές. Και θα πρέπει εμείς να σκεφτούμε πώς θα ενθαρρύνουμε τους πολίτες να ψηφίζουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι πολίτες που πολύ θα ήθελαν να ψηφίζουν. Αλλά επειδή υπάρχουν αυτά τα εμπόδια, πολύ συχνά δεν ψηφίζουν. Σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέρη υπάρχουν διάφορα προβλήματα, είτε τεχνικά είτε νομικά, που τους εμποδίζουν να ψηφίσουν. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ η έκθεση αυτή του κυρίου Πάτερ γιατί αναλύει την κατάσταση στα κράτη-μέλη και στόχος δεν είναι να επικρίνει, να θίξει τα κακό κείμενα, αλλά να ε, προβάλλει τα θετικά παραδείγματα. Και Αυτές είναι βέλτιστες πρακτικές ε, που μπορούν να βρουν μιμητές. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Δεν αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στα εκλογικά τμήματα, χρειάζεται και ενημέρωση έτσι ώστε να έχει και ο καθένας το δικαίωμα να επιλέξει που θέλει να ψηφίσει ε, και να είναι εύκολη πρόσβαση. Επίσης πιστεύω ότι το φυλάδι αυτό θα πρέπει να αναφέρει τις βέλτιστες πρακτικές, όλα τα καλά παραδείγματα και να αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους. Μ' αρέσει επίσης και το ίδιο το φυλάδιο, έτσι. Και καλό θα ήταν να το βγάλουμε και σε ε, μπράι ή και σε ε, μορφή ε, ηχητικού ντοκουμέντου. Ευχαριστώ. Ο Γιάννος Βέλντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σα συγχαίρω για την ε, θαυμάσια το θαυμάσιο κείμενό σα. Όταν διαπιστώνουμε τόσο μεγάλες ε, διαφορές ε, για τη δυνατότητα συμμετοχής των εκλογών από κράτο μέλο σε κράτος μέλος. Ε, Αρωτιέμαι πω θα έπρεπε να υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση ούτως ώστε οι συμπολίτε μας που έχουν αναπηρίε να έχουν όντως ισότητα ευκαιριών όσον αφορά τη συμμετοχή. Είναι το ερώτημά μου. Pietro Barbieri. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Κρίστοφ για τη δουλειά του και την ομάδα μελέτης. Αλλά να είμαστε λίγο ξεκάθαροι με το τι συμβαίνει. Εδώ, αυτό που προκύπτει το έγγραφο είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων πολιτών που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου. Ας ξεχάσουμε για λίγο και σας προσκαλώ όλους, ας ξεχάσουμε για λίγο τον ώρα αναπηρίας διότι μας πάει κάπου αλλού το θέμα αυτό. Εδώ μιλάμε για πολίτες όπως όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αυτό θα έπρεπε να κηρύξει μέχρι και παράνομες εκλογές σε μια χώρα. Είμαι πάρα πολύ ευστηρός ως, προ αυτό, ως προς αυτό και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Μιλάμε για αριθμό πολιτών που θα μπορούσαν να συγκριθούν με τον πληθυσμό της μεγαλύτερης χώρας της Ευρώπης, αυτή, είναι το μεγαλ... αυτής που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό. Μιλάμε για διαστάσεις του φαινομένου που είναι τεράστιες. Το γεγονός ότι υπάρχουν ε, άτομα, πολίτες που δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είναι ένα γεγονός πολύ σοβαρό, ε, σοβαρότατο Όλοι πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση και ζητώ από τον Πρόεδρο να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, γιατί το θέμα αυτό πραγματικά μας καίει. Μιλάμε για τη δημοκρατία. Οι μειονότητες πρέπει να προστατεύονται, αλλά ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ μιλάμε για την ίδια τη δημοκρατία. Ευχαριστώ τον Κρίστοφ. Ευχαριστώ Πιέτρο. Μέρις Γιώστα. Κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή. Πολύ εμπεριστατωμένη η γνωμοδότηση και η ενημέρωση που μας έκανε. Μ' αρέσει. Το ότι παρουσιάζει τόσο πολύ καλά τις νομικές δυσχέρειες και κάνει όμως και προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Λέει ότι είναι σημαντική η προσβασιμότητα. Η οργάνωσή μου καθημερινά ασχολείται με αυτά τα θέματα πρόσβασης. Είναι πολύ περίπλοκο θέμα. Υπάρχουν διάφορα είδη αναπηριών, ε, χρόνιες ασθένειες και γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ διαφορετικές λύσεις. Και δεν είναι απλό να καταλήξουμε σε τέτοιες λύσεις. Γι' αυτό σε κάθε κράτος μέλος ε, πρέπει να κάνουμε σημαντικά βήματα. Και κάτι που είναι πολύ καλό σε αυτή τη γνωμοδότηση είναι ότι παρουσιάζεται και το νομικό πλαίσιο και τα θέματα διεθνούς δικαίου που μας υποχρεώνουν να οδεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει, επικυρώσει αυτές τις διεθνείς συμβάσεις. Άρα και για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να εγγυώνται τη δυνατότητα συμμετοχή στι εκλογέ. Ψήφου. Στην Εστονία μπορεί να ψηφίσει και ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συμμετάσχουν πολύ περισσότερο. Από το σπίτι τους μπορούν να ψηφίσουν. Μπορούν να αξιοποιήσουν ε, τεχνική βοήθεια για να ψηφίσουν και ελπίζω ότι αυτές οι τεχνικές λύσεις και η νέα ψηφιακή πραγματικότητα θα βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία στο μέλλον, ούτως ώστε να συμμετέχουν περισσότερο στο πολιτικό γίγνεσθε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Άγνες Τέλμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Disabilities έχει ξεκινήσει μία εκστρατεία για να ενθαρρύνει τα άτομα με αναπηρία να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές. Στην εκστρατεία αυτή τονίζουμε ότι πολύ, λίγοι, πολύ λίγα άτομα με αναπηρία συμμετέχουν στις εκλογές και θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα άτομα με αναπηρίες να ασκήσουν το δικαιωμά τους ψήφου και συμμετοχής λοιπόν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Είναι, όλα αυτά έγιναν μάλλον το 2009, έκτοτε έχουν περάσει 10 χρόνια και Ακόμη έχουμε γύρω στα 50 εκατομμύρια ατόμων με αναπηρία, συμπολιτών μας ε, παντού στην Ένωση, που ακόμη δεν έχουν δυνατότητα να ψηφίσουν. Πρέπει λοιπόν να καταρτήσουμε τα άτομα με αναπηρία για τα πολιτικά τους δικαιώματα και πρέπει να καταλάβουν και οι κυβερνήσεις ότι πρέπει να παράσκουν τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας αυτούς να ψηφίζουν. Δεν αρκεί ευαισθητοποίηση. Πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένα τις αναγκαίες διευκολύνσεις στους συμπολίτε μας. Και είναι δουλειά αυτό. Πρέπει λοιπόν να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και επίσης να τονίσουμε ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα η ψήφος και πρέπει να ισχύει για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Άγνες. Ο Γιάτσε Κράφτσικ δεν, ε, δεν τον γράψαμε στο σύστημα εδώ, αλλά παρακαλώ να του δώσουμε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Συζητήσαμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας από την Πολωνία για τις Βρυξέλλες ε, για αυτή την έκθεση και ξέρω πόσο σημαντική είναι η έκθεση αυτή για μένα. Προσωπικά ενδιαφέρεσαι και δεσμεύεσαι για το θέμα. Εσύ έχεις ε, πρώτο χέρι εμπειρία ε, για τα άτομα αυτά. Έχω κάθε σεβασμό για την εργασία σου, Ξιστόφ. Και εδώ κάνεις μία περιγραφή, μία διάγνωση της κατάστασης και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πραγματικότητα που περιγράφεις. Τα άτομα σε αυτή την ε, κατηγορία συμπολιτών μας πρέπει να μπορούν επιτέλους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Δεν αρκεί όμως να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα. Πρέπει να δράσουμε και οι, τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ψηφίσουν. Μια σύντομη πρόταση από την πλευρά μου. Στην έκθεσή μου, που ελπίζω σήμερα να εγκριθεί ομόφωνα, ελπίζω να είναι βάση για να υπάρξει μια συνέχεια σε πολλούς τομείς γιατί χρειαζόμαστε να κάνουμε εργασία λόμπι με αποφασιστικότητα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στείλει σαφέ μήνυμα ότι τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρία πρέπει να τηρούνται και ε, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να προωθηθούν. Πρέπει όμως και στα κράτη-μέλη να υπάρξει συνέχεια. Η έκθεση αυτή πρέπει να σταλεί παντού όλες ε, οι αρχές και όλοι που είναι αρμόδιοι για να διορθωθεί η κατάσταση πρέπει να τη λάβουν. Και είναι πολύ επίκαιρη η έκθεση αυτή. Θα έλεγα ότι είναι ιδανική η συγκυρία που υποβάλλεται, αλλά θα ήθελα σε πέντε χρόνια να επανέλθουμε στο θέμα αυτό για να κάνουμε μια, έναν απολογισμό, για να δούμε τι ακριβώς θα έχουμε επιτύχει μέχρι τότε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δύο λεπτά για να απαντήσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα καλά σας λόγια. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Με δύο τρόπους μας λέει η έκθεση. Ε, μία από την κορυφή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η δεύτερη από τη βάση, ε, σε εθνικό επίπεδο. Από την κορυφή που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό αφιερώνεται το ε, κεφάλαιο 4 και έχουμε και στις δύο περιπτώσεις ε, νομικά βήματα και νομοθετικά που πρέπει να κάνει το νεοεκλεγέν ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, είτε να αλλάξει ο εκλογικό νόμος του 1976, είτε να αντικατασταθεί τελείως. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, το ευρωπαϊκό. Μετά είναι από τη βάση τα κράτη-μέλη όλα μαζί γίνεται αυτό. Βεβαίως, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίσει νομικά να κατοχυρώσει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν σε άλλη χώρα από την πατρίδα τους και λένε ότι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν και αυτό το λέει το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκλογική πράξη του 1976. Δεν υπάρχει λόγος να ισχύει κάτι διαφορετικό για τους Ευρωπαίους πολίτες με αναπηρίες. Αυτή ήταν κορυφή. Η βάση τώρα θα αλλάξει από το εθνικό επίπεδο με την πίεση των διαφόρων οργανισμών και οργανώσεων που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Σχεδόν πάντα ε, είναι οργανώσεις όπου συμμετέχουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι με αναπηρίες. Και θα πρέπει η φωνή τους να ακούγεται δυνατά σε όλη την Ευρώπη και στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί. Γιατί πιστεύω ότι Είναι διαφορετικό να ζητούν οι ίδιοι ε, οι άνθρωποι με αναπηρίε και οργανώσεις τους τα δικαιώματά τους και να τα διεκδικούν και διαφορετικό είναι να τα διεκδικεί ε, και η κοινωνία των πολιτών και ε, κάποιες άλλες οργανώσεις εξωτερικές. Γι' αυτό σας ζητώ να βοηθήσετε να φτάσει σε όλη την Ευρώπη η έκθεση. Την έχετε στα χέρια σας βέβαια στους φακέλους σας, αλλά έχετε και σε έξι γλώσσες εκτός της εθούσης ε, τις εκθέσεις αυτές. Σε λίγες εβδομάδες θα τις έχετε και σε όλες τις γλώσσες για να τις μοιράσετε στις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών έτσι ώστε να πιέζουν εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ Ξύστοφ. Και πριν προχωρήσουμε στη ψηφοφορία θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια ε, είναι πολύ σημαντικά αυτά. Εδώ μιλούμε για ένα θεμελιώδες δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Έτσι δεν είναι. Και επειδή με είχε ενημερώσει ο Ξυστοφ για το περιεχόμενο του κειμένου, παρουσίασα ήδη από την περασμένη εβδομάδα το κείμενο αυτό στον πρόεδρο Ταγιάννη, ο οποίος ε, θα ήθελε, προτίθετο να έρθει σήμερα ε, για την παρουσίαση ε, αυτού του θέματος, αλλά δεν μπόρεσε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και αυτός το θεωρεί σκάνδαλο που πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια σκληρή μάχη για να αλλάξει αυτό που πρέπει να αλλάξει. Και είχα την ευκαιρία την περασμένη εβδομάδα να παρουσιάσω την έκθεση αυτή και στη διαμεσολαβήτρια, στην κυρία Ορέιλη, η οποία ε, πραγματικά εντυπωσιάστηκε από την ε, έκθεσή μας, από την ποιότητα της εργασίας μας. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο και βεβαίως είναι στη διάθεσή μας για να συνεργαστούμε. Θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να αλλάξει η ε, ημερήσια διάταξη της ετήσιας ε, συνόδου των εθνικών ε, αρχών, ε, διαμεσολαβητών και συνηγόρων του πολίτη. Ε, έχει αρχίσει λοιπόν αυτή η προσπάθεια και θέλω πραγματικά να σας ζητήσω με την ψήφο μας να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και προς τα θεσμικά όργανα ότι εμείς έχουμε εργαστεί σοβαρά αλλά θέλουμε και τη δική τους βοήθεια για να συνεχιστεί αυτή η σοβαρή προσπάθεια. Έρχεται η ψηφοφορία. Subcommittee zero. 052 ε, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωφέλει για τους πολίτες και σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών. Μιχάη Βάσκου και Στεφάν Μπιφτό, οι συγητές τους καλώ στο Προεδρείο για να μας παρουσιάσουν την έκθεσή τους. se paladisait, donc... Et... Euh, <laughs> eh, mais toi, Yes, please go. Thank you very much and uh, good afternoon to everybody. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Όπως ακούσατε ήδη, ε, η Ρουμανική Προεδρία ζήτησε τη γνωμοδότηση αυτή, τη διερευνητική γνωμοδότηση και η διαδικασία ήρθε σε δύο τμήματα στο τμήμα το οικονομικό ΕΚΟ και στο ΞΟΚ το κοινωνικό. Και θέλω να ευχαριστήσω για την υποστήριξη, να σας ευχαριστήσω όλους σας και στα δύο τμήματα. Όπως βλέπετε είναι ένα μακροσκελές κείμενο. Εμείς θέλαμε να είναι και μεγαλύτερο, όπως σας είπα, θα μπορούσαμε να είχαμε γράψει και ένα τόμο και δύο για αυτό το θέμα, ε, εάν θέλαμε να συμπεριλάβουμε όσα ακούσαμε στις τρεις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής αυτής. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της υποεπιτροπής, μα της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ε, ε για ε, την προφορική του συνεισφορά, τη γραπτή του συνεισφορά, αλλά και τον συνεισηγητή, γιατί χρειάστηκε να πάρουμε πάρα πολύ γρήγορα αποφάσεις και καταλήξαμε σε ένα πολύ καλό τελικό κείμενο, κατά την άποψή μου. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση. Βεβαίως, η γνωμοδότηση αυτή είναι πολύτιμη για την ΕΟΚΕ και για την πολιτική συνεδρίαση στο Συμπίου. Γι' αυτό προσπαθήσαμε πρώτα απ' όλα να δώσουμε τη δική μας άποψη για το τι μέλη γενέστε, για το πώς θα προχωρήσουμε και με κάποια συμπεράσματα από παρελθούσες νομοδοτήσεις που είχαμε γκρίνει. Ταυτόχρονα όμως θελήσαμε να ε, αναγνωρίσουμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον, τα ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες από τη συμμετοχή της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικά νομίζω ότι το καταφέραμε. Ε, ξέρω ότι είναι το κείμενο μακροσκελές, επαναλαμβάνω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έτος, έτος ευρωεκλογών το 2019. Είναι ένα έτος όπου τα κράτη-μέλη αναμένεται να πάρουν σε δύο μήνες στο συμπίου μια πολιτική απόφαση. Και όταν συζητούμε για τα ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες και έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερώσει, Φυσικά θα πρέπει να αναφέρουμε και την οικονομική διασύνδεση, την ε, αυξημένη πολιτική και ε, κοινωνική συνεργασία, την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και βεβαίως την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών που δίνει αμέτρητες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες. Επίσης, Υπάρχουν ε, και συστήματα υγείας, αμοιβαιότητα. Όταν διαμένουν οι πολίτες σε μια άλλη χώρα, εποφελούνται από το σύστημα υγείας. Υπάρχει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που βοηθάει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Όταν γίνεται λόγος λοιπόν για την οικονομική βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη εσωτερική ενιαία αγορά στον κόσμο και χρησιμοποιεί το δεύτερο μεγαλύτερο νόμισμα. Είναι η πρώτη εμπορική δύναμη και ε, ε, ο πρώτος δωρητής ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. Επίσης, αναγνωρίζουμε ότι όταν ολοκληρωθεί ο ΝΕ, ναι, θα μπούμε σε μια νέα εποχή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα ενιαίο νόμισμα που μειώνει σημαντικά το κόστος των συναλλαγών και περιορίζει, καταργεί τους ε, κινδύνους από το εξωτερικό εμπόριο ε, και επίσης τους επενδυτικούς κινδύνους. Και επίσης με τα παγκόσμια πρότυπα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι ε, πλούσιες και ευημερούσες, αλλά υπάρχουν τεράστια ελλείμματα και διαφορές στην κοινωνική συνοχή και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις διαφορές. Σύγκληση προς τα πάνω, ε, καλύτερη ευημερία ε, και καλύτερη κινητικότητα. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα σταματήσω εδώ και θα αφήσω το Στεφάν να συνεχίσει και στη συνέχεια θα περάσουμε στις τροπολογίες που ε, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας, ιδιαίτερα στην τελευταία συνεδρίαση που είχαμε στην Υποπιτροπή μας και ε, όλα αυτά ε, τα οποία συμφωνήσαμε και προσπαθήσαμε να τα εντάξουμε στο κείμενο. Σεβόμαστε όλα τα μέλη, βέβαια κάποιες τροπολογίες αναγκαστήκαμε να τις απορρίψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Στεφάν Μπίφτο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Είναι σημαντικός ο τίτλος ε, της νομοδότησης. Το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ένωσης ωφέλει για τους πολίτες. Δύο στοιχεία. Είναι αρκετά τα ωφέλη για τους πολίτες ε, που είναι πια τόσο συνηθισμένα στην καθημερινή ζωή μας που οι πολίτες μας σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θεωρούν δεδομένα. Δεν, δεν, δεν καταλαβαίνουν πλέον ότι είναι ωφέλη που απορρέουν ή οφείλονται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και είναι σημαντικό να το θυμίσουμε αυτό. Έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύντομο κατάλογο που παραθέτουμε ε, και δεν είναι τυχαία όλα αυτά ε, και πολύ συγκεκριμένα ε, όπως είναι η εναρμόνιση στις ε, πρίζες ας πούμε στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά υπάρχουν και τα θέματα του μέλλοντος και εκεί δεν θέλησαμε να είμαστε σε μία άρνηση δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για ένα τέτοιο σύστημα από το να είσαι καθυλωμένο στην άρνηση, γιατί καταλήγεις σε ακραίες καταστάσεις. Τι είναι η άρνηση ότι να αρνηθούμε να δούμε ότι οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επικρίνουν. Υπάρχει ένας πειρασμός ε, που είναι ο δρόμος της ευκολίας από διοπομπέως ε, τράγους. Οι λαϊκιστές, η ρωσική προπαγάνδα, η ε, αντισυστηματική, η αντισυστημική μάλλον κατά του συστήματος, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί όμως έχουν ένα βάρος στην κοινή γνώμη, ε, άρα ε, εκφράζουν τις ανησυχίες της κοινή γνώμης και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει απαντήσεις σε αυτές τις αγωνίες. Γιατί αν στην Ευρώπη έχουμε μια περιφερειακή Ευρώπη ξεχασμένη της παγκοσμιοποίηση, για να το διατυπώσω έτσι, ε, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει δύσκολο μέλλον να αντιμετωπίσει. Merci bien, Ευχαριστούμε, Στεφάν λίγη η λίστα των αγορητών, ο κατάλογος των αγορητών. Ξεκινάμε με τον κύριο Λέσκι που ήταν πρόεδρος της ομάδας εργασίας. Ναι, ήμουν πρόεδρος της υποεπιτροπής που ασχολήθηκε με την εκπόνηση της επιτροπής. Συγχαίρω τους εισηγητές ε, για το, πόρισμα, το αποτέλεσμα των κοινών εργασιών. Δεν ήταν εύκολη η συζήτηση. Ένα έγγραφο πολλά ζητήματα που αφορούν το θέμα αυτό, το μέλλον της Ευρώπης. Η έκθεση σκοπό έχει να καλύψει ο σταθερό περισσότερα. Αλλά χρειάστηκαν τροπολογίε από του συναδέλφου τη ομάδα 2. Τροπολογίε που θα βελτιώσουν την εξισορρόπηση κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων στην έκθεση αυτή. Για να καλύψουν και όλε τι απόψει τη ΕΟΚΕ για το μέλλον τη Ευρώπη. Το πλέον σημαντικό για μένα στην έκθεση αυτή είναι το κεφάλαιο για την κοινωνική πρόοδο γιατί προέρχομαι από χώρα που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 και έχει αποφεληθεί τα μάλα από την ε, ε, συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ ε, πρέπει να ενισχύσουμε τους μισθούς και τις συνθήκες διαβίωσης. Πρέπει να προσέξουμε να μην ε, κάνουν οι εργαζόμενοι, να μην παίρνουν διαφορετικές αμοιβέ για την ίδια δουλειά, εφόσον μιλάμε για τα ίδια επίπεδα παραγωγικότητας. Γιατί κάποιοι κερδίζουν πέντε φορές λιγότερο από ό,τι οι συνάδελφοί του στη Δυτική Ευρώπη. Εδώ λοιπόν ε, πρέπει να προσέξουμε την αύξηση των μισθών ε, ανάλογα με την εργασία που προσφέρεται και να κοιτάξουμε να υπάρχει ένα πλαίσιο για τους κοινούς μισθούς Ω προ τη σύγκληση λοιπόν των μισθών, θα πρέπει όλα αυτά να τα κοιτάξουμε γιατί δημιουργούν αντιευρωπαϊκά ε, συναισθήματα. Πρέπει η Ευρώπη να εργάζεται για όλου και να προσφέρει σε όλου, όχι μόνο σε λίγου. Οι τροπολογίε που υποβλήθηκαν στην έκθεση αυτή επικεντρώνονται σε αυτό το θέμα ακριβώ. Τι δίκαιε κοινωνίε, τι δίκαιε ευκαιρίε, ίσε ευκαιρίε, τι ίσε συνθήκε εργασία για όλου ε, και τη λειτουργία τη δημοκρατία. Κυρίω ε, και την αυτονομία την αυτόνομη δράση των κοινωνικών εταίρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ζενεβιεύ Σοβινή για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να πω ότι προσωπικώς εργάστηκα στην ομάδα εργασίας αυτή, που ήταν ε, πολύ πλούσια σε συζητήσεις, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα, για να προασπιστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες και τα συμφέροντα των πολιτών. Και θα πρέπει να έχουμε πάντοτε και ένα κριτικό, μια κριτική θεώρηση του θέματος. Εδώ λοιπόν για την πρώτη έκθεση που μας απασχόλησε, το Συμπίου και παραπέρα, τα δύο κείμενα αυτά κοιτάξαμε να τα συνδυάσουμε λιγάκι. Και γι' αυτό συντάξαμε τη συγκεκριμένη αγνοδότηση με γνώμονα και τα όσα έλεγε η άλλη έκθεση και του Συμπίου ε, για το περιβάλλον ειδικώ και κοιτάξαμε να τα προσαρμόσουμε ώστε η διάσταση της βιωσιμότητας που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ να καλύπτεται επαρκώς. Στο πρώτο κείμενο ειδικά, ε, στο Συμπίου και πέρα από αυτό. Για μένα λοιπόν η διάσταση της βιωσιμότητας είναι πολύ σημαντική για το τι μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη στο παρόν και στο μέλλον. Ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στα δύο αυτά τα κείμενα και πώς συνδυάζονται. Πρέπει να τα δει κανεί παράλληλα και να έχει αυτή τη θεώρηση που είναι θετική και με κριτικό βλέμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι μπορεί να προσφέρει στους πολίτες. Επίσης, να μην ξεχνά και τη διάσταση Ανατολή-Δύση, Ανατολικές Δυτικές χώρες που συζητήθηκε πολύ στην ομάδα και καλύπτεται και αυτό αρκετά από το κείμενο. Ευχαριστούμε. Άντι Μελέν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πω ότι και εγώ συμμετείχα στην τρίτη συνεδρία της ομάδας εργασίας και πρέπει να πω για το περιεχόμενο του κειμένου ότι σωστά εντοπίζει ως καθήκον μας να, να εντοπίσουμε για τους πολίτες το τι όφελο αποκομίζουν από τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εργόδράση δράση του. Όμω πρέπει να παραμένουμε και αντικειμενικοί σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το τι δεν κάνει ή δεν κάνει επαρκώ. Εδώ λοιπόν κυρίως έχω υπόψη τα κοινωνικά ε, επιτεύγματα, την ε, κοινωνική πρόοδο για αυτούς τους ε, πολίτες. Ο κ. Μπιφτό έχει δίκιο όταν λέει ότι χρειάζεται μια συγκεκριμένη χειροπιαστή απάντηση για τις ανησυχίες των πολιτών. Ε, πρέπει να θυμίσουμε ότι οι κοινωνικές ανισότητες εντείνονται. Θα, ε, δεν έχουμε πετύχει να εξαλείψουμε τη φτώχεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο πλούτος ε, αυξάνεται και συγκεντρώνεται σε κάποια χέρια. Πρέπει η αύξηση της παραγωγικότητας να οδηγήσει και σε αναλογική αύξηση των μισθών και των αμοιβών. Δεν θα μιλήσω καν για την ποιοτική κοινωνική ασφάλιση, που σίγουρα δεν είναι προσβάσιμη πλέον σε όλου, ή τουλάχιστον όχι σε όλου του πολίτε των όλων των κρατών μελών. Για αυτού λοιπόν του λόγου, θέλω να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι οι τροπολογίε που υποβάλαμε μαζί με μια σειρά συναδέλφων από την ομάδα 2, σκοπό έχουν να υπογραμμίσουν τι προσπάθειε που απομένουν να γίνουν σε κοινωνικό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πιέσουμε και με αυτές τις τροπολογίες να εξισορροπηθεί καλύτερα το κείμενο για να παραμείνει εύληπτο και ε, εύστοχο καθώς και συνεπές σε σχέση με τα προηγούμενα κείμενα που εγκρίναμε. Δηλαδή το να αφουγκραστούμε τους πολίτες της Ευρώπης για ένα βιώσιμο μέλλον. Έχουμε εδώ δύο γνωμοδοτήσεις ε, που ακόμη και αν τις συναρτήσουμε θα πρέπει να έχουν εξισορροπηθεί ε, εσωτερικά πρώτα η καθεμιά με τον εαυτό της Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από τους εισηγητές να δεχτούν μια σειρά από, από τροπολογίες που θα επιτρέψουν αυτήν την σωστή εξισορρόπηση. Ευχαριστώ. Και για λίγα λεπτά θα αφήσω το λόγο στην ε, την Προεδρία στην Ιζαμπέλ Κάνιο. Θα επανέλθω εντάχει. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Μπαρμπούτσι. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω και εγώ ότι στο ίδιο πνεύμα με τους συναδέλφους που προηγήθηκαν, τον Άνταμ και την Άννα από την ομάδα εργασίας, ε, συμφωνώ. Συμμετείχα στην ομάδα μελέτης και ήταν πολύ challenging η δουλειά μας. Ε, ήταν κάτι που πραγματικά μας υποχρέωσε να στύψουμε το μυαλό μας. Ε, το συζητήσαμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την αφορμή του Συμπίου και πέρα. Και μετά θα τα ξαναδούμε και σε άλλες νομοθετήσεις όπου είμαι συνεισηγήτρια και εγώ για την παραπληροφόρηση. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, όλες οι νομοθετήσεις έχουν έναν κοινό στόχο και πάνε σε μια κοινή κατεύθυνση. Εδώ πιστεύω ότι ο εισηγητής και ο συνεισηγητής του ε, Δραμάτισαν ρόλο ανέλαβαν μάλλον ρόλο, αρκετά δύσκολο. Χρειάστηκε να δουλέψουν με μια ομάδα μελέτης που είχε πολλά να προτείνει. Διαφορετικά κιόλα. Προέβαλε διαφορετικά επιχειρήματα, διότι το θέμα είναι αχανές. Επίσης υπήρχε μεγάλη διάθεση συνεργασίας και μεγάλη διάθεση συμβιβασμού και ανοιχτό πνεύμα. Πρώτα να το αναγνωρίσω στον εισηγητή. Όμως και εγώ θεωρώ ότι το κείμενο αυτό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, πρέπει κι άλλο να το γυαλίσουμε, να το χτενίσουμε και να το βελτιώσουμε από κοινωνικής πλευρά. Γι' αυτό υποβάλαμε σχετικέ τροπολογίε. Αν μιλάμε για ωφέλη προ του πολίτε, μην ξεχνάμε ότι η καρδιά αυτών αφορά τα κοινωνικά δικαιώματά του. Ο κύριος Πετσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν πήρα μέρος στην ομάδα μελέτης. Όμως ε, διάβασα το κείμενο και μου άρεσε. Θα ήθελα πάντως να μην θεωρηθεί ως οριστικό και τελεσίδικο το κείμενο το πέρας του χρόνου. Στο μέλλον θα πρέπει να κάνουμε και άλλες προσπάθειες, διότι εάν συγκρίνω τις προσδοκίες που έχουν από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτες, από την Ευρώπη ε, πριν από 25 χρόνια όταν ξεκίνησα εδώ στην Επιτροπή, και τις προσδοκίες του σήμερα, βλέπουμε τεράστια διαφορά. Η διαφορά αυτή κατά πάσα πιθανότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρώπη ε, τα τελευταία χρόνια σίγουρα προέβαλε τις μεγάλες ευρωπαϊκές αξίες, όμως τι συνέβη, οι πολίτες έχασαν αυτό το συνέστημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, Γιατί πολλά από τα θέματα που τους ενδιέφεραν πάνω από όλα δεν φάνηκε να φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Για την ώρα δεν έχουν ε, ασφάλεια για το αυτοκίνητό τους, ας πούμε, που να ισχύει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτες. Ή μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά δεν επιτρέπεται να πάρουν όσα μπουκάλια κρασί θέλουν από μια χώρα στην άλλη. Διότι μερικοί προβάλλουν ειδικού φόρου και άλλα εμπόδια. Το μεγάλο μα λοιπόν πρόβλημα, και ολοκληρώνω με αυτό γιατί το θέμα είναι τεράστιο, ε, είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια παραπάνω προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γίνει πιο ισχυρή. Πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ε, δικαιώματα ω προ την εσωτερική αγορά για να μπορέσει να γίνει επιτέλου μια αυτή η αγορά. Σήμερα οι πολίτε ξέρουν ότι δεν έχουν ενιαία αγορά με το χρόνο θα θέλαμε να ξεπεράσουμε αυτές τις, ε, αυτούς τους διχασμούς, για να τους πω έτσι, τον κατακαιρματισμό που τελικά δεν αφήνει τους πολίτες να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Πάντως και πάλι συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Σμιτ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Ιζαμπέλ. Συμφωνώ με τους προηγούμενους όταν αρχίσαμε να ασχολούμεθα με το κείμενο αυτό, διαπιστώσαμε σε κάποια φάση ότι είναι ένα δεύτερο κείμενο για το ΣΥΠΙΟΥ. Και αυτό μάθαμε ότι θα υπάρχει και ένα άλλο κείμενο για το ΣΥΠΙΟΥ και μας εξενέβρισε αυτό το γεγονό όταν το διαβάσαμε. Αλλά τελικά είδαμε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιώδης επικάλυψη και τα διαχωρίσαμε. Και καλέσαμε τους συζητητές να τα συζητήσουμε και τελικά όλα αυτά ήταν πολύ επικοδομητικά και συμφωνώ με όσους είπαν ότι τα δύο κείμενα αυτά πρέπει να τα διαβάσουμε από κοινού. Και αν τα διαβάσουμε από κοινού, που θέτουν διαφορετικά ζητήματα. Παρακαλώ οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν να ειδωθούν στη λογική της σημερινής συζήτησης της κοινή αντιμετώπισης που αποδέχτησαν και οι συγητές των δύο κειμένων. Γιατί αλλιώς υπάρχουν κάποιες ε, ε, αντιρρήσεις. Θα μπορούσε κανείς να έχει αντιρρήσεις για αυτά που συζητήσαμε. Ζητώ λοιπόν τους συζητητές, ε, κοιτάξτε τις τροπολογίες, ούτω ώστε να υπάρχει συνέπεια μεταξύ αυτών των δύο κειμένων. Και γι' αυτό να τι αποδεχτείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κράτσικ, ο κύριος Κράτσικ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλό κείμενο, νομίζω. Παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και λέει με ένα πολύ σφαιρικό τρόπο τι είναι το, επιχείρημα, το εγχείρημα της Ένωσης. Καταλαβαίνω γιατί κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι ενδιαφέρονται μόνο για το κοινωνικό τμήμα του κειμένου αυτού. Αλλά εγώ θέλω να μας ενθαρρύνω να διαβάσουμε συνολικά το κείμενο, όχι μόνο το κοινωνικό τμήμα. Διότι νομίζω ότι αν δεν δεχθούμε τη βασική προϋπόθεση, ότι αν δεν είναι ανταγωνιστική η οικονομία μας, δεν θα έχουμε λεφτά για την κοινωνική προστασία στο επίπεδο που θέλουμε. Πάντα θα έχουμε ένα πρόβλημα να, επι... να επικοινωνήσουμε με το κοινό. Δεν είναι είτε είτε. Δεν αποκλείονται. Η Ένωση που δαπανά γύρω στο 50% των κοινωνικών δαπανών για το 20% του πληθυσμού είναι χώρος κοινωνικής αδικίας. Πρέπει να δείξουμε τα πράγματα πώς, ε, όπως είναι. Πρέπει να σταματήσουμε να διαμαρτυρόμεθα. Κανείς δεν δαπανά για την κοινωνική προστασία περισσότερα από εμά. Αλλά για να μπορέσουμε να τα δαπανίσουμε πρέπει να εργαστούμε όλοι σκληρά όχι απλώς να απαιτούμε περισσότερα χρήματα από τους φορολογουμένους για κάποιους δικαιούχους και κάτι άλλο που το κάνουμε κάθε καλή πίστη. Δεν ισχύει ότι η Ανατολική Ευρώπη έχει το ίδιο επίπεδο παραγωγικότητας με τη Δυτική Ευρώπη. Και επίσης αν δούμε την ε, διαφορά αγοραστικού επίπεδου δεν είναι τόσο μεγάλε διαφορέ μεταξύ Ανατολή Δύση. Εντάξει, υπάρχουν διαφορέ, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλε. Και δεν είναι δύσκολο να αρχίσει κανεί να ε, τυπώνει χρήμα. Και νομίζω ότι οι χώρε που είναι οι πιο χρεωμένε είναι και οι πιο χαλαρέ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους συντάκτες του κειμένου αυτού. Δεν συμμετείχα στη σύνταξή του. Και μόνο τώρα το είδα, λίγο πριν την ολομέλειά μας. Αναφέρεται σε κοινωνικά θέματα το κείμενο και το ανέφεραν και διάφοροι ομιλητέ. Αλλά εγώ θέλω να τονίσω μια άλλη πλευρά Καλύπτει βέβαια πολλά θέματα το κείμενο αυτό. Και ευχαριστώ πολύ τους συντάκτες γιατί όντως επιδεικνύουν το αναγκαίο θάρρος για να μιλήσουν για τον ανοιχτό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η Ευρώπη. Η Ευρώπη και πολλά κράτη-μέλη δυστυχώς ε, είναι σε ένα σταυροδρόμι. Θα συνεχιστεί ε, ο ανοιχτός χαρακτήρας της κοινωνίας και οικονομίας μας ή θα αρχίσει ο προστατευτισμός. Για μένα ο προστατευτισμός δεν θα ωφελήσει τους πολίτες. Και ιδίω τώρα, άμα δούμε τι γίνεται γύρω μας. Απογοητεύθηκα όταν πριν από μια εβδομάδα είδα να λέγεται στο Κοινοβούλιο ότι δεν θα δοθεί διαπραγματευτική εντολή στην Επιτροπή για να ξεκινήσουν οι εμπορικέ διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, ψηφίσω το παρόν κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Βόλφαν Γκράιχ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το παραδέχομαι ότι ήταν δυσχερέ το έργο. Πολλά θέματα αναφέρθηκαν. Και ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει συνέπεια στα κείμενά μας. Ιδιαίτερα ε, συνέπεια και με την ε, γνωμοδότηση για το συμπίου που ψηφίσαμε. Νομίζω θα ήταν καλό να κρυθούν δύο τροπολογίες. και μάλιστα με ευρία πλειοψηφία για να υπάρξει αυτή η συνέπεια με το προηγούμενο κείμενο. Όμω δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένο με το κείμενο και το είπα και στο στην ειδική ομάδα δεν υπέβαλα τροπολογίε. Για κάποια σημεία έχουμε ήδη αποφασίσει που αναφέρονται στο κείμενο αυτό και νομίζω ότι ορισμένα που λέγονται εδώ δεν ισχύουν. Για παράδειγμα, το 5-6 για την εμπορική μας πολιτική. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό, με αυτά που λέει εδώ. Ότι η Ένωση έχει συμφωνήσει Ε, σε μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες ε, για να υπάρξει ελεύθερες, ε, να υπάρξει να υπάρξει ελεύθερο εμπόριο στι υπηρεσίε και παράλληλα να γίνει σεβαστό και το περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Για ποιε λέτε. Έχουμε τη συμφωνία για την Ιαπωνία, έχουμε τη συμφωνία με τον Καναδά, τα έχουμε συζητήσει. Και δεν θεωρούμε ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα περιβαλλοντικά θέματα διασφαλίζονται με τον ίδιο τρόπο όσο το ελεύθερο εμπόριο. Μα τα είπαμε αυτά εδώ πέρα και Φυσικά στηρίζουμε την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στις περαιτέρω προσπάθειες για ένα δίκαιο πολιετές σύστημα. Δεν είναι αυτή η βάση της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής. Νομίζω ότι επαναρχόμεθα σε θέματα που τα έχουμε συζητήσει και απορρίψει εδώ. Και η παράγραφος για την αμυντική πολιτική. Στην Επιτροπή έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις. Έχω πραγματικά προβλήματα με αυτή τη γνωμοδότηση για να υπερψηφίσω αυτά τα δύο τα δύο ε, σημεία. Εάν δεν περάσουν οι δύο τροπολογίες της ομάδας δύο θα έχω πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάκο Ποσίβατσεκ και ζητώ συγγνώμη για την προφορά. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Πολύ ωραία το είπατε. Θα ε, ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές ε, για την γνωμοδότηση αυτή. Πραγματικά οφείλω να πω ότι το θέμα είναι ευρύτατο. Αυτό που έπρεπε να καλύψετε. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κείμενο για το ΣΥΜΠΙΟ. Ε, καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης τώρα, σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, πολλοί πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαρωτώνται και τι ωφελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ωφέλη οι πολίτες τα θεωρούν αυτονόητα και προφανή. Και η εξολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα μάτια των πολιτών είναι και αντικειμενική και υποκειμενική για τη χρησιμότητα, για την ωφέλειά της, για το εάν βοηθάει να λύνονται τα προβλήματά τους και να αντιμετωπίζονται οι σημερινές προκλήσεις. Θα πρέπει να τονίζουμε πάντα αφενός τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά ε, να μην αποσιωπούμε και τα προβλήματα που απομένουν ακόμα να λυθούν. Γι' αυτό κάναμε προτάσεις ε, ε, στην ομάδα 2 έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια στο κείμενο για το Συμπίου και Επέκεινα. Τα είπαν και προηγούμενοι μιλητές όλα αυτά. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχυθεί, τότε θα μπορεί να λύνει καλύτερα τα προβλήματα των πολιτών από οποιοδήποτε κράτος ξεχωριστά έχουμε εσωτερική ενία αγορά, ενία αγορά με κοινού κανόνε, αλλά και καλύτερες προποθέσει μπορούμε να δημιουργήσουμε για τους πολίτες μας. Με τις τροπολογίες μας μπορούμε να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω το κείμενο, αλλά και περιοδικά να έχουμε τέτοιες γνωμοδοτήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να τονίζουμε ε, τα ωφέλη για τους πολίτες και να τα αξιολογούμε κάθε φορά γιατί μπορεί ακόμα πολλά να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες της. Ωραία. Ο εισηγητής για να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ε, τοποθετήσεις και τις παρεμβάσεις σας. Πάρα πολύ σύντομα. Κύριε Προδολεύσκη, όπως είπαμε, βεβαίως το κεφάλαιο 6 είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο, όλο το έγγραφο είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ συνεπές και συνεκτικό. Η κυρία Σαφινή το συνέδεσε με την ομάδα ad hoc, αλλά και ο κύριος Σμιτ ε, και πραγματικά Κατά την εκπόνηση του κειμένου αυτού αναγνωρίσαμε και διαπιστώσαμε ότι τα δύο κείμενα πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και μάλιστα συνδέονται μεταξύ τους οι δύο γνωμοδοτήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο καταλήξαμε σε αυτό. Η κυρία Ντεμελέν ε, είπε ότι θα πρέπει να απαντούμε στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Συμφωνώ απολύτως. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έρθει πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό τα λέμε ξεκάθαρα στην γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ και σας κυρία Μπαρμπούτσι για τα καλά σας λόγια και τα επενετικά. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε και ε, είπαν και πολλά μέλη της Επιτροπής 2 ε, ότι υπάρχουν τροπολογίες και πρέπει να επαναλάβω κάτι που είπα στην αρχή. Εμείς προσπαθήσαμε να εντάξουμε στο κείμενο όλα ε, τα σημεία στα οποία συμφωνήσαμε στις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής, ιδιαίτερα στην τελευταία. Ε, Χρειαστήκε να ε, απορρίψουμε κάποιες τροπολογίες για να παραμείνει σε ισορροπία το κείμενο και να σεβαστούμε και τις συζητήσεις. Κύριε Πετσίνη, βεβαίως συμφωνώ απολύτως. Το κείμενο θα αλλάξει και θα αλλάζει όσο προχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνώ ότι πολλοί πολίτες δεν καταλαβαίνουν ότι εκτός από την εσωτερική αγορά υπάρχουν και ωφέλη, μάλλον έχουμε μια πραγματικά εσωτερική αγορά και ωφέλη από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε λοιπόν το κείμενο αυτό να το θέσουμε στη διάθεση όσων θέλουν να τα διαβάσουν αυτά τα ωφέλη. Ο κύριος Σμιτ βεβαίως. Ε, κύριε Σμιτ, ε, σε σχέση με τα δύο εγγράφα πρέπει να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε. Λυπάμαι, πρέπει να σταματήσω. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ, Μιχαήλ Στεφάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Κύριε Ροκαρεύσκη, είναι προφανέ ότι χρειάζεται μια Ευρώπη με ανωδική πορεία. Δεν ικανοποιηθούμε με Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Όσον αφορά το ονομαστικό μισθό, δεν είναι πραγματικά ονομαστικό ε, μισθό που μετράει, ε, ε, η δυνατότητα αγορά, η αγοραστική δύναμη τι αγορές μπορεί να κάνει με έναν μισθό. Κυρία Σαλβίνη, για τη βιωσιμότητα και την αθεκτικότητα στο κείμενο βάλαμε αυτή την έννοια. Κυρία Ντεβέλεν, συμμερίζομαι την άποψή σας. Εν μέρη, αριθεύει ότι μετά το τέλος του συστήματος του κομμουνιστικού στην Ευρώπη θεωρήσαμε όταν το τέλος της όλης ιστορίας και επευλήθη ε, λίγο πολύ σε όλο το σύστημα, σε όλο τον κόσμο, μια ιδεολογία νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποιημένη. Αλλά εφαρμόστηκε όμως ε, ε, λησμονήθηκε το σύστημα. Λησμονήθηκαν κάποια στοιχεία, όπως είπα στην ομάδα εργασία. Υπάρχουν κενά γεωγραφικά και κοινωνικά. Και θα πρέπει να δώσω μεγάλη προσοχή, ε, διότι τα έχουμε αγνοήσει. Και γι' αυτό στη Γαλλία πληρώνεται το τίμημα τώρα. Κυρία Μπαρμπούτσι. υπάρχουν προβλήματα πράγματι. Αλλά τα κοινωνικά δικαιώματα ε, ε, υποθέτουν για να ισχύουν και μια ζωντανή ε, οικονομία. Δόκτωρα Πετίνη, οι πολίτες δεν έχουν το συνέστημα ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι. Οι πολίτες ζουν στη χώρα τους. Η Ιταλία στην Ιταλία, στην Ιταλία Γάλλη στη Γαλλία, η Γερμανία στη Γερμανία. Πρώτα αισθάνονται ότι ανήκουν εκεί που ζουν, όχι μόνο στο κράτος, στην περιφέρεια, στην περιοχή τους, στο χωριό τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε πώς είναι. Είναι είναι ας πούμε όπως όταν ανακαινίζουμε ένα κτίριο βάζοντας μπροστά όμορφα σχέδια. Αλλά αυτοί που ζουν μέσα πριν ανακαινιστεί το κτίριο ζουν ακόμα στα παλιά διαμερίσματα. Ε, λοιπόν, έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας, λέει το δικό μου σχέδιο. Σταματά λοιπόν, λέει ο κύριος Στεφάν. Πάμε λοιπόν στην εξέταση των διαφόρων τροπολογιών. Υπάρχει κατάλογος. Πολλά. Τροπολογία 10. Το, ε, γίνεται αποδεκτή, είναι κάποιος κατά. Όχι, ευχαριστώ. Τροπολογία 3 για το σημείο 5-5. Μουνοβίτς ακυρώνεται αυτό, αποσύρεται. Τροπολογία 12 για το σημείο 5-5. Άντερσον Μούλεβιτς απορρίπτεται. Ένας από τους ε, τρεις που υπέβαλαν την ε, τροπολογία μπορούσαν να κάνουν μια παρουσίαση. Ποιος, ο κύριος Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή η γνωμοδότηση που έχουμε μπροστά μας, όμως επίσης μια καλή γνωμοδότηση μπορεί να βελτιωθεί. Και νομίζω ότι όσον αφορά το κείμενο, αυτό το τμήμα για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, για κάποιο λόγο το ΦΠΑ, η απάτη του ΦΠΑ δεν, αναφέρεται και σίγουρα θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται. Αυτό στον αυτή η Επιτροπή έχει εκφράσει άποψη όσον αφορά το κενό του ΦΠΑ και την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ επανειλημμένα. Και ζητούσαμε ε, να ληφθούν μέτρα και πιέζαμε. Το κείμενο προτείνει σε ομοσπονδιακό επίπεδο κάποιους φόρους, κάποια τέλη. Αυτό δεν μας βρήκε συμφώνους και τα κράτη-μέλη δεν φαίνεται να μπορούν να προχωρήσουν καθόλου σε αυτό το τομέα. Είναι σημαντικό λοιπόν να συμπεριλάβουμε την απάτη του ΦΠΑ και σημειώνω ότι αυτή είναι γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της Ρουμανικής ε, Προεδρίας. Η Ρουμανία είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ανώσους με το υψηλότερο κενό ΦΠΑ. Δεν συλλέγεται το ΦΠΑ. Ευχαριστώ, Κρίστιαν. Δεν κάνουμε τη συζήτηση τώρα της ομάδας μελέτης. Ευχαριστώ. Οι συγητές... Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Άντερσον, συζητήσαμε αυτό στο τμήμα το οικονομικό και, το, και στην Επιτροπή το προωθήσαμε. Η πρότασή σας για αυτή την τροπολογία προσπαθεί να διαγράψει αυτά που έχουμε γράψει σε άλλη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ και γι' αυτό πρέπει να την απορρίψουμε. Αν δεν σφάλω, δεν έχω το κείμενο μπροστά μου, αλλά είμαι αρκετά σίγουρος ότι ήταν του, κυρίου Θρίας Πίντο η γνωμοδότηση. Προτείνεται να περικόψουμε κάτι από την προηγούμενη γνωμοδότηση, οπότε δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε. Εντάξει, άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est 76 υπέρ, 98 κατά, 16 αποχές. Απορρίπτεται η εν λόγω τροπολογία. Τροπολογία 11 για το σημείο 5-6. Φιλ Παρενσόν απορρίπτεται. Κύριε Πέλ και κυρία Παρενσόν, θέλετε να παρουσιάσετε την τροπολογία. Τζόναθαν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια καλή παράγραφος, η 5-6 λέει πολλά που πρέπει να υποθούν για τις παρούσες εμπορικές συμφωνίες, αλλά ξεπλάγει τα μάλα, διότι η αναφορά στην Ιαπωνία πιο συγκεκριμένα έπρεπε να είχε διαγραφεί αυτό το έγγραφο σε αρκετά, που διαγράφηκε σε αρκετά καστερημένο στάδιο. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσης Ιαπωνίας είναι ακρογωνίως λήθος είναι η πρώτη μεγάλη συμφωνία μεταξύ σημαντικών οικονομιών από την Ευρώπη και την Αποανατολή. Και νομίζω ότι θα πρέπει να την επενέσουμε και να την αναφέρουμε. Φαίνεται ότι ακολουθούμε διχασμένη προσέγγιση προ το εμπόριο. Είτε είναι καλό είτε κακό. Αν είναι κάτι καλό, τότε η συμφωνία από την Ιαπωνία ξεχωρίζει σαν μια ειδική συμφωνία και συνεπώ θα ήθελα να συμπεριλαμβάνεται αυτή η μηνύα στην Ιαπωνία ξανά. Οι συγκητέ. Ευχαριστώ κύριε Πίλ. Συζητήσαμε αυτό το θέμα στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής και ο κ. Γκράιφ προλίγου, πριν από μερικά λεπτά, είπε ότι δεν πιστεύει ότι οι εμπορικές συμφωνίες με Ιαπωνία και Καναδά είναι πλήρως επωφελείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε βλέπετε την απόκληση που υπάρχει. Συνέβη στην Επιτροπή μας και εφόσον δεν συμφωνήσαμε, δεν συμπεριλάβαμε αυτή τη μνήμα στο έγγραφο, προσπαθώντας να σεβαστούμε αυτό που επεξεργαστήκαμε από κοινού. Όπω κάναμε και με άλλε τροπολογίε, έπρεπε λοιπόν να την απορρίψουμε βάσει τελευταία συζητήσεω που είχαμε και κάποιε αντιρρήσει από κάποια μέλη τη υποεπιτροπή όσον αφορά τη συμπερίληψη του Καναδά και της Ιαπωνίας στο συγκεκριμένο σημείο. Ευχαριστώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 73 υπέρ, 111 κατά, 11 αποχές. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 2 για το σημείο 5-6 γίνεται δεκτή. Αυτή υπάρχει κάποιος εναντίον. Καλώς. Τροπολογία 5 για τους 6-2 και αυτή γίνεται δεκτή. Υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση. Καλώς. Τροπολογία 6 για το σημείο 6.3 απορρίπτεται. Α, υπάρχει συμβιβαστική. Ευχαριστώ. Παρουσιάστε τη συμβιβαστική παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συζητήσαμε με τον κύριο Ροκαλεύσκη το θέμα λίγο πριν. Πριν έρθουμε εδώ. Προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστική, διότι μου εξήγησε ότι είναι σημαντικότατο το να έχουμε συλλογικέ διαπραγματεύσει και το σεβασμό τη αυτονομία των κοινωνικών εταίρων να συμπεριλαμβάνονται αυτά. Θα σα διαβάσω λοιπόν τη φράση που προσθέτουμε σε αυτή την παράγραφο, που βασικά παραθέτει προηγούμενη γνωμοδότηση. Τελευταία φράση θα λέει: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τι συλλογικέ διαπραγματεύσει και να σέβεται την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Τελεία. Ε, συμφωνείτε εσείς που υποβάλλατε τις τροπολογίες με αυτή τη συμβαστική. Ρογκρέφσκι, πού είσαστε. Α, ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος εναντίον της συμβαστικής. Ευχαριστώ. Δεκτή. Τροπολογία 13, το σημείο 64. Γίνεται δεκτή. Υπάρχει κάποιος που είναι εναντίον. Α, δεν σε είδα, Ελένη, συγγνώμη. Στη συνεδρίαση της ομάδας μελέτης, την τελευταία, θεωρήσα ότι είχαμε συμφωνήσει με τον Κρίστα Σφέγκ στη γαλλική εκδοχή του κειμένου. Έκανα σύγκριση και με την Ιταλική. Δεν ξέρω τι λέει η αγγλική εκδοχή. Εν πάση περιπτώσει είναι σαφές ότι μιλάμε για κοινή ευθύνη και συμφέρον ε, και μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Λογικά θα έπρεπε να μιλάμε για κοινά συμφέροντα και όχι για ευθύνε κοινέ. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει μια επαλήθευση, ένας έλεγχος των κειμένων. Διότι στο γαλλικό κείμενο, στην εκδοχή που έχω, μπορούμε να κάνουμε ό,τι επαλήθευση θέλετε. Τώρα γίνεται, γίνεται η τροπολογία από τον συγκητή τις εκδοχές επιτάπητος. Δεν θα κάνω τώρα εξακρίβως και παλήθευση κειμένων. Είναι κοινά συμφέροντα και ευθύνε, λέει το κείμενο στα αγγλικά. Εάν μιλάμε για συμφέροντα και ευθύνε, εγώ είμαι αντίθετη και ζητώ ψηφοφορία. Ξεκάθαρο. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν τη συμβιβαστική. Ορίστε, ξεκινάει η ψηφοφορία. Καλώς, τελείωσε η ψηφοφορία μας. 103 υπέρ, 61 κατά, 20 αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 για το σημείο 6, 4. Απορρίπτεται. Ποιος θέλει να παρουσιάσει. Ποιος. Α, εσείς ορίστε. Σας ευχαριστώ z Κοιτάξτε, αναφέρεται εδώ στην τεχνητή νομοσύνη, αυτοματισμούς κλπ. Ε, θέλουμε να αναφέρουμε την ανάγκη για υπεύθυνε και βιώσιμες επενδύσεις σε ποιοτική εκπαίδευση. Είναι προϋπόθεση αυτή για την έρευνα και ανάπτυξη. Η τροπολογία λέει ότι θα έπρεπε να βελτιώσουμε τη διαβίω εκμάθηση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων για όλους τους Ευρωπαίους εργαζομένους. Είναι για κοινή ωφέλη. Αυτό που είναι σημαντικότατο, ο σκοπός της τεχνολογικής εξέλιξης θα πρέπει να είναι η βελτίωση της θέσης του ανθρώπου. Να δημιουργήσουμε καλύτερε συνθήκες εργασίας, διαβίωσης, καλύτερες θέσεις απασχόλησης, πιο ισότιμη κοινωνία και όχι το αντίστροφο. αυτό είναι κάτι που απασχολεί τους πολίτες. Πιστεύω ότι αυτή η τροπολογία ευθυγραμμίζεται με την γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, οι Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, όταν αναφέρει το πρώτο τμήμα της τροπολογίας ταχείες αλλαγές, που αυτό υπονοεί και μια βιώσιμη ανταπόκριση αυτό, δεν χρειάζεται προσθήκη, και εξυπακούεται αυτό. Μετά, στο τέλος, η φράση εξηγεί τη μετάβαση, την αλλαγή που αναφέραμε στο κείμενο και εγώ και οι συνεισηγητές πιστεύουμε ότι δεν ήταν απαραίτητο να προσθέσουμε συγκεκριμένη μνήμα επιπλέον. Συζητήσαμε το θέμα στην τελευταία συνεδρία του Επιτροπή και όπω κάναμε και με τι τροπολογίε για την ομάδα 1, θα πρέπει να είμαστε συνεπεί, να παραμείνουν συνεπεί και να απορρίψουν τροπολογία, διότι δεν καταλήξαμε πάνω σε αυτό σε συμφωνία στην τελευταία συνεδρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Τέλος is Τέλος ψηφοφορίας. 449 κατά, 78 υπέρ, μάλλον 300, πρώτο ήταν υπέρ, το δεύτερο κατά, εγκρίνεται η τροπολογία. Η Κρίστα ζήτησε το λόγο για ένα διαδικαστικό. Ε, λυπάμαι, συγγνώμη που δημιουργώ μια σύγχυση, αλλά Μόλις ψηφίσαμε την 6.4, τη δική μου τροπολογία και τώρα φαίνεται το ίδιο ψηφίζουμε με άλλη, για άλλη τροπολογία. Ενώ η δική μου έχει εγκριθεί και τώρα για την ίδια παράγραφο έχουμε δύο διαφορετικές ε, τροπολογίες. Ποια είναι η σωστή τελικά, γιατί ψηφίσαμε για την ίδια παράγραφο δύο διαφορετικές τροπολογίες. Ποια ισχύει. Οι υπηρεσίε μου λένε ότι δεν είναι αντιφατικές μεταξύ τους οι δύο τροπολογίες. Δεν είναι η μία η άλλη, είναι ελοσυμπληρώμενες. Οπότε, αν ευσταθεί φυσικά η ενημέρωση που μου έκαναν οι υπηρεσίες, ότι δεν είναι αντιφατικές μεταξύ τους οι τροπολογίες. one part of... Είναι ένα τμήμα της τροπολογίας μόνο που ε, είναι αντιφατικό με τη δεύτερη τροπολογία. Αλλά η Ολομέλη τελικά υπερψήφισε και τις δύο, οπότε δεν, έχουμε να, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα πια για να το αλλάξουμε. Διαδικαστικό. Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι για να κάνουμε σωστά το έργο μας είτε θα πρέπει να διακόψουμε κάτι που είναι δύσκολο ή να επανέλθουμε στην γνωμοδότηση αυτή αύριο το πρωί για να μπορέσουν οι συντάκτες των τροπολογιών και οι συγητές να καταλήξουν μια ενιαία τροπολογία. Είναι νομίζω άσκοπο να συνεχίσουμε την ψηφοφορία για την γνωμοδότηση αυτή όταν έχουν δημιουργηθεί κάποιες ασυνέπειες, ασυναρτησίες και αντιφατικά σημεία. Ναι, πολύ εύστοχη η πρότασή σας. Και προτείνω το εξή Να αφήσουμε εκρεμές αυτό το θέμα και για το σημείο 6.4 που έχουμε δύο εν μέρει αντιφατικές τροπολογίες μεταξύ τους να το αφήσουμε. Θα συμπληρώσουμε τώρα την ψηφοφορία με τις υπόλοιπες τροπολογίες αλλά την ανάλυση για το 6.4 ε, θα την κάνουμε σε μία ώρα, μέσα σε μία ώρα. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε για αύριο, έχουμε άλλε και πολλέ γνωμοδοτήσει. Μέσα σε μία ώρα θα πρέπει να βρεθεί μία λύση ώστε να καταλήξουμε σε μία ισορροπημένη και συνεκτική διατύπωση για το 6-4. Διαφωνεί κανεί, Όχι. Οπότε, η τελική διατύπωση του σημείου 6-4 ε, θα οριστικοποιηθεί σε λίγο, γιατί διαπιστώθηκε αντίφαση μεταξύ δύο τροπολογιών. Οπότε, μέσα σε μία ώρα θα συνεννοηθούν οι συντάκτε με του συζητητέ για να υποβάλουν ένα κείμενο στην Ολομέλεια αργότερα για να το ψηφίζουμε. Πάμε στο 6-6 που έχει αποσυρθεί. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ρογκαλεύσκη να μα παρουσιάσει την τροπολογία του. Η τροπολογία αυτή ουσιαστικά ε, είναι μια παράθεση του 6-6 γιατί το 6-6 είναι πιστή αντιγραφή της ε, ε, τροπολογίας 564 για, το, για την κοινωνική διάσταση και τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, την έκθεση της Γκάβι Μπίσοπ και Γιούκα Άτελα. Ουσιαστικά αντιγράφουμε πιστά ένα σημείο στην 6-6. Οπότε, από τη στιγμή που έχουμε μία μνήα ή αναφορά, καλό θα ήταν να είναι πιστή αυτή η αναφορά μία πραγματική παράθεση και όχι στο περίπου χονδρικά. Βέβαια εδώ δεν έχουμε την, αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, το μόνο που έλειπτε από την παράθεση. Γι' αυτό την καταθέσαμε και τη σχετική τροπολογία. Το ίδιο είχαμε και στο σημείο 12 που είπε ο εισηγητή ότι θα πρέπει όταν κάνουμε μια παράθεση να είναι πλήρη. Και γι' αυτό ακριβώ ε, κατέθεσα τη σχετική τροπολογία για να συμπληρώσω την μερική παράθεση που είχε γίνει προηγούμενης γνωμοδότησης που είχε ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή. Ήταν γνωμοδότηση συναδέρφων των ομάδων 1 και 2. Ευχαριστώ. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου αυτή, ε, αυτής δεν παραθέτει παράγραφο από άλλη γνωμοδότηση. Και το μικρότημα που όντως περιλαμβάνει παράθεση ήταν πιστό. Και η τροπολογία είναι κάπως αφήσιμη. Ε, ε, γιατί λέει θεσπίζει ή ζητά. Και αυτό ήταν κάπως αόριστο. Και το συζητήσαμε στην τελευταία συνεδρίαση υποεπιτροπής και υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις, ιδιαίτερα από μέλη της ομάδας 1. Δεν μπορούμε λοιπόν εγώ και ο συνεισηγητή μου να γνωρίσουμε τι συζητήσει τη Υποεπιτροπή και από τη στιγμή που δεν ε, επετεύχθη συμφωνία, εκτό ε, από τη συμφωνία για το τμήμα που αναφέρουμε, δηλαδή για να ε, εξασφαλίσουμε να αλλάξει το εισόδημα, να κατώτατο το εισόδημα για του Ευρωπαίου πολίτε, αυτό το συμπεριλάβαμε. Και αυτό το συμπεριλάβαμε ω συμβαστική λύση μετά τη συζήτηση που είχαμε στην Υποεπιτροπή. Γι' αυτό και πρότεινα να απορριφθεί η τροπολογία 6-6. Καλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 497 υπέρ, 77 κατά, 18 αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία. Πάμε στην τροπολογία 9 που προτείνει την προσθήκη ενός νέου σημείου. Οι εισηγητές είναι κατά. Οπότε θα ζητήσω και πάλι από τον συντάκτη, τον κύριο Ρογκαλεύσκη, να μας την εξηγήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι έχουμε εδώ μια τροπολογία που αντικατοπτρίζει τη συζήτηση που είχαμε στην υποεπιτροπή για την κινητικότητα και την διαρροή εγκεφάλων. Θέλουμε να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας και μάλιστα ανταποκρίνεται σε προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Επαναλαμβάνω πολύ συχνά όταν έχουμε μία των κοινωνικών εταίρων είπαμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να μιλούμε για τη δίκαιη κινητικότητα και να πώς αποτρέψουμε τη διαρροή εγκεφάλων και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Γιατί είναι πραγματικότητα η διαρροή εγκεφάλων. από την Πολωνία έχουμε έξοδο γιατρών, νοσοκόμων, νοσηλευτικού προσωπικού ε, και τα νοσοκομεία μας ε, αντιμετωπίζουν πολλές ελλείψεις λόγω αυτής της ε, εξόδου της μαζικής εργαζομένων στον ιατρικό κλάδο. Στο 1-9 μιλούμε για την αγορά εργασίας. Μάλιστα όπως προβλέπουν και οι συστάσεις και τα συμπεράσματα. Και επίσης λέμε ότι θα πρέπει να προσφέρουμε τα εφόδια στους πολίτες ώστε να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές αλλαγές. Μιλούμε για τη σημασία που έχει το, η κατάρτιση, η επιμόρφωση, η αναβάθμιση των προσόντων, τα προγράμματα διαβίου κατάρτισης και τα θέματα εις ευκαιρίες και δίκαιης κινητικότητας. Τα λέμε σε πολλά σημεία. 1, 6, 2, 13, 4, και ούτω καθεξής. Οπότε οι σχετικές πληροφορίες ήδη περιλαμβάνονται κατά τη γνώμη μας στο κείμενο της γνωμοδότησης. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε κάτι που ήδη αναφέρουμε στο κείμενο. Και γι' αυτό προτείνουμε να απορριφθεί η τροπολογία σας 1-12. Καλώς άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο Τέλος 103 υπέρ, 490 κατά και 6 αποχές εγκρίνεται. Πάμε στα 1-5 Προτείνεται διαγραφή του κειμένου. Έχει γίνει δεκτή από τους συγγητές. Ε, κατά κανείς. Όχι και ένα 12 Μα είναι ίδια με την εννέα. Απλώς διορθώνει τα συμπεράσματα και τις στάσεις με βάση προηγούμενη τροπολογία που έχουμε εγκρίνει. Για να είμαστε συνεπείς. Από τη στιγμή που έχουμε, την έχουμε ήδη την προηγούμενη τροπολογία πρέπει να την ευθυγραμμίσουμε. Δέχονται οι συγγητές. Είναι κανείς κατά. Ωραία. Τελική ψηφοφορία αργότερα, γιατί εκκρεμεί ένα σημείο, το 6-4. Πριν τις 7 παρακαλώ να μας υποβάλλετε την οριστική διατύπωση για το 6-4. Παρακαλώ τον εισηγητή και τη γραμματεία να διαθετήσουν αυτή την σύγκρουση των διατυπώσεων αν όντως υπάρχει τέτοια σύγκρουση και αντίφαση. Πάμε στο 1687 σχέδιο δράσης ε, κατά της παραπληροφόρησης Ούλριχ Σάμ και Τζούλια Μπαρμπούτσι. Grazie. Danke. Es geht um Desinformation. Πρόκειται για την παραπληροφόρηση. Παραπληροφόρηση, κοιτάξτε, υπάρχει από τότε που έχουν αρχίσει οι άνθρωποι να επικοινωνούν μεταξύ τους. Από τότε βεβαίως επίσης που επινοήθηκε η τυπογραφία και άρχισε τότε να κυκλοφορεί επίση παραπληροφόρηση και τώρα βέβαια με τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας έχουμε φτάσει σε άλλες διαστάσεις, διότι εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν την ίδια ακριβώς στιγμή, την ίδια είδηση μέσα στα ε, κοινωνικά μέσα και μπορεί έτσι να πολλαπλασιαστεί η πληροφορία, είναι δυνατόν να γίνουν εκστρατείες παραπληροφόρησης που να επηρεάζουν ολόκληρες κοινωνίες και μάλιστα μπορούν να σημάνουν και κίνδυνο για επικείμενες εκλογές. Είναι λογικό λοιπόν και συνεπές που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο προβλέπουν τώρα μια σχεδιαζόμενη δράση και κυρίω λόγω των ευρωεκλογών. Νομίζω ότι είναι κάπω καθυστερημένα, ελπίζω να μην είναι υπερβολικά αργά, ώστε με συντονισμένο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι στην παραπληροφόρηση. Πρόκειται για σχέδιο δράσεων που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Αφενός τον συντονισμό των διαφόρων αναγκαίων μέτρων σε όλες τις χώρες, σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις περιφέρειες, συντονισμό λοιπόν λέω, στο ευρωπαϊκό επίπεδο όλων αυτών. Δεύτερο, τα υφιστάμενα όργανα, εδώ της Ένωσης δηλαδή, τα οποία παρατηρούν συστηματικά την παραπληροφόρηση, την καταγράφουν και ενημερώνουν τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά τα όργανα εργάζονται θαυμάσια. Είναι όμως πολύ μικρά και οι δυνατότητέ τους περιορισμένες. Τρίτο λοιπόν η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, με την έννοια να ασκηθεί πίεση στις μεγάλες πλατφόρμες όπως Google ή Facebook ώστε να αναγκαστούν οι μεγάλες αυτές πλατφόρμες να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, για παράδειγμα με κώδικα συμπεριφοράς. Και τέταρτο, ευαισθητοποίηση των κοινωνιών. Δηλαδή, να διατίθεται σωστές πληροφορίες, ποιοτική δημοσιογραφία από όλες τις ε, διαθέσιμες πηγές. Εδώ ρόλο καλείται να παίξει και η κοινωνία των πολιτών και επομένως και η δική μας επιτροπή. Τώρα στο τμήμα μας και ιδίω στην ομάδα μελέτης συζητήσαμε πολύ και διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ιδιαίτερα το ρόλο τη ρωσική κοινοπολιτεία. Εξετάζοντα κάπω επιφανειακά, θα μπορούσε να θεωρήσει κανεί ότι πρόκειται μονάχα για τη Ρωσία. Συζητήσαμε όμω το τμήμα μα και κατέστη σαφέ από τι συζητήσει αυτέ ότι δεν είναι μόνο η Ρωσία. Υπάρχουν και πολλέ άλλε πηγέ παραπληροφόρηση. Και γι' αυτό καταθέσαμε και σχετική τροπολογία, όπου καθιστούμε σαφέ ότι υπάρχουν ποικίλοι κίνδυνοι από ποικίλε πηγέ. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να προκληθεί εντύπωση που είπα προηγουμένως και γι' αυτό θα παρακαλέσω τώρα δά που θα ψηφίσουμε την έκθεση να μην εξετάσετε αν έχουμε γράψει υπερβολικά πολλά, υπερβολικά λίγα για τη Ρωσία. Πρόκειται για κάτι άλλο. Κυρίως μας ενδιαφέρει δομικά, διαρθρωτικά να ενισχυθεί ξεπεράσατε το χρόνο σας λέει ο πρόεδρος Πολύ κακό γερμανικό στυλ αυτό. Η Τζούλια Μπαρμπούτσι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, να πω το εξής εγώ. Αυτό το σχέδιο δράσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή την ιστορική στιγμή. Γιατί έχει στόχο την προστασία των δημοκρατιών μας και να σταματήσει τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που οδηγούν στην καχυποψία, στην, στο διχασμό και στους θεσμούς και στην πολιτική. Και αυτές οι ψευδείς ειδήσει πολύ συχνά παράγονται από πολιτικές δυνάμεις εθνικιστικές που επίθενται κατά της Ευρώπης και διαδίδουν φόβο, αβεβαιότητα στους πολίτες. Έχουν συγκεκριμένο πολιτικό στόχο. Αυτό είναι ο βασικός λόγος, κατά την άποψή μου, για τον οποίο αυτή η γνωμοδότηση θα πρέπει να ψηφιστεί να υπερψηφιστεί. Προφανώς πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια συντονισμένη δράση για την προστασία της ενώσεως και των θεσμών της και των πολιτών κρατά της παραπληροφόρησης. Και αυτό σίγουρα πρέπει να υποστηριχθεί. Πιστεύουμε όμως ότι και αυτό θα πρέπει να γίνει γρήγορα, διότι οι ευρωεκλογέ επίκυνται. Οπότε, όπως έλεγε ο συνάδελφος, Ελπίζουμε αυτό το σχέδιο δράσης να έχει αποτέλεσμα και αντίκτυπο ε, στις επόμενες ευρωεκλογέ. Είχαμε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα να εργαστούμε. Χρειάστηκε μεγάλη συνεργασία, πολλή συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας μελέτης. Θέλω να υπογραμμίσω εντάχει το εξής, ότι στο κείμενο υπάρχει σαφής αναφορά στην ε, εμπλοκή των ενδιαφερομένων φορέων και των διαφόρων φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει και αναφορά στη θετική προσπάθεια που να κάνει η ομάδα επικοινωνίας της ΕΟΚΕ, διότι μας απασχολεί πολύ αυτό το θέμα και έχουμε ειδική υπηρεσία που μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα, λίγο αργά άνοιξε με τον κατάλογο των ομιλητών. Ολοκληρώνω το κατάλογο. Στιερή Λιμπέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που επιτέλου η Ευρώπη συνειδητοποίησε το πρόβλημα των φαλκιδευμένων ειδήσεων, των fake news και των ολέθριων συνέπειών του στη δημοκρατία και τις εκλογικές διαδικασίες. Και φυσικά έχουμε κατά νου τι ε, επικείμενε ευρωεκλογέ. Η γνωμοδότηση που θα ψηφίσουμε σήμερα και στην οποία συμμετείχα για την εκπόνησή της στην ομάδα εργασίας σίγουρα ακολουθεί πολύ σωστή άγουσα. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή έχει συντάξει μια πολύ άρτια έκθεση. Στις 13 Μαρτίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απεφάνθη σχετικά και χθε 19 σημαντικά ευρωπαϊκά ΜΜΕ συσπηρώθηκαν, συγκέντρωσαν τις προσπάθειές τους και τους πόρους τους για να αντισταθούν και να καταρρύψουν τα fake news, τις ψευδείς ειδήσει. Οπότε πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη σύσσωμη σε αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς ακόμη δεν αναδεικνύουμε αρκετά τα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη που έχουν πολλές αρμοδιότητες στα θέματα της κοινωνικής ψυχολογίας, της μελέτης, της φημολογίας, της επιστήμης, της επικοινωνίας, της κοινωνιολογίας. Και επειδή ήμουν και εγώ διευθυντή ενό ερευνητικού κέντρου, σα διαβεβαιώ ότι υπάρχει ένα χρυσορυχείο γνώσεων και ικανοτήτων που μπορούμε και εμεί να αξιοποιήσουμε στον αγώνα αυτό κατά των ψευδών ειδήσεων. Επίση, έχω κάποιες παρατηρήσεις. Έχουμε 5.000 ε, περιπτώσεις παραπληροφόρησης που εντοπίστηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην ε, Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Έχουμε ουσιαστικά ένα πόλεμο της ε, πληροφόρησης και δεν μπορούμε μόνο με άμυνα να κερδίσουμε ένα πόλεμο. Δεύτερον, δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις συνέπειες και να τις αντιμετωπίσουμε αν δεν εξετάσουμε και δεν καταπολεμήσουμε τις αιτίε. Γιατί αυτές οι ψευδείς ειδήσει, τα, fake news δεν αναπτύσσονται τυχαία. πρέπει να βρουν γόνιμο έδαφος για να ευδοκιμήσουν. Ε, δυστυχώς ε, ε, έχετε υπερβεί το χρόνο σας και κατά 15 δευτερόλεπτα μάλιστα. Λούση Στρουντνίτσα. Έχουμε 5-6 ακόμη γνωμοδοτήσεις. 7. Οπότε πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο αγόρευση γιατί θα το στερήσουμε ιδέα από του συναδέλφου. Δύο λεπτά. Λούση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζομαι καν δύο λεπτά. Θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω του συνεισηγητές ε, για την άρτιά του γνωμοδότηση και να επαναλάβω κάτι που ήδη είπε η Τζούλια. Εδώ δεν μα ενδιαφέρουν μόνο οι επικείμενε ευρωεκλογέ Έχουμε πολλές άλλες εκλογικές διαδικασίες που έγιναν ή θα γίνουν στο μέλλον. Και τα fake news, αυτές οι ψευδείς ειδήσεις είναι απειλή για όλες τις εκλογές. Γιατί πλησιάζουμε και στο Brexit και κανείς δεν αφιβάλλει πια ότι και το Brexit σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε από τα fake news, από αυτές τις ψευδείς ειδήσεις. Και ίσως η έκβαση του δημοψηφίσματος επηρεάστηκε πολύ. Επίσης, δεν υπάρχει αρκετός ψηφιακός αλφαβητισμός θα πρέπει η ψηφιακή εκπαίδευση να προσφέρεται από την σχολική ηλικία. Και δυστυχώς συστερούμε σε σχέση με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα και που δυστυχώς ευνοούν την εξάπλωση των ψευδών ειδήσεων. Και το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Και φυσικά είναι ε, προσωπικό και ατομικό θέμα, αλλά έχουμε και διαδικασίες και κανονισμούς που πρέπει να ρυθμίσουν το φαινόμενο αυτό. Είμαι υπέρ της γραμμοδότης και ευχαριστώ τους συνεισηγητές. Μάρκο Βεσάνη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξετίμησα πολύ αυτή τη γνωμοδότηση. Θεωρώ ότι είναι πολύ ισορροπημένη και θαραλέα. Ταυτόχρονα. Ευχαριστώ τον Ούλρικ και την Τζούλια. Εξετίμησα ιδιαίτερα κάποιες έννοιες που διευκρινίστηκαν άριστα, όπως η άνση κατάχρησης ελευθερίας της έκφρασης, η διεύρυνση της ενίας των ψευδών ειδήσεων, των fake news και η πρόσκληση να μην βασιζόμαστε μόνο επιθυλοντικών οικειοθελών δράσεων για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων. Όσον αφορά τη Ρωσία, δεν έχω τίποτα κατά της Ρωσίας. Όμως σήμερα πιστεύω ότι είναι αντικειμενικό, κανείς δεν παντηρηθεί ότι αυτή η χώρα βασίζεται στον πόλεμο της παραπληροφόρησης. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες απειλές, καλά τα είπε ο Ούλρικ, αλλά πιο ε, επικίνδυνη η κατάσταση φορά τη Ρωσία. Για να την Ιταλία, σήμερα υπάρχουν ε, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και ιστοσελίδες διαδικτύου ε, που είναι στα χέρια Ρώσων που διαδίδουν εμφανώς και συνεχώς ψευδείς ειδήσει που επηρεάζουν την πολιτική μας ζωή και η Λέγκα του Σαλβίνη, το κόμμα που σύμφωνα με τι δημοσκοπήσεις θα έχει περισσότερε περισσότερες στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε επαφές με το κράτος, με το ρωσικό κράτος, ε, επιδιώκοντα χρηματοδότηση. Όπως αυτό τεκμηριώθηκε πριν από 15 μέρε από το Εσπρέσο και κανένας ούτε η ίδια η Λέγκα δεν το διέψευσε αυτό. Λοιπόν, πολύ καλά τα έκαναν ο Ούλρικ και η Τζούλια, επέτυχαν ισορροπημένο κείμενο, είναι σαφή, πιστεύω όμω ότι όχι όλες οι απειλές είναι ίσες, άρα χρειάζεται να το πούμε αυτό και να μην φοβόμαστε να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των μεν και των δε. Ευχαριστώ Μάρκο. Κβανταράιτε για δύο λεπτά. Buvau šios studijų grupės narė. tikrųjų. Εγώ ήμουν μέλος της Επιτροπής Μελέτης, της ομάδος μελέτη. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ βεβαίως και τους ε, δύο εισηγητάς. Έχω να πω ότι ήταν πολύ ε, ενδιαφέρον συζητήσει στην ε, ομάδα μελέτης και νομίζω ότι ήταν και αντικειμενικές. Καθώς συζητούσαμε δηλαδή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. δεν συζητήσαμε μόνο απειλές που προέρχονται από μια χώρα. Τονίσαμε την ανάγκη ε, σεβασμού της ελευθερίας έκφρασης. Και επίσης είπαμε ότι αυτή η νοοτροπία της δυσφήμισης και ε, των επιθέσεων, ε, φραστικών επιθέσεων πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να προστατεύσουμε τις αξίες, πρέπει ωστόσο να μιλήσουμε και για τη σημασία της παιδείας. Να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας και βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε και τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και αυτούς που ζουν σε τρίτες ε, ε, χώρες και εννοώ ιδίως εδώ τις χώρες της ανατολικής γειτονίας καθώς και άλλες χώρες οι οποίες βέβαια συνεργάζονται μαζί μας σε κοινά έργα. Ευχαριστώ. Πάβελ Τρακίνα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση να μπορέσω να συνεργαστώ με τους δύο μεσήνες ως πρόεδρος της ομάδος ε, μελέτης. Ε, διαπνέονταν από συνενετικό πνεύμα οι συζητήσεις μας και νομίζω καταλήξαμε στην βέλτιστη δυνατή ισορροπία. Μια ισορροπία που συνεχίζει το έργο μας του περσινού χρόνου όταν είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φανεί πλέον φιλόδοξη και πράγματι φάνηκε πλέον φιλόδοξη. Και για το λόγο αυτό βεβαίως εμείς ε, συμφωνούμε με την ε, πλειονότητα των προτάσεων. Ας μην υπάρχει αμφιβολία, όπως είπαν και άλλοι συναδελφοί μου προηγουμένως, ότι η διάδοση της παραπληροφόρησης είναι ένα είδος υβριδική διεξαγωγής πολέμου, με ξεκάθαρους στόχους ωστόσο. πολλέ από τι παραπληροφορήσει αυτές προέρχονται από την επικράτεια τη ε, ε, ρωσική κοινοπολιτεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, έχει επιβεβαιωθεί. Υβριδικό πόλεμο λοιπόν, ο οποίο χρησιμοποιεί την παραπληροφόρηση καθώ και χρηματοδότηση εξτρεμιστικών δυνάμεων σε όλε τι χώρε μέλη τη Ένωση. Όπω είπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προεβδομάδο, ακριβώ στην παρούσα αίθουσα. Οι βουλευτέ μάλιστα τάχθηκαν υπέρ των ίδιων πραγμάτων που λέμε και εμεί εδώ δηλαδή ενίσχυση χρηματοδότηση μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση τη προσπάθεια, της ε, αυτής. Γι' αυτό και πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μα, διότι πρόκειται για ε, ολόκληρε στρατιέ τρόλ από την ε, Ρώσικη Κοινοπολιτεία, οι οποίοι υποσκάπτουν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού καθημερινά. Είμαι λοιπόν αντίθετο και με τι τροπολογίε του κ. Παυλίκα. Τέλο. Λίνα Σαουζιάκα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Χωρίς αμφιβολία πρέπει να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να υπάρξει μια συντονισμένη αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης γιατί μεμονωμένες δράσεις δεν αποδίδουν όπως σωστά λέχθηκε ήδη. Με τις ευρωεκλογές που έρχονται έχουμε αντιληφθεί ποιο είναι το μέγεθο του διακυβεύματο και μάλιστα έχει αναφερθεί ονομαστικά μία χώρα. Την, είπαν, ε, την ανέφεραν πολλοί συναδελφοί μου προηγουμένω. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Μιλώ και εγώ για τη ρωσική κοινοπολιτεία. Και στη βάση των δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουμε μετρήσιμε απειλέ που προέρχονται από την χώρα αυτή. Δεν θα πρέπει να διστάζουμε να αναφέρουμε την ε, Ρωσία με το όνομα της. Και πρέπει να τοποθετηθούμε καθαρά γιατί και η δική μας Επιτροπή πρέπει να έχει ξεκάθαρες θέσεις και κάτι άλλο που λέχθηκε ήδη προηγουμένως. Χρειαζόμαστε κριτική αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας παραπληροφόρησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά τώρα καθίσει εκ των εισηγητών για να απαντήσει. Ούλριχ, ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που εκδηλώσατε δια των λόγων σας. Επαναλαμβάνω ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται καθυστερημένα. Εμείς θα θέλαμε να είχε αρχίσει νωρίτερα και μάλιστα και πριν από τον Brexit. Αλλά τώρα πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες μας. Η έρευνα είναι σημαντική για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η παραπληροφόρηση γιατί υπάρχουν χώρες που είναι πιο ευαίσθητες από άλλες και ε, πώς κυκλοφορούν οι ειδήσει αυτές. Είναι σημαντικό πάντως να έχουμε ταχύτατη, ταχύτατο έλεγχο των γεγονότων, fact-checking δηλαδή, και η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πραγματικά καλή και να κοιτάξετε και τις υπόλοιπες. Έμαθα στην παρούσα Επιτροπή και εξεπλάγει από τις πληροφορίε που είδα στις εκθέσεις των συναδέλφων μας. Πρόκειται για την καταπολέμηση των λεγόμενων fake news και ιδίω το τμήμα τύπου, το δικό μας τμήμα τύπου δηλαδή, κάνει σημαντική προσπάθεια και νομίζω μάλιστα και ωφελεί και όλον τον τύπο. Σας ευχαριστώ. Η Τζούλια. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω εκείνους που παρενέβησαν διότι πραγματικά αξιολόγησαν θετικά τις προσπάθειές μας. Και εδράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της ομάδας, τον Πάβελ, με τον οποίο συνεργαστήκαμε πραγματικά άριστα. Καθώς και τη γραμματεία θέλω να ευχαριστήσω. Θα έλεγα ότι δεν έχω πολλά να προσθέσω στα είδη υποθέντα από τον Ούλριχ. Να πω μόνο ότι, παραδείγματος χάρη όπως έλεγα, τρία είναι τα θεμελιώδη σημεία. Συνοψίζοντάς τα. Αυτό που ανέφερα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών και τη συμμετοχή της ΕΟΚΕ. Δεύτερον, κάτι που ήδη αναφέρθηκε, δηλαδή ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το ζήτημα αυτό και να δούμε πώς μπορούν να αναπτύξουν κριτική σκέψη μέσω της παιδείας και άμεσης ενημέρωσης για τα ΜΜΕ. Θα πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο, από το δημοτικό πρέπει να ξεκινήσει αυτή η παιδεία και πρέπει να είναι μια παιδεία που να διαρκεί για όλη τη ζωή διότι προφανώς δεν πέρα τούτε μόνο στα θρανία του σχολείου. Και τέλος να πω και κάτι εντάχει για την προσπάθεια, την οικειοθελή, την εθελοντική που έχουν κάνει κάποιες πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κάποιες εταιρείε ε, διαφήμισης που είναι κάτι θετικό. Αλλά στην γνωμοδότηση λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν θεωρήσει ότι αυτή η προσπάθεια δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες, θα πρέπει, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δράσει με πιο συγκεκριμένες και περιοριστικές απαιτήσει. δεσμευτικές, μέσω ρυθμιστικών δράσεων που θα είναι ε, ισχυρότερες. Ευχαριστώ. Πάμε στις τρεις τροπολογίες. Υπαριθμών 3. Παυλίκας και για να απορριφθεί όλο το κείμενο. Ανδρέας, θες να παρουσιάσεις την ε, τροπολογία σου. Η τροπολογία 3, απορρίπτεται από ό,τι ξέρουμε. Εκτός αν άλλαξες γνώμη, ε. Ωραία. Ανδρέας. Αποσύρω την ε, τροπολογία Ανδρέα το σημείο 2.6. Αυτή τη στιγμή έχει ε, υπάρχει ε, συμβιβασμός για τις άλλες δύο μου τροπολογίες. Αποσύρετε την τροπολογία. Okay, thank you. Καλώς, σας ευχαριστώ. Τροπολογία 2 για το σημείο 4-3. Υπάρχει πρόταση συμβιβαστική οι εισηγητές παρακαλώ μπορούν να παρουσιάσουν τη συμβιβαστική. Η συμβιβαστική τροπολογία αναφέρεται σε ποιον αριθμό ήταν, για πέστε μου. Α, βλέπετε το κείμενο στην οθόνη. Λοιπόν, το σημείο 1-3 και το 3 κάτι. Τροπολογία 2, συνάδελφοι, για το σημείο 4-3, λέει ο πρόεδρος. Είναι ταυτόσιμες. Αλλάζει το κείμενο που αναφέρεται στη Ρωσική Ομοσπονδία και προσθέτονται και άλλες πηγές παραπληροφόρησης. Μπορείτε αυτό να το διαβάσετε. Όλοι μπορούν να το διαβάσουν στην οθόνη. Διευρύνεται λοιπόν ο κατάλογος πηγών παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων και εξισορροπείται η προσέγγιση του κειμένου στο πνεύμα που ανέφερε ο συνάδελφος. Παρ' όλα αυτά, αναφέρει επίσης ότι υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία στον αφορά τις πληροφορίες που έχουμε. Η Ευρωπαϊκή Task Force έχει πολλές πληροφορίες για εκστατείες παραπληροφόρησης. Σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν στη διάθεσή τους. Καλό θα είναι να διευρυνθεί το πεδίο και να δούμε και άλλε εκστρατείε παραπληροφόρηση. Για την ώρα δεν διαθέτουμε τι κατάλληλε πληροφορίε και δεν έχουν οι πληροφορίε που διαθέτουμε την ίδια ποιότητα που έχουν πληροφορίε περί Ρωσία. Στο τέλο, παροτείνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ληφθούν αντίμετρα σύμφωνα κλπ. κλπ. Αυτό αναφέρουμε. Και αυτή η διατύπωση αντικατοπτρίζει αυτές τις διάφορες απόψεις που υπάρχουν. Αντρέα, συμφωνείς με τη συμβιβαστική. Συμφωνώ, την αποδέχομαι. Okay, Καλώς, υπάρχει κάποιος που είναι εναντίον. Δεκτή τροπολογία 1 για το σημείο 1-3. Συνδέεται με τις άλλες, έτσι. Δεν υπάρχει ανάγκη να ψηφίσουμε. Δεκτήκαμε την πρώτη συμβαστική και η ίδια συμβαστική ισχύει και για αυτήν. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να πάμε στην τελική ψηφοφορία για τη 10 687 σχέδιο δράσης για παραπληροφόρηση ως ετροποποίηθη. Και άρχεται η ψηφοφορία. The vote Πέρας ψηφοφορίας. 142 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στους εισηγητές λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα. Το White Dove Way, ο δρόμος του Λευκού Περιστεριού, μια πρόταση για μια παγκόσμια στρατηγική, Παγίου ειρήνης, γνωμοδότης πρωτοβουλίας. Jane, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Είναι τέλος μιας μεγάλης ημέρας. Δεν φτάσαμε ακόμα στο τέλος, βέβαια. Ο καλύτερος τρόπος να περιγράφει την κατάσταση είναι ότι υποφέρω από τη στενοχώρια του Brexit, του Brexit, το Brexit Blues. Δείξτε υπομονή λοιπόν. Απεγνωσμένα πρέπει να, να, να βελτιώσω κάπως τα, την ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι η πρόθεση και του White Dove Way. Ξεκινώντας να εξηγήσω περί τίνος πρόκειται ο δρόμος του Λευκού Περιστεριού. Λογοπαίγνιο είναι. Είναι κάτι παραπάνω από ένα μονοπάτι ειρήνης. Είναι ένας τρόπος ζωής τρόπος εκμάθησης, τρόπος του να ηγείται κανείς, να ηγηθεί, να οδηγήσουμε την Ευρώπη και τον κόσμο μακριά από την τρέλα της ε, διέρεσης που έχει κατακλείσει τις κοινωνίες μας κατά το παρελθόν και μας απειλεί και τώρα. Σαν το μεγαλύτερο έργο, το μεγαλύτερο εγχείρημα ειρήνης στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί την εμπειρία αυτή και να γίνει προασπιστή τη αποφυγή των συγκρούσεων στο μέλλον, προθώντα την αρχή τη ειρήνη, ανοχή, το μηδέο σεβασμού, τη κατανόηση. Λοιπόν, βάσει αυτών ιδρύθηκε εξάλλου. Και ανησυχία υπάρχει ότι έχασε το δρόμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει σίγουρα πολύ σοβαρά υπαρξιακά προβλήματα. Και να μην πούμε ότι βασικά φταίει και το Brexit γι' αυτό, αλλά δεν χάθηκαν τα πάντα. Χρειάζεται ηγεσία, σαφή κατεύθυνση, σαφήνεια κλπ και να συμμετέχουν και οι πολίτες στην προσπάθεια. Ο Πρόεδρος το ονόμασε μια αναγέννηση. Αυτό χρειαζόμαστε, μια αναγέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε όμως και κάποιον που να μας ε, καθοδηγεί, κάτι να μας καθοδηγεί. Εδώ το White Dove Way είναι ένας οδικός χάρτης για ένα ταξίδι στο οποίο θα συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα τους δώσουμε μια, ένα συνέστημα ότι ανήκουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, ανοίγοντα ένα καινούριο δρόμο βάση της αποστολής που είναι η ειρήνη. Το μονοπάτι ξεκίνησε στη Βόρεια Ιρλανδία και σε πτώση στον 6ο αιώνα ο Κολομπάνος έφυγε για ταξίδι και πήγε στην Ευρώπη ε, ένας προσκυνητής και είναι ο Άγιος ο Πατρίκιος που είναι προστάτης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ο πρώτος που ποτέ ε, ανέφερε τη λέξη ε, Ευρώπη. Αν το μονοπάτι της ειρήνης πρέπει να προχωρήσει κι άλλο, να περάσει από μέρη τα οποία πλήττονται σκληρά από τη σύγκρουση, από τη Φλάνδρα, από τα Βαλκάνια και να καταλήξει και στη Λευκοσία, να συνδέσει τα δύο διερεμένα νησιά από τις δύο πλευρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναντώντα ξένου στον κόσμο, οι ταξιδιώτε θα μάθουν η μένα από του δε. Θα μάθουν πώ οι άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα, θρησκεία, ηλικία, φύλλο έχουν την ίδια ανθρωπιστική υφή. Και για εκείνου που δεν θα κάνουν αυτή την πορεία, θα υπάρξει ένα μονοπάτι εικονική πραγματικότητα. Τρισδιάστατη εμπειρία του μονοπατιού αυτού. Ήδη αναπτύσσεται αυτό ε, και αυτό το μονοπάτι και διαδικτυακή μορφή μπορεί να γίνει ένα ιστορικό βιβλίο ύψης της τεχνολογίας για τη νέα γενιά των παιδιών που πάνε στο σχολείο των μαθητών. Θα μάθουν τα παιδιά, θα έχουν την εμπειρία του πώς οικοδομήθηκε βάσει της ειρήνης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα τελικό πράγμα να πω, ότι το όνομα Κολουμπάνους δεν είναι σύμπτωση, είναι λευκό περιστέρι στα αγγλικά. Κολουμπάνους και όπως σας είπα περιγράφηκε σαν ο προστάτης της Ευρωπαϊκής Ενότητας. Ο Κολομπάνος δεν είναι ηρωνικό ότι ξεκίνησε από εκεί που είναι η Βόρεια Ιρλανδία, τότε ήταν η Ιρλανδία και είναι στο επίκεντρο τώρα της καταιγίδα του Brexit η Βόρεια Ιρλανδία με πολλές προσπάθειες που καταβάλλονται να προστατευτεί η ειρηνευτική διαδικασία και να προωθηθεί η ειρήνη και να προστατευτεί η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής Πάση Θυσία. Εν κατακλείδη να πω ότι η Βόρεια Ιρλανδία είναι στο μάτι του κυκλώνα και μπορεί να δώσει τη λύση. Μια λύση που προστατεύει την ειρηνευτική διαδικασία, θα προωθεί την ειρήνη σε όλο τον κόσμο και θα διαδίδει ένα απλό αλλά ισχυρότατο μήνυμα που ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν. Όταν κανείς θέλει υπάρχει και ο δρόμος, ανοίγει και ο δρόμος για το λευκό περιστέρι. Μου μένουν τυπώσα 26 δευτερόλεπτα. Α, ούτε δεν έβλεπα το ρολόι. Τέλος πάντων, κακό που δεν ξεκίνησα να ευχαριστήσω την ομάδα και την ομάδα μελέτης και τον πρόεδρο είναι εδώ και ίσως ε, δείξατε, δείξαν κάποια υπομονή ε, τώρα εδώ που έδειξα τόση δημιουργικότητα και εξίσου σημαντικό πήγαμε στο Belfast και είδαμε τις τοποθεσίες των γραμμών των διχαστικών που διαιρούσαν τον Belfast και έδειξα πόσο σημαντικό είναι αυτό το εγχείρημα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν. Ευχαριστώ, Τζέιν. Μάλιστα. Έκλεισε ο κατάλογος των αγορητών. Σα Father. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια Τζέιν. Μπράβο σου για την εξαιρετική σου γνωμοδότηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, σε αυτούς τους πολιτάρχους καιρούς ε, που αντιμετωπίζουμε και λόγω του Brexit να γυρίσουμε στις ρίζες μας, να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και να θυμηθούμε γιατί δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, κατασκευάσουμε ένα σχέδιο, να καταρτήσουμε ένα σχέδιο που θα το αντιληφθούν, θα το καταλάβουν, θα το κατανοήσουν και οι επόμενες γενναίες και θα νιώσουν την, το δεσμό που υπάρχει μεταξύ Ευρώπης και ειρήνης. Και Πολύ καλή αυτή η ιδέα σου και θα πρέπει να την προβάλλουμε όσο γίνεται την ιδέα του δρόμου του Λευκού Περιστεριού. Και πιστεύω ότι και οι ε, τροπολογίες θα εμπλουτίσουν την έκθεση ώστε να δουν όλοι και οι νέοι στην Ευρώπη που δεν βρίσκονται ακόμη σε αυτό το μονοπάτι, το συγκεκριμένο μονοπάτι του Λευκού Περιστεριού, να κάνουν και αυτοί κτήματος αυτή την προσπάθεια και να συμπαραταχθούν ε, σε αυτή την ε, ειρηνευτική προσπάθεια και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ιρλανδία είναι πολύ ε, ε, έντονο αυτό το αίσθημα. Αναφέρω τον Κολουμπάνο η Τζέιν και από το... Ε, σίγουρα είχαμε τον πολιούχο που προήλθε και από την Βόρεια Ιρλανδία και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό και στις τροπολογίες. Ευχαριστώ θερμά, Τζέιν, γιατί είναι περίλαμπρη απόδειξη ότι δεν νοείται απόσχηση από την αλληλεγγύη. Και θα πρέπει αυτή την αλληλεγγύη να την προτάξουμε έναντι του φόβου. Ευχαριστώ, Τζόναθαν Πίλ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Τζέιν για την αρτιότατη της γνωμοδότηση και χαιρόμαστε πάντα όταν μιλούμε για, τους, ε, για τις ε, των ε, Ιρλανδών στο Μεσαίωνα και πώς βοήθησαν ε, την υπόλοιπη Ήπειρο να φτάσει στη γνώση. Και νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη αυτή η γνωμοδότηση Πολλό δε μάλλον που αμφισβητείται ακόμη και η συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή, κάτι που δεν είχε γίνει την τελευταία 20 ετία. Η συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή έχει ξαναέρθει στο προσκήνιο και στο φω τη δημοσιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, είναι ένωση, ε, κοινότητα ειρήνη. Ήταν, είναι και θα είναι. Και γι' αυτό είμαι φιλοευρωπαίο και στρατευμένο φιλοευρωπαίο. Και έχουμε φυσικά αυτή τη, τη διαίρεση στη, στο νησί της Ιρλανδίας και μάλιστα ήδη από τότε που ήμουν στο Πανεπιστήμιο το επισήμανα και είναι κάτι που ε, μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές ε, και είχα ευαισθητοποιηθεί από την αρχή. Δεν θέλω επουδενή σκληρό σύνορο στην Ιρλανδία και πάλι η κατάσταση δεν είναι σίγουρη και έχει επανέλθει αυτό το θέμα. Και δεν πρέπει να θυμίζουμε μόνο την Παραϊλανδία ή δηλαδή, την Κύπρο. Υπάρχουν και άλλες ε, ε συγκρούσεις που χάρη στο ευρωπαϊκό ιδεώδες ε, ξεπεράστηκαν και ελπίζω να μην ξαναβγούν ποτέ στην επιφάνεια. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να δώσουμε στο 1-5 έμφαση στην εκπαίδευση, στην καλλιέργεια, στην επιμόρφωση και φυσικά να αναμίξουμε και τους νέους. Και σίγουρα η παιδεία είναι το υπέρτερο αγαθό και η απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ειρηνικό μέλλον. Πιέρ Κοραλμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ θερμότατα τη Τζέιν για την ε, καταπληκτική της πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτά τα μονοπάτια της ειρήνης, ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται ότι χάνουμε ένα πολύ σημαντικό μέλος της κοινότητάς μας ένα πολύ αξιόλογο μέλος της κοινότητάς μας. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε αυτό το δρόμο του Λευκού Περιστεριού. Χρειαζόμαστε και άλλα τέτοια μονοπάτια της ειρήνης. Ίσως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και την ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα τέτοιο μονοπάτι. Να δει ο κόσμος ε, πώς ε, μπορεί να συνεργαστεί με τον συνάνθρωπό του απολαμβάνοντας την ειρήνη και την ελευθερία. Στην ε, Βόρεια Ευρώπη το καλοκαίρι ο ήλιος δεν δει ποτέ. Μπορεί κανείς ε, να μείνει άγρυπνος όλη τη νύχτα απολαμβάνοντας το καλοκαίρι. Το λέω από προσωπική πείρα. Πάντως ε, η πρόταση είναι θαυμάσια, συγχαρητήρια και ελπίζω να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρομάτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα την τιμή να είμαι ο πρόεδρος της σχετικής ομάδας εργασίας και πραγματικά εκτίμησα ιδιαίτερα τις ε, συζητήσεις που έγιναν και ε, είμαστε όλοι υπόχρεοι στην Τζέιν και στη δημιουργικότητά της γιατί είναι πραγματικά οραματίστρια, πιστεύει στην ειρήνη και στην επανασυμφιλίωση και η επίσκεψή μας στο Μπέλφα στη Βόρεια Ιρλανδία μας άνοιξε πραγματικά τα μάτια και μας ευαισθητοποίησε μια κατάσταση για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανη. Γιατί αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχαμε ειρηνική επανασυμφιλίωση στη Βόρεια Ιρλανδία, κάτι που μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε, να διαφημίσουμε, να προβάλλουμε όσο μπορούμε αυτά τα επιτεύγματά μας στον τομέα της ειρήνης και δεν θα πρέπει ε, να, είμαστε, να, να είμαστε συναισθαλμένοι γι' αυτό οι διακριτικοί. Δυστυχώς, λόγω της παταγώδους αποτυχίας του Brexit, όλη η διαδικασία τη ειρηνευτική στη Βόρεια Ιρλανδία ε, κινδυνεύει με κατάρρευση, αν δεν την προσέξουμε ιδιαιτέρως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Γι' αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να ενθαρρύνω την Τζέι να συνεχίσει την αξιόλογη της προσπάθεια, όχι μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και να προωθεί και να προβάλλει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέα ειρήνης και επανασυμφιλίωσης, προσφέροντας τις βέλτιστες πρακτικές της και σε άλλες χώρες και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Η Κολομβία είναι επίσης ένα εύστοχο παράδειγμα. Εκεί μπορούμε να δείξουμε πραγματικά την ακολουθητή απορία. Μπράβο σου Τζέιν και καλή τύχη. Ισβαν Κομορόφσκι, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, αντίθετα με τους ε, προηγούμενους ομιλητές, εγώ θα σε συγχαρώ, Τζέιν, γιατί στην Ουγγαρία δίνουμε συγχαρητήρια όταν έχουμε μια επιτυχία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να μιλούμε για τον Brexit και τα αποτελέσματά του, δεν είναι επιτυχία. Και για να σα πω την αλήθεια, ως ε, ε, πρώην του Προεδρείου δεν ήμουν υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας. Είχα καταψηφίσει ε, αυτή την πρόταση. Γιατί να ξοδεύουμε χρήματα για κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως θα λάβει χώρα το Brexit στα τέλη Μαρτίου. Αντιλαμβάνομαι πάντως την, την ιδέα σου για το διαιρεμένο νησί και ήταν σημαντικό να έχουμε τελικά αυτή την πρόταση. Πριν από λίγο μιλήσαμε για την παραπληροφόρηση, για τα fake news και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν την κατάσταση. Γιατί και στη, στα σύνορά μας, στην Ουκρανία, ε, την Κρυμαία, τη Ρωσία, έχουμε πολλά γεγονότα. Και η δική μου πατρίδα Ουγγαρία είναι πολύ κοντά σε αυτά τα ανατολικά σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν σίγουρα να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία και στη σταθερότητα στην Υπηρώ και στη γειτονία της. Τώρα, ποιε είναι εξελίξει για το Brexit, ε, ρώτησα πολλού συμπολίτε σα. Ακόμη και σήμερα, 20 Μαρτίου, λίγε μέρε πριν το Brexit, δεν έχουμε ιδέα πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα γίνει. Δεν θέλω λοιπόν να σα συγχαρώ, μια και δεν πρόκειται για επιτυχία, αλλά σίγουρα είναι πολύ άρτια, τεκμηριωμένη και επίκαιρη η γνωμοδότησή σου. Ο κύριος Μέτσλερ ο τελευταίος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Jane, ε, προέρχομαι μια χώρα, τη Γερμανία δηλαδή, που μπόρεσε να ρίξει το τείχος που την χώριζε και είναι σε κεντρική θέση στην Ευρώπη. Γι' αυτό και θεώρησα ότι με... ήταν συναρπαστικό το ταξίδι στην ε, Βόρεια Ιρλανδία. Και θυμούμαι καλά επίσης και τον τοίχο που χωρίζει την Λευκοσία ε, στη μέση. Αυτά τα μνημεία, θα τα πω μνημεία, η σύνδεση των μνημείων αυτών ε, είναι και ο στόχος της δράσης της Τζέιν, την οποία ξεκίνησε για λογαριασμό μας. Και συγχαίρω όλες και όλους που υποστήριξαν τη συναδελφό μας, η οποία ακολουθεί ένα δρόμο και στην οποία πορεία θέλουμε και εμείς να την συνοδεύσουμε και να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το έργο αυτό. Υπάρχουν στην Ευρώπη πολλές περιοχές που χρειάζονται υποστήριξη. Βόρεια Ιρλανδία και Κύπρος. Πρέπει να βοηθήσουμε και τις ε, περιοχές αυτές και τις χώρες αυτές να μπορέσουν να υπερβούν τις διαιρέσεις. Άρα δίνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα μέσα από την καρδιά της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τζέιν, έχεις ένα λεπτό για να απαντήσεις. Σας ευχαριστώ και σε ένα δευτερόλεπτο αν θέλετε. Καταρχήν, ευχαριστώ τους συναδέλφους για την θερμή υποστήριξή τους. Χρειαζόμαστε την ελπίδα, σίγουρα. Και παρόλα αυτά, μας έχει συνταράξει το Brexit. Ε, έχουμε μεραχολήσει, έχουμε πάθει κατάθλιψη, αλλά δεν θα πρέπει να μας αποσταθεροποιεί. Ξέρουμε τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Τώρα για το κόστος. Ε, κάποιο κόστος χρειάζεται. Δεν χρειαζόμαστε πάντα αυτοκινητόδρομο, καλά είναι και τα ποδήλατα, αλλά υπάρχουν ανάγκες παρόλα αυτά. Επίσης, το θέμα της παιδείας. Πολύ σημαντικό το θέμα της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και το λέμε και σε άλλες γνωμοδοτήσεις. Θα πρέπει να αρχίσουμε να επιμορφώνουμε τα παιδιά, να τα διαπαιδαγωγούμε και να μπορέσουμε ε, μέσω μιας εικονικής πραγματικότητας ε, να δουν τα χαρακόμματα, να περπατήσουν στα Βαλκάνια, να δουν τις διαφορές μεταξύ του Βορρά και του Νότου, ε, να, δει να δουν την κατάσταση στη Σκοτία. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο ε, συμπλήρωμα για να ξυπνήσουμε την περιέργεια των νέων να επισκεφθούν τα διάφορα μέρη. Και αν μπορούσαμε όλοι να αρχίσουμε να περπατάμε με το σωστό τρόπο το, στο δρόμο του Λευκού Περιστεριού, αυτό θα μας οδηγήσει στη διέξοδο. Και να βρούμε κάτι που να έχει σημασία, να μιλάει στην καρδιά του πολίτη και να εμπλακούμε όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Ας περπατήσουμε όλοι μαζί στο δρόμο του Λευκού Περιστεριού. Ευχαριστώ, Τζέιν. Πάμε στις τροπολογίες. Δεν έχουμε και πολλές. Τροπολογία 1. Είναι δεκτή από την εισηγήτρια. Είναι κανείς κατά. Όχι. Τροπολογία 2. Επίσης τη δέχεται η εισηγήτρια. Είναι κανείς κατά. Όχι. Και τροπολογία 3. Επίσης δεκτή από την εισηγήτρια. Είναι κανείς κατά μήπως. Όχι. Οπότε τελική ψηφοφορία του ΡΕΞ 504 το νοδρόμο του Λευκού Περιστεριού, Wide of Way, για μια στρατηγική παγίου ειρήνη υπό την ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρχεται η ψηφοφορία. Η συγγήτρια ήταν η κυρία Τζέιν Μόρις. The vote Τέλος ψηφοφορίας. 164 3 κατά αποχές. Εγκρίνεται και μπράβο σου Τζέιν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Τζέιν για το έργο της που ξεκίνησε όταν ήταν πρόεδρος της ομάδας 3. Ήταν κοινή μας προσπάθεια και σου είχα υποσχεθεί τότε Τζέιν ότι και να συμβεί με αυτές τις δημιουργικές και ενδιαφέρουσες ε, διαπραγματεύσεις του Brexit. Ε, εγώ θα δώσω το παρόν στο Belfast όταν ανοίξουμε, κάνουμε τα γένεια του δρόμου για το Λευκό, του Λευκού Περιστεριού και στη Λευκοσία επίσης για τη συνέχιση αυτού του μονοπατιού. Ένα λεπτό για να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για κάτι πολύ δυσάρεστο που συνέβη στην πατρίδα μου την Ιταλία το απόγευμα. Κοντά στο Μιλάνο ένα λεωφορείο με 51 μαθητές με οδηγό από τη Σενεγάλη ε, αποφάσισε να ε, βάλει φωτιά στο λεωφορείο για να πάρει εκδίκηση από, για τα παιδιά και τις γυναίκες που χάνονται στη Μεσόγειο κατά δήλωσή του. Ευτυχώς χάρη στην ταχύτατη παρέμβαση της αστυνομίας, επέμβαση αστυνομίας δεν μπόρεσε να επιτύχει διότι σώθηκαν όλα τα παιδιά και συνελήφθη ο τρομοκράτης. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι το εξή. Ο Ιταλός συντονιστής της Ευρωπαϊκής Task Force κατά της παραπληροφόρησης και των fake news αμέσως, την, την αμέσως επόμενη ώρα ξεκίνησε εκστρατεία κατά τον τρόλ τα οποία άρχισαν να στοχεύουν, να επιτίθενται κατά των μεταναστών, των μαύρων και να ζητούν μποϊκοτάρισμα όλων των πολιτικών δυνάμεων που τάσσονται υπέρ των ανοιχτών θυρών για τους μετανάστες. Άρα η γνωμοδότηση την οποία ψηφίσαμε προηγουμένως έχει προφανή αξία για, το, για την ελευθερία και δημοκρατία και το πόσο σημαντικές είναι αυτές για την κοινωνία μας. Τώρα, επειδή έχει βρεθεί στο μεταξύ η συμβαστική ε, λύση, η συμβαστική τροπολογία δηλαδή, θα παρακαλέσω τον συνάδελφό μα να έρθει εδώ στο Προεδρείο και να την παρουσιάσει. Μάλιστα. Με υπερηφάνεια σας ανακοινώνω ότι για το 6.4 καταλήξα σε συμβασμό οι ομάδες 6.2 και 6.4. Λέμε λοιπόν η ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν ταχείες αποκρίσεις και ταχεία και επίγουσα χρηματοδότηση σε ποιοτική παιδεία, έρευνα και ανάπτυξη, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί χρονικά απέναντι σε άλλες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις σε ό,τι αφορά τη δαπάνη ποσοστού του ΑΕΠ για την αύξηση των δεξιοτήτων για να υπάρξει ανταγωνιστικό περιβάλλον. Να λοιπόν τώρα η συμβαστική τροπολογία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κοινό ενδιαφέρον και κοινή ευθύνη εργοδοτών και εργαζομένων να συμβάλλουν στην εκπαίδευση για την αύξηση των δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, νέων και ενηλίκων, για να ενισχυθεί η ικανότητα του εργατικού δυναμικού και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών μελών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών. Συνεχίζει η παράγραφος με μια τελευταία φράση, ώστε να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία πιο ψηφιακή. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το απαραίτητο μεταβατικό πλαίσιο για την τεχνολογική αλλαγή, ώστε να διασφαλιστεί η βελτίωση των βιωτικών και εργασιακών συνθήκων, βελτιωμένης ποιότητας απασχόλησης και πιο ισότιμη κοινωνία. Σας ευχαριστώ για την καλή σας εργασία, δηλαδή για την συγχώνευση των δύο κειμένων. Υπάρχει κανείς ο οποίος είναι κατά. Ωραία. Επικυρώνουμε λοιπόν την, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προηγουμένως και ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδοτήσεως. Για το μέλλον όπως έχει ζητήσει η Ρουμανική Προεδρία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Τελείωσε η ψηφοφορία. 147 υπέρ, 6 και 9 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Θα δώσω τώρα τα ε, η νέα της συζήτησης στην κυρία Κάνιο. Συμφώνησα με την Αντιπρόεδρο. Από εδώ και μπρο κάθε παρέμβαση το πολύ ενός λεπτού. Θα είμαστε λοιπόν αυστηρότατοι ώστε να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε στον προβλεπόμενο χρόνο. Ορίστε Ιζαμπέλ. Μάλιστα. Θα εξετάσουμε τη γνωμοδότηση του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων ΡΕΚΣ 505 Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Τζόναθαν Πιλ και έχει τρία λεπτά για να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του. Σας θέλουμε παρακαλώ να είμαστε αυστηροί στην τήρηση του χρόνου γιατί μας έχουν μείνει τέσσερις γνωμοδοτήσεις. Τρία λεπτά αντί για πέντε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερω που είμαι ακόμη εδώ, κοντά σα. Και βλέπω ότι έχουν μείνει πολλοί συνάδελφοι και στην αίθουσα. Χαίρομαι και γι' αυτό. Έγινε τελευταία στιγμή η γνωμοδότηση αυτή, γιατί έπρεπε να υποβληθεί στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το τι συμβαίνει στο κανάλι της Μάχης, αλλά γιατί η έπρεπε μέσα σε τέσσερις μήνες να απαντήσει okay. και επειδή λίγο πριν τα Χριστούγεννα λάβαμε την πρόταση, είχαμε μόλις ένα τρίμηνο για να καταρτήσουμε γνωμοδότηση. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία και την ομάδα μελέτης για τη βοήθεια και κυρίως την ομάδα μελέτης για τις πολύ χρήσιμες προτάσεις και την υποστήριξη. Αυτή η κοινή ανακοίνωση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απογοήτευση γιατί έχει πολλά κενά, πολλά στρατηγικά κενά και πραγματικά είναι μια χαμένη ευκαιρία. Στη γνωμοδότηση ε, επισημαίνουμε 16 βασικά κενά και με μια ε, τροπολογία του, της κυρίας Μόρης 17 ε, κενά. Θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα ακόμη. Δεν υπάρχει ούτε σχέδιο δράσης, ο δικός χάρτης, ούτε όραμα για το μέλλον, για την επόμενη δεκαετία. Ε, θα είναι συμπληρωματικές αυτές οι σχέσεις με την Ασία ή οι ανταγωνιστικές με, και με την Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ινδονησία έχουμε πολλές ε, συστημικές οικονομίες στην Ασία και έχουμε πολλές παγκόσμιες οικονομίες, όχι μόνο την Κίνα και το Ιράν και την Ευρασιατική ίσω ε, Οικονομική Ένωση. Η ανακοίνωση όμω Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελάχιστα ε, μας βοηθά να κατανοήσουμε την Ασία και τις διάφορες, τα διάφορα χαρακτηριστικά της και τη μεγάλη διαφοροποίηση. Και δεν λέει τίποτα για τις ε, προκλήσεις που έρχονται από την Ασία, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Ινδία, από όπου και προέρχονται. Ε, είχα, ε, μάλιστα είχαμε εμπορικές συμφωνίες με την Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και Βιετνάμ. Αλλά ούτε και αυτό το λέει η Επιτροπή. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε για το εμπόριο. Έτσι φαίνεται. Επίσης, τα, οι φορεί παρακολούθηση κοινωνία των πολιτών. Σημαντική καινοτομία για την Κεντρική Ασία. Ούτε και αυτά αναφέρονται. Ούτε και τα κοινωνικά κριτήρια που θέλαμε να συζητήσουμε. Δεν αναφέρεται σχεδόν η Ινδία πουθενά. Πρώτα απ' όλα όμως δεν αναφέρεται η πρωτοβουλία της Κίνας ένας δρόμος μια ζώνη. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα και κάθε ασιατική χώρα θα πρέπει να περιμένει ε, μια αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρωτοβουλία της Κίνας ένα ένας δρόμος μια ζώνη. Και αν μιλούμε για σφαίρες επιρροής, τότε αυτή η πρωτοβουλία της Κίνας, One Belt, One Road, ίσως είναι η δική της προσπάθεια δημιουργίας ε, σε πυρών. Τι είναι, απειλή ευκαιρία η σχέση με την Ασία. Και όταν επισερχόμαστε σε πιο διεξοδικε αναλύσεις, ενέργεια για παράδειγμα, υπάρχει τεράστιο θέμα στην Κεντροανατολική Ασία και στρατηγική πρόκληση σε ό,τι αφορά του υδρογονάθρακε. Και αυτό το τιμά όμω είναι πολύ σύντομο. Για το νερό δεν υπάρχει τίποτα στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τίποτα για το περιβάλλον, για το πώ θα αντιδράσουμε στην αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων, Μεταφορέ, επανάληψη ουσιαστικά των προτάσεων του 2011 και 2015 και για τον ψηφιακό κόσμο. Τι γίνεται με τι χώρε που έχουν διαφορετική άποψη από εμά, αλλά και οι διαπροσωπικέ σχέσει. Ε, Εκείνη που έχουμε τεράστια κενά στην Ένωση, στι διαπροσωπικέ σχέσεις. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Πιλ. Περνάμε στη συζήτηση. Το λόγο έχει η κυρία Σλάβοβα. Και σας υπενθυμίζω ότι μόνο ένα λεπτό έχει ο κάθε ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Τζόναθαν για αυτή τη γνωμοδότηση. Είναι πολύ επίκαιρη αυτή η ανακοίνωση και υποστηρίζουμε ότι εστιάζεται αυτή επί βιώσιμη διασυνδεσιμότητα που βασίζεται επί κανόνων. Πρέπει να είναι σαφέ. Η ανακοίνωση αναφέρεται στι χαμένες ευκαιρίες μέσω τη επικοινω... της ανακοίνωσης αυτής. Εκεί δεν το τόνιζε καλά η ανακοίνωση. Η ομάδα Μελέτη και ο Τζόναθαν το τόνισαν στο κείμενο όπω έπρεπε. Και τα στατηγικά κενά και σημασία που έχουν. Σωστά καλύπτονται με τις προτάσεις που αναφέρονται στη γνωμοδότηση. Ελπίζω όλες οι προτάσεις μας που απαριθμούνται σαφώς στην ε, γνωμοδότηση να ληφθούν υπόψη στο μέλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβουλίο Συγχαρητήρια λοιπόν στον Τζόναθαν και σε όλη την ομάδα που επεξεργάστηκε το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ευχαριστούμε κυρία Σλάβοβα και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που τηρήσατε το χρόνο σας. Ο κύριος Ματσόλα έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να τονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η γνωμοδότηση και η έκθεση της, Ευρω... Επιτροπής που σχετίζεται με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Κίνας που θα γίνει αρχές Απριλίου και χώρα μου, στη χώρα μου θα έρθει μεγάλη αντιπροσωπεία και ο Κινέζος Πρόεδρος θα έρθει στη χώρα μου και θα συζητήσουν και την πρωτοβουλία αυτή. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να πω κάτι. Τα δίχτυα επικοινωνιών, μεταφορών, ενέργειας. Ε, λοιπόν, ο, Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται από το Open Road Initiative και με μεγάλη πρωτοβουλία που έχουμε σε διεθνέ προσκήνιο για οικονομική ανάπτυξη. Είναι μια πρωτοβουλία με την οποία οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει πολύ συχνά ε, την βλέπουν με αρνητικό μάτι. Εγώ προσωπικά μπόρεσα στην Ινδονησία, στην Ταϊλανδία, σε διάφορε περιπτώσει μπόρεσα να έρθω σε επαφή με την κινέζικη πρωτοβουλία και λέω ότι θα πρέπει οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να έχουν τα μέσα τους να έχουν μια ανάλογη πολιτική για να μπορούν να συμμετέχουν στις μεγάλες προσπάθειες κατά σε επίπεδο όσον αφορά τα δίκτυα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάτερ. Κύριε Πάτερ, μπορεί να βλέπετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η ανακοίνωση αυτή είναι πραγματικά μια χαμένη ευκαιρία. Φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τόσο επιφανειακά, τόσο σοβαρές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια τόσο περίπλοκη ήπειρο όπως είναι η Ασία. Και μάλιστα έχουμε και ε, συνόδους κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασίας που πραγματεύονται πολύ σημαντικά θέματα. Δεν μπορούμε να τόσο το θέμα να το αντιμετωπίζουμε τόσο απλά. Και δεν μπορούμε φυσικά να είμαστε εξαντλητικοί, γιατί είναι ένα ευρύτατο ζήτημα. Σταθήκαμε στα ουσιώδη που μας τα παρουσίασε και ο εισηγητής ή άλλωστε και το, η ομάδα εργασία, ε, η υποεπιτροπή δέχτηκε την έκθεση του. Πολύ άρτια η προσπάθειά σου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί τελευταία στιγμή υπέβαλε την ανακοίνωσή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σε έκανε ό,τι μπορούσε και νομίζω ότι η ΕΟΚΕ στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα και στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει με πολύ πιο υπεύθυνο και πολύ πιο θεματικό και πιο διεξοδικό τρόπο να πραγματεύεται τα ζητήματα που αφορούν την Ασία. Και όχι όπως το έκανε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Σας ευχαριστώ κύριε Πάτερ. Το λόγο έχει και πάλι ο εισηγητής μας. Το πολύ για δύο λεπτά, αν μπορείτε και λιγότερο τόσο το καλύτερο. Και φυσικά θα έχετε το λόγο και αργότερα στις ε, τροπολογίες. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές. Πολύ, πολλά σημαντικά θέματα έχουμε συνέσω, όχι μόνο την Κίνα. Και να παράγει δεκατή σελίδο κείμενο Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού του θέματος, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία που χάθηκε. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε. Ευχαριστούμε κύριε Πιλ. Περνάμε στις τροπολογίες. Τέσσερις τροπολογίες έχουμε και δύο συμβαστικές τροπολογίες, δύο εγκεκριμένε. Ξεκινάμε με την τροπολογία 3 του κυρίου Ματσόλα. Έχουμε μια συμβαστική τροπολογία που θα μας διαβάσει ο κύριος Πύλο, εισηγητής μας. Ναι, χρειάστηκε πολλή συζήτηση, περισσότερο από ό,τι θεωρούσα και περισσότεροι άνθρωποι συμμετείχαν από ό,τι περίμενα. Ε, λοιπόν, ε, μπορείτε να διαβάσετε, θα να διαβάσω ή μπορεί να διαβάσετε από τον πίνακα, από την οθόνη, τη συμβαστική είναι νέα σημείο 4.2.2. 4.2.2 που λέει η Επιτροπή σημειώνει ότι εκτιμώντας ότι στην Αφρική υπάρχουν μέσα υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ενώσεως για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και διάφορα κονσόρσια, αυτά δεν υφίστανται για τις διασυνδέσεις Ασίας-Ευρωπαϊκής Ευρώπης. Και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με κινέζικες εταιρείες που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία Build and Road και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επεκτείνει αυτή την πολιτική και να την εφαρμόσει και για την Αφρική. Και το Invest EU θα πρέπει να καλύπτει και κινδύνους επενδύσεων και στην Ασία καθώς και σε άλλα μέρη του κόσμου. Τέτοια υποστήριξη θα εφαρμόζεται ε, εξίσου σεβόμενη τα δικαιώματα των εργαζομένων σε διαγωνισμού σε τρίτες χώρες ε, που δέχονται ξένες επενδύσεις. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε κύριε Πίλ. Έχει κανεί αντίρρηση με τη συμβαστική τροπολογία. Όχι, οπότε περνάμε στην τροπολογία 1. Τροπολογία 1 του κυρίου Μόρκης. Γίνεται δεκτή. Έχει γίνει δεκτή μάλλον. Περνάμε στην τροπολογία 2 του κύριου Μόρκης και πάλι και αυτή έχει γίνει δεκτή. Είναι κανείς κατά μήπως. Όχι. Και τελευταία τροπολογία, η τροπολογία 4 του κύριου Ματσόλα. Θα μας εξηγήσει τη συμβαστική τροπολογία ο συγγετής ο κύριος Πίλ. Ευχαριστώ. Είναι ένα συμβαστική πολυσχηδής. Έχουμε ένα σημείο 1-6 που λέει η Επιτροπή φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επεκτείνει το μέσο για οικονομική και εξωτερική πολιτική που στηρίζει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κυρίως τα διάφορα κονσόρτσια που ήδη υπάρχουν για την Αφρική υπό την αιγίδα του Invest EU για να καλυφθεί η Ασία και άλλα μέρη του, του κόσμου. Τέτοια υποστήριξη θα πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου σεβόμενη στους διαγωνισμούς στα δικαιώματα των εργαζομένων σε τίτες χώρες ε, που δέχονται αυτές τις, είναι ε, επιλέξιμες για αυτές τις ξένες επενδύσεις. Μάλιστα. Είναι κανείς κατά της συμβαστική τροπολογία. Όχι, οπότε ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. 133 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Πίλ. Ε, Περνάμε στην επόμενη γνωμοδότηση του τμήματος Απασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων και Δικαιωμάτων του Πολίτη, υπαριθμό 575, με θέμα τη ευκαιρία απασχόληση για τον οικονομικό μη ενεργό πληθυσμό. Πρόκειται για γνωμοδότηση πρωτοβουλία και θα ήθελα να καλέσω τον εισηγητή, τον κύριο Κουστόντιο Λεϊριάου, να μα παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του εδώ στο βήμα. Δύο λεπτά έχει ο εισηγητή μα για να μα παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Α, τρία, τρία, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Α, τρία, τέλεια. Το σχέδιο γνωμοδότησης είναι απόρρια μελετών που έγιναν από την Επιτροπή μας και άλλο φορέα και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Φαίνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 23% ε, άνω των 60 ετών που είναι οικονομικά ανενεργοί πολίτες και 15 με 64 4 ε, ενήλικες 15, ηλικιες 15 64 τώρα ανήκουν στην κατηγορία του μη ενεργού πληθυσμού και δεν συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία ούτε έχουν επαρκές δεξιότητες, έχουν προβλήματα στην πρόσβαση στον υγειονομικό τομέα και μερικές φορές αντιμετωπίζουν ε, και προβλήματα στην οικογένεια. Υπάρχει αρκετή παροχή φροντίδας. Τέσσερι είναι αυτές είναι οι φραγμοί. Κυρίως οι νέοι αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα όταν έχουν αναπηρία και εντοπίσαμε τέσσερις ομάδες στόχους. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μία μελέτη για το θέμα αυτό. Τα αποτελέσματα όμως της μελέτης ε, δεν έδωσαν κάποια συνέχεια, δεν σε συγκεκριμένες δράσεις. Χρειάζονται νέες πολιτικές ε, και σχέδια δράση για να βοηθηθούν αυτές οι ομάδες του πληθυσμού και να δημιουργηθούν ε, ευκαιρίες απασχόλησης, ε, κυρίως για μη ενεργά τμήματα του πληθυσμού. Και να μην μείνει εγκαταλελειμμένο αυτό το τμήμα του πληθυσμού όταν θέλει να εργαστεί. Επίσης είναι σημαντικό με τις πολιτικές αποφάσεις σε κάθε κράτος μέλος να αρθούν τα εμπόδια που υπάρχουν και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που έχουν τα άτομα αυτά για να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην κοινωνία. Και φυσικά να λάβουμε υπόψη ιδιαιτερότητες στις ανάγκες των γυναικών ή σε άλλα τμήματα του ανενεργού πληθυσμού. Και επαναλαμβάνω ιδιαίτερα τους ε, ανθρώπους που είναι σε ηλικία 15 με 64 χρόνια. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ε, να προσφέρουν ειδική αρρωγή σε ανθρώπους που θέλουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, ικανότητες, τα εφόδια και τις ειδικέ ανάγκες κάθε υποομάδας από αυτές που εντοπίσαμε και στη μελέτη της Eurofound. Επίσης, ε, να στηρίξουμε τη μεγαλύτερη κινητικότητα του πληθυσμού, να δούμε που υπάρχουν και νέες θέσεις εργασίας, που υπάρχει έλλειμμα και να λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε υποομάδας. Επίσης, να δοθούν ενισχύσεις στους εργοδότες που είναι πρόθυμοι να προσλάβουν άτομα αυτών των ειδικών ομάδων. Να δώσουμε ιδιαίτερα επιδόματα σε εργοδότες που θέλουν να συμπεριλάβουν στις επιχειρήσεις τους ε, τέτοιους τέτοια άτομα. Τελειώνεται, λέει πρόεδρο. Καλώ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα της πρότασης για την βιομηχανία 4.0. Ε, γιατί στη νέα αυτή εποχή θα χαθούν πάρα πολλέ θέσει εργασία, οπότε θα πληγεί ακόμη περισσότερο αυτό το ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού που ήδη βρίσκεται εκτό τη αγορά εργασία. Θα ήθελα λοιπόν να σα συστήσω να εγκρίνετε τη γνωμοδότηση. Δυστυχώ δεν μπόρεσα να σα αναλύσω όλα τα επιμέρου σημεία αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Καλώ. Περνάμε στη συζήτηση. Ένα λεπτό χρόνο θα έχει ο κάθε ομιλητή. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Κόλε. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτή η γνωμοδότηση πραγματικά είναι σημαντική. Πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, παρόλα αυτά ε, δεν εμφανίζονται στα στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασία, σαν να μην υπήρχαν. Δεν εμφανίζονται στα στατιστικά. Από αυτή την οπτική γωνία θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία, εκ νέου να επανέλθουν στην αγορά εργασία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όχι μόνο αυτοί που θέλουν να εργάζονται λιγότερο ή δεν θέλουν να δουλέψουν. Μιλάω για εκείνους που θέλουν να δουλέψουν διότι θέλουν να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία. Να αισθανθούν ότι είναι χρήσιμοι και να έχουν και αύξηση του εισοδήματο θα έχουν πρόσβαση εισόδημα, σε μια αμοιβή και αυτό με τη σειρά του έχει αντίκτυπο στην καθημερινή του ζωή, στην οικογένειά του, στην ύπαρξή του. Μιλάμε λοιπόν για ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων εδώ και το βλέπουμε από αυτό το σημείο. Και βλέποντα το από εκεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι όλοι οι πολίτε Ευρωπαϊκή Ενώσεω έχουν το δικαίωμα στην απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένου τομεί πολιτική που θα εξετάζει αυτή την κατηγορία του πληθυσμού πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ να υποστηρίξετε αυτή την γνωμοδότηση. Muchas Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκραμπάλοβα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι πράγματι αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Στο τμήμα κοινωνικών υποθέσεων όλοι το επιβεβαίωσαν αυτό. Υπερψηφίσαμε αυτή τη γνωμοδότηση στην ΣΟΚ εγώ συνέταξα κάποιες τροπολογίες, δεν συμφωνώ με αρκετά σημεία. Αν θέλουμε να συμμετάσχει ο κόσμος στην αγορά εργασίας, πρέπει να δούμε τι δεξιότητες έχουν, ποιες φιλοδοξίες έχουν, αυτό βέβαια, αλλά και τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας πρέπει να δούμε. Διαφορετικά δεν μπορούμε να συντονίσουμε την προσφορά με τη ζήτηση. Και κάτι άλλο με το οποίο δεν συμφωνώ, ότι όλοι πρέπει να εργαζόμαστε λίγο. Αυτό σημαίνει η μείωση του αριθμού των ωρών εργασίας τον 21ο αιώνα υπάρχουν νέε τεχνολογίε, νέε μορφέ εργασία και σαν τέτοιο περιβάλλον η αδίποτε μείωση του αριθμού ωρών εργασία δεν είναι καλή λύση κατά την άποψή μου. Πιστεύω ότι και έχουμε και άλλε λύσει. ευχαριστώ. Η κυρία Μοντζεζέρσκη έχει το λόγο. <laughs> Κύριος είμαι, Μποντζεγεύσκη, όχι κυρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση αυτή, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε δύο θέματα. Καταρχήν, το ρόλο των τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, το, της τοπικής αυτοδιοίκησης ε, και των οργανώσεων που στηρίζουν αυτούς τους οικονομικά ανεναργούς ε, ε, συνανθρώπους μας. Για παράδειγμα, οι γιατροί που πηγαίνουν, επισκέφτονται αυτούς τους ανθρώπους, ε, κάνουν ε, τη διάγνωση και θα μπορούσαν ε, σε συνεργασία με τους εργοδότες να διευκολύνουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους την επαναφορά τους στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο της γνωμοδότησης. Άλλο θέμα είναι τα εμπόδια στην αγορά εργασίας για τις υποομάδες αυτές. Μερικές φορές έχουμε διακριτική μεταχείριση ανάλογα με τον τόπο διαμονής. Για παράδειγμα, κάποιοι που μένουν σε απόμακρες περιοχές, στην Ήπεθρο, σε αγροτικές περιοχές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμη πιο περιθωριοποιημένοι, πιο αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας λόγω της απόστασης. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε εδώ και το θέμα της επικοινωνίας και της πρόσβασης. Πάντως θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το συντάκτη της γραμματοδότησης και σας διαβεβαιώ ότι θα υπερψηφίσω ευχαρίστως την πρόταση αυτή. Μάλιστα, ευχαριστώ ο Πρόεδρος ναι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε ένα λεπτό θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους συνέβαλαν στην διατύπωση αυτού του σχεδίου γνωμοδοτήσεως που είναι έξοχο. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους θαραλέους που ήταν τα μέλη της ΕΟΚΕ που είναι ακόμα εδώ σε αυτή την αίθουσα στις 7 και 4. Θέλω να συγχαρώ στο τέλος ιδιαίτερα ε, τον εισηγητή διότι έχουμε την απόδειξη ότι πρόκειται περί ενός άντρα θαραλέου που βλέπει κατάφατσα τα κοινωνικά προβλήματα σε όλες τις κοινωνίες, έχει το θάρρος να λέει τα πράγματα που κάποιοι αμφισβητούν. Εν ίδια απαντήσεως στον Βλαντιμίρ, τον αγαπητό συνάδελφο που είπε ότι υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει όσον αφορά τη μείωση του χρόνου εργασία, θα ήθελα να ξέρω ποιε λύσει. Διότι κάθε φορά που προτείνουμε κάτι, αντιμετωπίζουμε μία δογματική αντίθεση. Αγαπητοί φίλοι, τις τελευταίε δεκαετίες. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε, τα κέρδη αυξήθηκαν, όλα αυξήθηκαν και η ανεργία όμως. Εάν θέλετε αυτή η Ευρώπη να συνεχίσει να υφίσταται, κάντε μια χειρονομία προς εκείνους που δεν έχουν τίποτα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Ποντέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θέλω να εξηγήσω γιατί κα, ε, κατέθεσα κάποιες, την 4, την 6 και τη 2, τις τροπολογίες. Αναφέρεται στην τυπολογία των εμποδίων που υπάρχουν για τους ε, ενεργά μέλη της κοινωνίας. Σε αυτά τα εμπόδια έχουμε και τις ε, μικρές δεξιότητες, εμπειρία περιορισμένη, επαγγελματική, προβλήματα υγείας και την ανάγκη εξασφάλισης των μελών της οικογένειας. Η μείωση του ωραρίου δεν είναι λύση για αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό λέγω ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε προβλήματα έλλειψης δυνατοτήτων, προβλήματα υγείας, ούτε την ανάγκη να διασφαλίσει κανεί την οικογένειά του μέσω τη μειώση του ωραρίου εργασία. Υπάρχουν χώρε, υπάρχει μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού και η μείωση του ωραρίου εργασία την εβδομάδα θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα για τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πολύ ισχυρό και αναλυτικό μήνυμα. Είναι πραγματικά απίστευτο πόσο στοχεύει ο εισηγητή στις περιθωριοποιημένες ομάδες ανθρώπων με αναπηρίες. Και μάλιστα μερικοί με 82,5% και πάνω. Συζητεί τη σημαντική πτυχή της ανάγκης ύπαρξης επιδοτούμενων προγραμμάτων που θα ενισχύσουν και το ΑΕΠ όλων των χωρών μελών. Και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ θετικό και αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Ο εισηγητή θα ήθελε το λόγο για να απαντήσει σε δύο λεπτά στους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που σχολίασαν την γνωμοδότησή μου. Θα ήθελα να φερθώ σε αυτά που είπαν η κυρία Μαγκλόβα και το Ποντέα. φαίνεται ο, η γνωμοδότηση μιλά για τον εβδομαδιαίο ωράριο εργασία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μείνει λίγοι εδώ, αλλά όσοι ήμασταν το πρωί εδώ, για πολλά χρόνια εργαζόμασταν έξι μέρες τη βδομάδα. Μέχρι τη δεκαετία του 70 ήταν έξι μέρες τη βδομάδα ο χρόνος εργασίας. Μετά το Σαββατοκύριακο απελευθερώθηκε. Και έτσι με την αλλαγή αυτή στο 72 χρόνο εργασία από 6 σε 5 μέρε, βελτιώθηκε το βιωτικό επίπεδο, βελτιώθηκε η ποιότητα ζωή. Και η μείωση του ωραρίου εργασία δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί και το βιωτικό επίπεδο. Το αντίθετο, βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο με τη μείωση του ωραρίου εργασία. Γιατί απελευθερώνοντα κάποιε ώρε εργασία, ε, ανοίγουμε την αγορά εργασία σε περισσότερα άτομα που αναζητούν ευκαιρία για να εργαστούν και φαίνεται ότι με την ψηφιοποίηση και τη βιομηχανία 4.0 θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης την επόμενη δεκαετία. Οπότε θα έχουμε χιλιάδες ανέργους. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση ε, για αυτούς τους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό η σημείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας ήταν μια λύση. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από το δημόσιο τομέα και μετά να επεκταθούμε στον ιδιωτικό. Πάντως αυτό θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό, γιατί αλλιώς μέσα στην επόμενη δεκαετία θα αντιμετωπίσουμε πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Καταστροφικά θα έλεγα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάντως συναδέλφους που υποστήριξαν την γνωμοδότηση και να πω ότι είναι σημαντικό να δοθεί μια συνέχεια στο μέλλον, να μην μείνουμε μόνο σε αυτή τη γνωμοδότηση. Γιατί το θέμα αυτό σίγουρα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του προβληματισμού και των ανησυχιών των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λέιραου. Θα περάσουμε στις ψηφοφορίες των τροπολογιών. Τέσσερις τροπολογίες έχουμε. Από ό,τι έμαθα, η πρώτη τροπολογία αφορά την τροπολογία... Έχει σχέση με την τροπολογία 3. Συμφωνεί ο εισηγητής. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες 1 και 3 ή θέλετε να τις ψηφίσουμε ξεχωριστά. Ξεχωριστά. Τροπολογία 1 πρώτα. Ζητά διαγραφή κάποιου τμήματος του κειμένου και έχει απορριφθεί. Θα μας εξηγήσετε γιατί, κύριε Σιγητά. Ή ποιος θέλει να υποστηρίξει πρώτα την τροπολογία. Κυρία Τερμπάλοβα, ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εάν πρόκειται για την τροπολογία της ομάδος 1, πρέπει να την εξηγήσουμε εάν την απορρίπτει ο εισηγητής. Ε, πρέπει να εξηγηθεί γιατί. creo que primero... Νομίζω ότι πρώτα θα πρέπει η συντάκτη της γνωμοδότησης να παρουσιάσει, ε, της, ε, της τροπολογίας, να μας παρουσιάσει την τροπολογία. Ευχαριστώ. Έχει καλώς. Όπως ε, είπα προηγουμένως, δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι θέλουμε να μειώσουμε τις τα εβδομαδιαία ωράρια εργασίας, διότι στην Ευρώπη Έχουμε προβλέψεις για ίση αμοιβή, για ίση ποσότητα εργασίας, αλλά θα βάλουμε τώρα και ίδιο ωράριο. Έχουμε σχετικές εμπειρίες στην τσεχική δημοκρατία από παλαιότερα, αλλά δεν αποτελεί λύση. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους να μπουν και αυτοί στην αγορά εργασίας. Ο εισηγητής μας έχει ένα λεπτό για να εξηγήσει γιατί είναι κατά της τροπολογίας αυτής. Μα ήδη σας το είπα προηγουμένως. Νομίζω ότι από τις αποτελεσματικότερες λύσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων αυτών είναι να μειώσουμε τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας. Και πριν από αρκετά χρόνια είχαμε αντίστοιχη περίπτωση και με τη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασία καταφέραμε να συμπεριλάβουμε στην αγορά εργασία πολύ περισσότερου ανθρώπου. Γιατί άνοιξαν θέσει απασχόληση, βελτιώθηκε το βιωτικό επίπεδο, έγινε καλύτερη κατανομή του πλούτου και όλα αυτά χάρη στη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασία. Γι' αυτό και είμαι κατά τη διαγραφή του σημείου αυτού. Νομίζω ότι με τη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους στην αγορά εργασία που σήμερα είναι άνεργοι. Και οι δύο ακόλουθε τροπολογίες συζητήθηκαν στην υποεπιτροπή και απορρίφθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν είμαι κατά. Καλώς. Ας ψηφίσουμε την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Y luego ya la, esta. ¿Quién, lo presenta? Ah, que necesita agua. Agua. mais il a, on n'a pas de verre, le problème. On a besoin d'un verre. Se cierra la votación. Τέλος ψηφοφορίας. A favor de la enmienda. 42 υπέρ, 63 κατά. 5 αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία. Περνάμε στην τροπολογία 2 που τροποποιεί κάπως το κείμενο και αυτή έχει απορριφθεί από τον εισηγητή. Θέλει κανείς να μας παρουσιάσει την τροπολογία. Έχει ένα λεπτό. Η κυρία Ντερμπάλοβα έχει το λόγο για ένα λεπτό να μας παρουσιάσει την τροπολογία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν κατανοώ καλά γιατί ο εισηγητής την αποδέχεται. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μπουν στην αγορά εργασίας, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Να δούμε ποιες είναι οι φιλοδοξίες τους, ποιες είναι οι ικανότητές τους, ποιες είναι οι απαιτήσει για την αγορά εργασίας και να μπορέσουν να προσαρμόσουν οι άνθρωποι αυτοί τις ικανότητες και τις γνώσεις τους. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την κατάσταση της αγοράς εργασίας το τι προσωπικό χρειάζονται οι επιχειρήσεις και πώ διαμορφώνονται οι ανάγκε του. Bien, ahora el... Μάλιστα, ένα λεπτό έχει ο Συγητή για να μας παρουσιάσει τη θέση του. Δεν συμφωνώ με την τροπολογία. Γιατί τροποποιεί την ουσία του κειμένου και βλάπτει τη συνέπεια και τη συνοχή του κειμένου. Γι' αυτό ε, σας προτείνω να την καταψηφίσετε. Μάλιστα. Περνάμε στην ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Se cierra Τέλος ψηφοφορίας. 38 ψήφισαν υπέρ, 66 κατά και 6 αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 4, που επίσης τροποποιεί το κείμενο. Έχει γίνει δεκτή όμως από τον εισηγητή. Συμφωνείτε με την τροπολογία 4. Κυρία Ντερμπάλοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για τροπολογία του εισηγητού. Δεν ήμουν προετοιμασμένοι ή διατεθειμένοι ε, να συζητήσω το θέμα αυτό, αλλά ε, νομίζω δεν μπορώ να συμφωνήσω, διότι ζητούμε από τις χώρες μέλη να βάλουμε ποσοστώσεις για την απασχόληση ανθρώπων με αναπηρίες και άλλα σχετικά. Έχουμε όμως 28 χώρες μέλη και αυτές έχουν δικά τους εθνικά συστήματα. είναι προφανέ ότι θα διαφέρουν τα εθνικά αυτά συστήματα. Έχω ένα παράδειγμα από την Τσεχική Δημοκρατία. Την στιγμή που συζητήσαμε την πρόθεση ποσοστώσεων, αντιτάχθηκαν οι ίδιες οι οργανώσεις αναπήρων. Ένα λεπτό ο εισηγητής και μετά θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν νομοθετικές ρυθμίσεις για τη συμπερίληψη περισσότερων ατόμων με αναπηρίες στις επιχειρήσεις τους και στις δημόσιες υπηρεσίες τους, στο δημόσιο. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, από φέτος τον Ιανουάριο ισχύει σχετική διάταξη. Άλλες χώρες όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ένα τέτοιο σύστημα ποσοστώσεων για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες. Γι' αυτό και προτείνω να προτρέψουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσουν ένα τέτοιο σύστημα, ένα, κάποιες ελάχιστες ποσοστώσεις απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρίες, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν και τον κύκλο εργασιών πολισεών τους, ώστε να απασχοληθούν περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρίε στην οικονομία. Μάλιστα. Ψηφίζουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Se cierra el voto. Τέλος ψηφοφορίας. 62 υπέρ, 41 κατά, 7 αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία 4. Και περνάμε στην τελευταία τροπολογία, την τροπολογία 3, που προτείνει διαγραφή μιας παραγράφου. αμα αυτή είναι η ίδια τροπολογία με την 1, που ήδη την ψηφίσαμε. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για δεύτερη φορά. Το κείμενο είναι ε, ταυτόσιμο. Οπότε έχει... Έχουμε ήδη ψηφίσει. Η κυρία Τερμπάλοβα. Όχι, όχι. Δεν είναι το ίδιο. Μάλλον παρόλο που είναι η ίδια τροπολογία, κατά το κύριο σώμα αυτή αλλά και στα συμπεράσματα, ωστόσο δεν συμβαίνει. Υπάρχουν διαφορετικέ αιτιολογήσει, να το εξηγήσω. Είπα ήδη για ποιο λόγο είμαι αντίθετη. Αλλά μια και μου δίνεται κάθε φορά μονάχα ένα λεπτό, είμαι υποχρεωμένη ε, να χωρίσω τα επιχειρηματά μου. Ο εισηγητής λησμόνησε να πει ότι το σύστημα εισήχθη στην Πορτογαλία, όχι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και δεύτερο, στο τμήμα ΣΟΚ, πολλοί αντιτάχθηκαν. Ακόμα και ο εισηγητής είπε ότι διερωτήθηκε γιατί υπήρχαν τόσες πολλές διαμαρτυρίες. Άρα δεν πρόκειται, δεν απηχείται εδώ η άποψη ολόκληρης της Επιτροπής δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα οποιοδήποτε συναδέλφου να διαφωνεί, να έχει αντιρρήσει, αλλά θα πρέπει να τηρήσουμε τον εσωτερικό κανονισμό που ισχύει εδώ και για 15 χρόνια στην Επιτροπή. Από τη στιγμή που έχουμε ε, ψηφίσει μια τροπολογία ε, ε, για το κείμενο ε, και μια άλλη τροπολογία έχει το ίδιο περιεχόμενο και αφορά τις συστάσεις, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τη δεύτερη τροπολογία από τη στιγμή που είναι ταυτόσιμες. Εγώ απλώ θέλω να τηρήσουμε τον εσωτερικό κανονισμό. Yo creo que... Νομίζω ότι όντω, και δώσαμε το δικαίωμα στην κυρία Νταρμπάλοβα να μα μιλήσει και να μα εξηγήσει τη θέση τη. Αλλά θεωρώ ότι εκπίπτει αυτή η τροπολογία. Μια και με βάση τον εσωτερικό μα κανονισμό και από τη στιγμή που έχουμε ψηφίσει τροπολογία που είναι ταυτόσιμη, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τη δεύτερη που είναι ίδια. Οπότε α ψηφίσουμε το σύνολο τη γνωμοδότηση. Διαδικαστικό θέλει να υποβάλει η κυρία Ντερμπάλοβα και μετά να τελειώνουμε. Ευχαριστώ. Βέβαια, δεν θέλω να υπονομεύσω την όλη διαδικασία, αλλά εσείς ε, οι ίδιοι δεν την τηρούσατε πάντα. Είχαμε και πριν ευαίσθητε γνωμοδοτήσεις, στην τελευταία ολομέλεια Φερρυπίν, και ψηφίσαμε την ίδια τροπολογία. Είτε ήταν για το κείμενο, είτε για τα συμπεράσματα. Οπότε, εν τη αυτή περιπτώση δεν είναι βολικό και στην προηγούμενη περίπτωση βόλευε. Σε αυτή την περίπτωση θα ψηφίσουμε. Όμω, α έχουμε υπόψη ότι οι τροπολογίε θα πρέπει να Εμφανίζω τις γνωμοδοτήσεις. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το να ψηφίσουμε. Bien, Όπως είπα και πριν, θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. El dictamen.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 Μάλιστα. 97 ψήφισαν υπέρ, 20 κατά και 6 αποχές. Οπότε η γνωμοδότηση του κυρίου Λιράου εγκρίνεται. Θα ήθελα να πω στην κυρία Τερμπάλοβα Επαναλαμβάνω, θα ήθελα να πω στην κυρία Ντερμπάλοβα και στην Ομίγυρη ότι τηρήσαμε πιστά το άρθρο 55 παράγραφος 4 του νέου εσωτερικού κανονισμού που το λέει ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Απλώς θέλω να εξηγήσω γιατί έλαβα τη σχετική απόφαση και σε ποιο άρθρο στηρίχθηκα του εσωτερικού κανονισμού. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά για την γνωμοδότησή σας. Ε, σας ευχαριστούμε κύριε Κουστόδιο. Λιεϊράου. Muy bien. Vamos a pasar... Πολύ ωραία. Περνάμε στην επόμενη γνωμοδότηση του τμήματο Εξωτερικών Σχέσεων υπαριθμών 506, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρωμεσογειακή περιοχή, ενημερωτική έκθεση. Η συγγήτρια είναι η κυρία Σύνθια Ντελρίο, που θα έρθει για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή της. Eh, Ευχαριστούμε. Έχει τρία λεπτά, Σύνθια, για να μα παρουσιάσει την γνωμοδότησή σου. Λοιπόν, με τα βίας που μπορώ να πάρω τρία λεπτά, αυτή η έκθεση για την κατάρτιση είναι αποτέλεσμα κοινή προσπάθειας που καταβάλαμε όχι μόνο στην ομάδα μελέτης αλλά και στην Επιτροπή Euromed και ετοιμάσαμε αυτό το σχέδιο κειμένου που το υποβάλαμε στην Ευρωμοσυγειακή Σύνοδο Κορυφής και βάλαμε και διάφορες παρατηρήσεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωμοσυγειακής. Δεν θέλω να κάνω εξαντλητική ανάλυση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελματικής στις ευρωμεσογειακές χώρες, διότι υπάρχουν άλλα κέντρα έρευνας. Το, το Ίδρυμα του Τωρίνου καταρχάς, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, όπου έχουν άλλες δυνατότητες λεπτομερούς ανάλυσης με επικαιροποιημένα στοιχεία. Εμείς ε, βρήκαμε κάποια προβλήματα κοινά, κάναμε προτάσεις παρέμβασης, ξεκινώντας πάνω απ' όλα από μια ανάγκη συντονισμού με τους άλλους ε, δωρητές στην περιοχή, διότι υπάρχουν και διεθνείς οργανώσεις, υπάρχουν και χώρες δωρητές που δραστηριοποιούνται με το στόχο να υπάρχουν προγράμματα στις διάφορες αυτές χώρες και όχι κατακαιρματισμένες και μη συντονισμένες παρεμβάσεις όπως σήμερα με μια διασπάθηση των πόρων. Θα μπορούσε να είναι συγκολητική ουσία των πρωτοβουλειών η Ευρώπη λοιπόν να παίξει το ρόλο το συντονιστικό η Ευρώπη και γεωπολιτικές προτεραιότητες σε αυτή την περιοχή, διότι η περιοχή αυτή έχει αυτή τη σημασία γεωπολιτική. Ε, σε τρει φάσει δημιουργήθηκε αυτή η έκθεση, σε τρία τμήματα μάλλον. Πρώτα απ' όλα ε, είδαμε τα προβλήματα που αφορούν τα βασικά συστήματα παιδεία, ανωτέρα παιδεία, μετά τα συστήματα επαγγελματική κατάρτιση τεχνικού περιεχομένου και τρίτον πώ να περάσουμε από την τεχνική κατάρτιση προ την πρακτική διάφορες ε, εκμάθησεις επιχειρήσεις και στις εταιρείες, εμπειρία μέσω δραστηριοτήτων επιτοπίων και σε, στις επιχειρήσεις. Το πρόβλημα που εντοπίσαμε, που είναι σαφές στη σπάση, είναι η οικονομική κρίση, η πολιτική αστάθεια και αυτά δεν επέτρεψαν να υπάρξει επενδυτική πολιτική μέσω μακροπρόθεσμη, αλλά ήταν επενδύσεις περιορισμένες χρονικά, Βρήκαμε προβλήματα στον με την πρόσβαση στην βασική παιδεία, κυρίως για τα κορίτσια, έλλειψη ανάληψης ευθυνών από τα κράτη να έχουν αποτελεσματικά και ποιοτικά συστήματα. Η επαγγελματική κατάρτιση παραμένει πολύ λίγο ελκυστική, διότι τα προγράμματα είναι πολύ απερχιωμένα, με σχολές που δεν είναι τόσο επαγγελματικές όσο θα έπρεπε και είχαμε κάποια θετική εμπειρία όσον αφορά την κατάρτιση και διάφορε δοκιμέ όσον αφορά την πρακτική κατάρτιση που εφαρμόζουν ευρωπαϊκέ εταιρείε, αλλά σίγουρα θα χρειαζόταν να δημιουργηθεί ένα σύστημα τουλάχιστον μαθητεία σε επίπεδο επιχείρηση με μαθήματα κατάρτιση σε υπερεθνικό επίπεδο που θα επιτρέπουν μια εργασιακή κινητικότητα, των εργαζομένων. Θα σταματήσω τώρα εδώ γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο. Σχεδόν. Το ξεπεράσετε. Περνάμε στη συζήτηση. Για ένα λεπτό το λόγο, κυρία Νταβουραουσκίν. Ευχαριστώ πολύ. Ούτε λεπτό δεν χρειάζομαι. Να συγχαρώ την εισηγήτρια. Πολύ πλούσια και χρήσιμη έκθεση για τους ανθρώπους της Μεσογείου να δουν ποια είναι η κατάσταση στι διάφορε μεσογειακές χώρες. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση. Όταν στιάζεται κανεί επί ενό προβλήματος, επί των προκλήσεων σε ένα τομέα και μπει σε βάθο, δεν έχουμε τα μέσα όπως το ETF αλλά το SEDEFOP, αλλά σε πολιτικό επίπεδο διαπιστώνουμε τα προβλήματα. Αυτοί οι φορεί που προανέφερα δεν πάνε πίσω στην κοινωνία των πολιτών, δεν, δεν εξετάζουν το θέμα τόσο πρακτικό, δεν μιλάνε με του νέου όπω κάναμε. Γιατί και εγώ προσεκλήθην σε μία από τι συναντήσει και είδα ότι έγινε αυτό. Είναι πολύ καλή η προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Και προτείνω και άλλε περιοχέ να ακολουθήσουν παρόμοια προσέγγιση, να εστιαστούν σε ένα θέμα και να το συζητούν ει βάθο το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η, κυρία Ντεφελή Πελετώνε. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Τελερίο, την εισηγήτριά μας, για το έργο της. Είχα τιμή να είμαι πρόεδρο τη ε, Επιτροπής Μελέτης και είχαμε και την ε, Ευρωμεσογειακή Σύνοδο στο Τωρίνο. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προσμίμηση για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και τη Μέση Ανατολή που μας έχουν ως παράδειγμα άσκηση πολιτικής για τα θέματα αυτά. Πραγματικά από τον Αύγουστο εργαστήκαμε πυρετοδός με την εισηγήτρια, αλλά νομίζω ε, το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την ε, Σύνθια για την αρτιότητα της γνωμοδότηση. και μόνο ο τρόπος ε, ε, εκπώνησης της γνωμοδότησης ε, και η διατύπωση ε, αναδείχθηκε στο Τωρίνο και έδειξε πόσο εύστοχη ήταν και πόσο απαραίτητη στην περιοχή και κυρίως στη νότια πλευρά της Μεσογείου που υπάρχει ψηλή ανεργία, κυρίως νέων στην, για την Αίγυπτο ακούσαμε ότι περίπου ένα εκατομμύριο νέοι κάθε χρόνο βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, δεν μπορούν να βρουν θέσεις απασχόλησης ε, νέα άτομα με πολύ ψηλή δίκευση. Ενώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση τεχνικών δεξιοτήτων. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν καλά εκπαιδευτικά συστήματα και επαγγελματικής κατάρτισης ε, με πρόσβαση σε όλους φυσικά. Δυστυχώς τα συστήματα στις χώρες αυτές δεν είναι τόσο καλά ανεπτυγμένα όπως αναφέρεται και στη γνωμοδότηση. Είναι παλιωμοδίτικα αυτά τα συστήματα, παροχημένα. Εν πάση περιπτώσει, είμαι υπέρ της γνωμοδότησης και σας συστήνω να την υπερψηφίσετε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γέλιτς, τελευταία μιλήτρια για ένα λεπτό επίσης. Ευχαριστώ. Πολύ λακωνικά. Εγώ δεν είμαι μέλος του τμήματος απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, αλλά ένιωσα την ανάγκη να λάβω το λόγο και να εκφράσω το θαυμασμό μου για την έκθεση αυτή. Θα πρέπει να βαθύνουμε περισσότερο σε αυτά τα θέματα. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι η παρουσίαση τέτοιων επαγγελμάτων ώστε να γίνουν ελκυστικά κυρίως τους νέους. Θα πρέπει να προσελκύσουμε τους νέους ε, σε τέτοια επαγγέλματα, αλλά να πείσουμε και τους γονείς ότι θα πρέπει να οθούν τα παιδιά τους σε επαγγελματικά αλήκεια και επαγγελματικές σχολές, γιατί αυτές θα τους εξασφαλίσουν σίγουρη επαγγελματική διέξοδο. Ε, θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση των προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και των επιχειρήσεων. Επίσης, θα πρέπει να ανασχεδιάσουμε το πρόγραμμα σπουδών ώστε να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Γιατί αν δεν συνδέσουμε την παιδεία με τις ανάγκες αγοράς εργασίας δεν πρόκειται να έχουμε ποιοτικό εργατικό δυναμικό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Για όλα αυτά θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και να εκφράσω την υποστήριξή μου για την γνωμοδότηση. Η κυρία Ντελερίο για δύο λεπτά για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ξεκινώντας από τη συνάδελφο Ντεφελίπε διότι μου έδωσε μεγάλη βοήθεια, διότι ακολουθήσαμε διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις άλλες ευρωμοσαγικές συνόδους κορυφής. Εντοπίσαμε ένα θέμα, όπως είπε και η Τατιάνα, και μετά το θέσαμε στην προσοχή και των συναδέλφων των επιτροπών της, ε, των νοτίων ακτών της Μεσογείου. Είχαμε ε, ένα κοινό έγγραφο για συζήτηση το υποστήριξαν όλοι. Να υπογραμμίσω αυτή την πτυχή που είναι σημαντική. Θα είναι ένα έγγραφο αυτό, το οποίο θα είναι ένα εργοτάξιο, work in progress, και στην επόμενη σύνοδο θα είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα συζητηθεί για να κατανοήσουμε ποια βήματα προόδου έχουν επιτευχθεί. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να δουν τις προτάσεις που κάνουμε προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προς τις κυβερνήσεις και προς τις διεθνείς ε, οργανώσεις, την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και να υπάρχει μεγάλο συντονισμός για να αποφύγουμε ε, μια διασπάθηση των πόρων. Τελευταίο σημείο, οι νέοι σίγουρα έχουμε εκθετική αύξηση των νέων που αντιμετωπίζουν την κατάρτιση και την παιδεία το θέμα των κοριτσιών στο σχολείο είναι ένα πρόβλημα ακόμα πιο διαχυτό σε κάποιες από αυτές τις χώρες και ίσως υποχρέωση ε, για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο που δεν υπάρχει ίσως να είναι μια λύση. Αλλά θα ήθελα να παρέμβουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Ευχαριστώ όλους για μια ακόμη φορά και την εμπειρογνώμονά μου που συνεργάστηκε μαζί μου ακόμα και το καλοκαίρι. Pues muchas gracias. Σας ευχαριστώ, Σύνθια. Θα ψηφίσουμε τώρα. Και θα διαβιβάσουμε αυτήν την ενημερωτική έκθεση στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Άρχεται η ψηφοφορία. se ha ido. Tampoco se pasa nada por 10 segundos y luego hay dos, tres. Muy bien, cerramos. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται παμψηφή η γνωμοδότηση της κυρίας Δελρίο. Συγχαρητήρια. και για τους γενναίους συναδέλφους που παρέμειναν μέχρι το τέλος συνεδρίασης. Περάμε στη τελευταία γνωμοδότηση, την υπαριθμό 484 του τμήματος ΕΚΟ, ΟΝΕ και Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής, με θέμα το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή. Πρόκειται για διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν ετήματος της Ρουμανικής Προεδρίας. Η είναι ο κύριος Στέφανο Μάλια και συνεισηγητής ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Περνάμε στη συζήτηση της έκθεσης αυτής μετά την παρουσίαση. Δύο λεπτά για τον εισηγητή και δύο λεπτά για τον συνεισηγητή. Θα ξεκινήσει ο κύριος Μάλια με την παρουσίαση της νομοδότησης. θα μιλήσω στα Μαλτέζικα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ και που βρίσκεστε εδώ, που είναι αργά τώρα. Εκτιμώ την εδώ παρουσία σας τέτοιες ώρες. Αυτή η έκθεση, όπως εξηγήθηκε άριστα από την Πρόεδρο, ζητήθηκε από τη Ρουμανική Προεδρία. Όταν ξεκινήσαμε την σύνταξη της γνωμοδοτήσεως, είχαμε παρουσιάσει διάφορες γνωμοδοτήσεις περί πολιτικής συνοχής. Ήταν τμήμα Ήμασταν ο πρώτος φορέας τη Ευρωπαϊκής Ενώσεω που γνωμοδότησε πάνω στην πολιτική συνοχής. Αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί με τον συνάδελφό μου ήταν λοιπόν να βασιστούμε σε αυτά που ήδη είχαν γραφτεί, στα κείμενα που υπήρχαν, αλλά να δίνουμε νέα μηνύματα και για το μέλλον. Νέα μηνύματα για το μέλλον μετά το 2020. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Είχαμε αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες στην Οι ελληνικές αρχές μας είχαν προσκαλέσει να πάμε να δούμε διάφορα έργα, διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής και να συζητήσουμε δημόσια με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και εμπλεκόμενους φορείς που μας βοήθησαν να διαμορφώσουμε αυτή τη γνωμοδότηση που έχετε μπροστά σας. Δεν θα επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, όμως θα ήθελα να στείλω κάποια μηνύματα. Είναι απαράδεκτο να μειώνεται ο προϋπολογισμός κατά 10%, κάτι που προτάθηκε. Αυτό που λέμε είναι ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Θα πρέπει να ανασχεδιαστεί, ούτω ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στο μέλλον. Και να ανταποκρίνεται στα προβλήματα όπως η αλλαγή του κλίματος, και η βιώσιμη μετάβαση προς νέες τεχνολογίες. Κλείνω λέγοντας ότι δεν μπορούμε να λησμονήσουμε τις παραδοσιακές προκλήσεις, τα προβλήματα, τα παραδοσιακά, όπως είναι η φτώχεια, όπως είναι η ανάγκη για την κατάρτιση ε, για τους εργαζομένους. Και τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Γιάννη. Ευχαριστώ. Θα ακολουθήσω το παράδειγμα του Στέφανο και θα μιλήσω ελληνικά. Πριν ε, μιλήσω για αυτήν την επιτροπή θέλω 20 δευτερόλεπτα να χρησιμοποιήσω γιατί για ένα άλλο θέμα δεν ήμουν εδώ όταν συζητήθηκε του Κρίστοφ Πάτερ το report για το δικαίωμα στο ψήφο των ε, Ευρωπαίων πολιτών με αναπηρία ε, όμως ε, την ώρα που ο κύριος Πάτερ μίλαγε εδώ και συζητούσατε και το υποδεχτήκατε πολύ θερμά, εγώ παρέδιδα το report στον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τίμερμαντς. Συνεπώς ήδη έφτασε σε σπουδαία χέρια. Όπως ο Στέφανο ανάφερε, αυτή η γνωμοδότηση έρχεται να κεφαλαιοποιήσει όλη τη δουλειά που κάναμε και που στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου εγκρίθηκε για το πακέτο της πολιτικής συνοχής 21-27. Συμφωνώ απολύτως με ό,τι ανάφερε. Εγώ θέλω επίσης τρία μηνύματα να αναφέρω. Το πρώτο είναι ότι τα δικαιώματα είναι αφηρημένες κατασκευές εάν οι πολίτες δεν μπορούν να τα ισχύσουν και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Και η πολιτική συνοχής είναι το εργαλείο που από τη μια μεριά αντιμετωπίζει τις ανισότητες ανάμεσα στις περιφέρειες της Ευρώπης και από την άλλη μεριά τις ανισότητες ανάμεσα στους πολίτες. Συνεπώς κάνει τα δικαιώματα χειροπιαστή πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι ότι η πολιτική συνοχή πρέπει να συνδεθεί με την Ατζέντα 2030 και τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ. Έχει υποχρέωση την επόμενη δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει την ατζέντα και η πολιτική συνοχής είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο να το κάνει αυτό. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί η εταιρική σχέση και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όχι μόνο στο σχεδιασμό, αλλά και στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση της πολιτικής συνοχής και στο επίπεδο των κρατών μελών, αλλά και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ευχαριστήσω και εγώ τους συμπατριώτες μου στην Ελλάδα για τη φιλοξενία τον εισηγητή και την γραμματεία, τον Γκίλμπερ, τον Στέφανο και την Ραφαέλα και όλα τα μέλη της Επιτροπής, την Έστερ, την πρόεδρο ε, της ομάδας μελέτης για την εξαιρετική συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στη συζήτηση. Η κυρία Βιτάλ έχει το λόγο. Για ένα λεπτό όμως, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχα την τιμή να προεδρεύσω αυτής της ομάδας μελέτης και μπορώ να πράγματι να πω ότι είμαι μάρτυρας πόσο ο εισηγητής και ο συνεισηγητής κατέβαλαν άοκνες προσπάθειες για να ετοιμάσουν αυτή τη γνωμοδότηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής που πώς να το πω που πρέπει να, ε, να βρούμε μέτρα που να αντέξουν στο μέλλον να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη σχέση με τις τοπικές αρχές, με την περιφέρεια, ε, να βελτιώσουμε την επικοινωνία, πρέπει να ευνοήσουμε τη συμμετοχή ε, των διαφόρων φορέων και τη συνεργασία. Αυτό προϋποθέτει μια αύξηση των ιδίων πόρων της Ένωσης. Είναι απόλυτα αναγκαίο αυτό, αν θέλουμε να δώσουμε ζωή, καλύτερη ζωή, μέσω της πολιτικής συνοχής. Αυτό σωστά αναφέρεται στη γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι είναι μια γνωμοδότηση αρκετά εξαντλητική παρά το γεγονός ε, ότι το θέμα ήταν τεράστιο έπρεπε να εξεταστεί, αλλά οι δύο εισηγητέ έκαναν εξαιρετική δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Καλό όλους να υπερψηφίσουν τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ τον Στέφανο και τον Γιάννη για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ καλή γνωμοδότηση. Κρίμα που τη συζητούμε προς το τέλος συνεδρίασης αργά. Συμβαίνουν όμως αυτά, αραιά και πού. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές, ευχαριστώ και την ομάδα μελέτης. Υπέροχη δουλειά που έκαναν. Συνήθως δεν παίρνω το λόγο στην Ολομέλεια, αλλά πρέπει να πω ευχαριστώ πολύ για μια καλή γνωμοδότηση. Προσωπικά πιστεύω ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάμβανε τουλάχιστον, ελάμβανε υπόψη μάλλον κάποιε συμβουλές αυτές για τη συνεργασία και την πολιτική συνοχής, θα βοηθούσε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό και θα μπορούσε να καλύψει το κενό που υπάρχει μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Μιλάμε για συμπράξη, συνεργασία, μιλάμε για συμμετοχή και να στηρίξει το κοινό την πολιτική και νομίζω ότι αυτά είναι τα διάφορα ελλείμματα που έχουμε και γι' αυτό οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις ισχυροποιούνται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια υπέροχη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι μια έξοχη αυτή η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές. Δύο πράγματα θα ήθελα να τονίσω. Το ένα είναι ότι θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι γίνεται μνήα της επικοινωνίας. Επικοινωνία όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει καλή ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Μπορούμε όλοι να μάθουμε ημένα από τους δε. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η πρόσβαση των μικρών και πολύ μικρών εταιριών και των μεσαίων επιχειρήσεων και είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών, διότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν αυτή τη συνεισφορά. Ένα λεπτό, έχουμε τώρα για τον εισηγητή και τον συνεισηγητή μας για να απαντήσουν ε, στους συναδέλφους. Ευχαριστώ εκ νέου, ευχαριστώ πολύ για τα διάφορα υποστηρικτικά σχόλια που τα εκτιμώ όλους ιδιαίτερος και κάποια σημεία που ήθελα να αναφέρω για την επικοινωνία, για την ε, πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο σύστημα. Όλα αυτά είναι στα συμπεράσματα και ήλπιζα ότι ακόμα και σαν Επιτροπή μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε συνέχεια με περαιτέρω συστάσεις και άλλη δουλειά στον τομέα αυτό, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι συμβάλλουμε σε μια ισχυρή πολιτική συνοχή για το μέλλον. Ευχαριστώ τον συνσηγητή και συνάδελφο τον Γιάννη, συνεργάστηκα άριστα μαζί του και την κυρία Βιτάλια για την υποστήριξή της και τους, τα διάφορα μέλη της ομάδας μελέτης που είναι εδώ σήμερα. Νομίζω ότι πέρα από καλή δουλειά απολαύσαμε αυτή τη συνεργασία και ευχαριστώ και τον πρόεδρο του τμήματο ΕΚΟ. Ευχαριστώ για τη συνεχή υποστήριξή σα. Ευχαριστώ. Um, Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον πρόεδρο της ομάδας μελέτης και να σας υπενθυμίσω ότι η γνωμοδότηση αυτή έγινε από τρεις νησιώτες, τον Στέφανο από τη Μάλτα, ε, την έστερα τη Σικυλή και το υποφαινομένο που είναι από τη Ζάκυνθο. Νομίζω ότι φερθήκαμε καλά. Θα σας πω το εξής. Είπα στο Φρανς Τίμερμανς πριν από λίγο όταν του έδωσα την έκθεση ότι μια ισχυρή πολιτική συνοχής με ουσιαστική ανάμειξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούσε να είναι πραγματικά ε, η τροχοπέδη στον νευροσκεπτικισμό και τον εξτρεμ, εξτρεμισμό στους, τον καιρό, καιρούς μας. Ωραία, περνάμε στην ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Cerramos Τέλος ψηφοφορίας. 71 ψήφι υπέρ και μία αποχή. Ή μάλλον 72, γιατί φυσικά και ο κύριος Βαρδακαστάνης ψηφίζει. 72 ψήφι υπέρ λοιπόν και μία αποχή. Μπράβο σας και στους δύο. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που παρέμεινα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, κύριε Πρόεδρος. Και Αύριο θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση από τις 9 το πρωί. Καλό σας βράδυ.